Ja, liebe Kolleginnen und Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα παρακαλώ να ξεκινήσουμε την απογευματινή συνεδρίαση της Επιτροπής Άγκρη με το σημείο 10 που προβλέπει παρουσίαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη Γενική Διεύθυνση Υγείας, των κατεξιοδότηση πράξεων που συμπληρώνουν τον κανονισμό του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την υγεία των ζώων. Υπάρχει εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην αίθουσα. Ο κύριος Φαγκούτεν, κανονικά. Okay, so I give immediately... Θα δώσω αμέσως λοιπόν το λόγο σε εσάς κύριε Φανγκούτεν, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας εξηγήσω τι γίνεται με αυτό το πακέτο των τεσσάρων κατεξοδότηση πράξεων που ε, είναι προσυζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Θα ήθελα καταρχήν να σας κάνω μια εισαγωγή στη διαδικασία, γιατί πρόκειται για μια διαδικασία που ξεκίνησε εδώ και πολύ καιρό και διαπιστώνουμε ότι η αξιολόγηση του συνολικού ευρωπαϊκού συστήματος για την υγεία των ζώων ολοκληρώθηκε το 2006. Και το σλόγγαν της στρατηγικής ήταν «Καλύτερα πρόληψη παρά θεραπεία» και είχαμε διάφορες αξιολογήσεις και διαβουλεύσεις. Η νέα νομοθεσία για την υγεία των ζώων απορρέει από μια σειρά κανονισμών και οδηγιών που υιοθετήθηκαν από τις αρχές της δεκαετίας του 60 όταν δημιουργήθηκε η ΚΑΠ ε, για ε, Ζώο, όπως ε, ζωικής προέλευσης, ε, για την εξάλληψη νόσων όπως αυθόδη πυρετό, αφρικανική παρνόλη χείρων, για την εισαγωγή κρέατος και ζών των ζώων, για τη σπογκώδη κεφαλοπάθεια. Είχαμε πολλές οδηγίες, ήταν 60 τότε οι βασικές νομοθετικές πράξεις του Συμβούλιο και ε, περίπου χίλιε λίγο λιγότερες από χίλιε ε, εκτελεστικές πράξεις, αυτό που σήμερα αποκαλούμε εκτελεστικές πράξεις. Και αυτό ήταν το πλαίσιο τότε της ε, Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για την υγεία των ζώων. Υπήρξε ανάγκη λοιπόν αξιολόγηση και εξορθολογισμού αυτών των νομοθετικών πράξεων που μέχρι το 1992 ε, ολοκληρώθηκαν με την εσωτερική αγορά. Χρειάστηκε όμως μία αναδιατύπωσή τους και μία ομαδοποίησή τους σε μία ενιαία πράξη, νομοθετική πράξη που τώρα αποκαλούμε το Ευρωπαϊκό Νόμο, την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για την Υγεία των Ζώων. Περί τίνος πρόκειται λοιπόν. Πρόκειται για μεταδοτικές ζωονόσους που έχουν αντίκτυπο στο εμπόριο και στους κτηνοτρόφους και καλύπτει και ε, προϊόντα ζωικής προέλευσης, ε, βόλιο κρέας, χείριο κρέας, γάλα, οτιδήποτε προϊόν δηλαδή προέρχεται από ένα ζώο και που είναι πιθανό να μεταδώσει τις, την ασθένεια περιλαμβάνεται. Καλύπτουμε και υδρόβια ζώα, ψάρια και ερπετά. Και όπως βλέπετε στο κατάλογο έχουμε διάφορα κεφάλαια στην νομοθεσία, ε, πρόληψη, επιτήρηση, έλεγχο και εξάλληψη, κανόνες που ισχύουν για τις ενδοκοινοτικές μετακινήσεις, όταν μεταφέρονται ζώα από τη μία την άλλη, προς την άλλη περιοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, κανόνες που ισχύουν για την είσοδο ε, από στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τι ισχύει για το προϊόντα βοήου κρέατος που εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επίσης υπάρχουν και κάποια μέτρα εκτάκτου ανάγκης που ενεργοποιούνται όταν εσκύπτει μια κρίση. Πάντως, η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για την ε, ε, υγεία των ζώων δεν αφορά την ευζοία, την καλή μεταχείριση των ζώων, δεν αφορά χρηματοδότηση της εξάλληψης των ζωνώσεων, δεν αφορά τις ζωτροφές και τις φαρμακοχές ζωοτροφές, δεν αφορά τα κτηνιατρικά φάρμακα, ούτε τους επίσημους ελέγχους. Όλα αυτά δεν είναι λοιπόν η νομοθεσία για την υγεία των ζώων. Αυτές, αυτοί οι τομείς εμπίπτουν σε άλλες νομοθετικές πράξεις, όχι στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για την υγεία των ζώων. Επίσης, ε, έχουμε άλλες νομοθετικές πράξεις που έχουν ε, ή αντίκτυπο στην υγεία των ζώων ή στη δημόσια υγεία, όπως, ε, είναι τα υποπροϊόντα τα ζωικά. Ε, στα σφαγεία, για παράδειγμα, ζωικά υποπροϊόντα μπορεί να χρησιμοποιηθούν για ζωτροφές. Έχουμε τους κανόνες ε, για την βόδια εγκεφαλοπάθεια ή τη μεταδοτική σπογγόδια εγκεφαλοπάθεια και κάποιες ζωονόσους. Αυτά που είναι σε κόκκινο στις δεν καλύπτονται από την νομοθεσία για την υγεία των ζώων. Όπως σας είπα, είχαμε πολλές οδηγίες και κανονισμούς, κυρίως του Συμβουλίου, και είχαμε περίπου 50-60 βασικούς κανονισμούς που αν τους ε, συνδυάσουμε καταλήγουμε σε μια νέα νομοθετική πράξη του 1996 που ε, χωρίστηκε σε 8 διαφορετικά κεφάλαια. Γενικοί κανόνες, προειδοποίηση, ενημέρωση, επιτήρηση, προγράμματα εξάλληψης, τρίτο κεφάλαιο επαγρύπνηση, ετοιμότητα και έλεγχος των νόσων. Το τέταρτο κεφάλαιο αφορούσε την καταγραφή, έγκριση και ηχνηλασιμότητα των κινήσεων, καταγραφή των εκμεταλλεύσεων, των αγορών από τις οποίες πέρασαν τα ζώα. Κεφάλαιο 5. Είσοδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τι κανόνες ισχύουν δηλαδή για την είσοδο ζών των ζώων ή προϊόντων ζωικής προέλευσης που εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το έκτο κεφάλαιο αφορούσε τα ζώα συντροφιάς ε, μη εμπορικού χαρακτήρα. Το κεφάλαιο 7 αφορά μέτρα εκτάκτου ανάγκης που πολύ συχνά θα χρησιμοποιούνται σε εξαιρετικέ επίγουσε καταστάσει, όπω είχαμε την Αφρικανική Πανόλη των Χείρων ή την ε, γρήπη των πουλερικών. Και το τελευταίο κεφάλαιο είναι κοινέ και μεταβατικέ διατάξει. Τώρα να σας εξηγήσω τη διαδικασία. Όπως σας είπα, η έγκριση της σχετικής νομοθεσίας έγινε το 2016 και οι ομάδε εμπειρογνωμόνων 2017 ε, με 2019 ανέπτυξαν τις διάφορες ε, ε, νομοθετικές πράξεις. Το ίδιο ισχύει και για την καταχώρηση σε καταλόγους των ζώων με εφαρμοστικέ εκτελεστικέ εκατεξοδότηση εκτελεστικές πράξεις και οι περισσότερες νομοθετικές πράξεις τώρα δρομολογούνται, είναι σε φάση υιοθέτηση ώστε στι 21 Απριλίου του 2021 που θα τεθούν σε ισχύ να έχουν προετοιμαστεί όλα τα κράτη-μέλη για την άμεση εφαρμογή τους. Επίσης βλέπετε στην οθόνη πόσες ομάδες εργασίας και πόσες ομάδες εμπειρογνωμόνων ασχολήθηκαν με το θέμα αυτό στα κράτη-μέλη, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Χρειάστηκαν όλες αυτές οι συνεδριάσεις των εμπειρογνωμόνων για να αναπτύξουμε τα διάφορα τμήματα αυτής της νομοθεσίας για την υγεία των ζώων είναι ένας τρόπος λισαβονοποίησης τρόπον τεινά όλων αυτών των νομοθετικών πράξεων που ίσχυαν στο παρελθόν. Δεν κάνουμε κάτι ρηξικέλευτο, δεν αλλάζουμε τον κόσμο. Έχουμε τη νομική υποχρέωση να προσαρμόσουμε αυτό το πολυσύνθετο νομικό πλαίσιο του παρελθόντος στο νέο νομικό πλαίσιο που διαμορφώθηκε μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας. Και γι' αυτό σκεφτήκαμε ότι καλό θα ήταν να καταργηθούν οι 60 βασικές πράξεις και οι 900 περίπου εκτελεστικές πράξεις και να τα ομοδοποιήσουμε όλα σε ένα νομοθέτημα συνεκτικό και συμπαγές που θα πρέπει να εφαρμοστεί τώρα εξού και η κατεξοδότηση και εκτελεστικές πράξεις που εξετάζεται και που ουσιαστικά πραγματοποιούν έναν εξορθολογισμό, μια πλούστευση και μια διατύπωση βάση κινδύνου των προηγούμενων νομοθετημάτων. Είδαμε τη διαδικασία, έχει εγκριθεί η σχετική νομοθεσία και τώρα με το πακέτο των τεσσάρων πράξεων που θα εξετάσετε. όσες εγκρίθηκαν και δημοσιεύθηκαν πράξεις αφορούσαν το κατάλογο των ζωονόσων, την κατηγοριοποίηση των ζωονόσων και τον κατάλογο των ζωικών ειδών που συμπληρώνουν το πρώτο τμήμα των κατεξοδότηση πράξεων της νομοθεσίας για την υγεία των ζώων. Και έχουμε και δύο διαφορετικούς κανονισμούς. Ο πρώτος ε, αφορούσε τις κατεξοδότηση πράξης και υιοθετήθηκε το 2018 και κάτω δεξιά έχουμε σε κάθε, σε κάθε καταχωρημένη νόσο ε, προσαρτούμε μια... ή συνδέουμε μια κατηγορία και ένα συναφές ζωικό είδος. Κάτι άλλο που έχει διεγκριθεί και δημοσιευθεί είναι μια κατεξοδότηση πράξη για την ταυτοποίηση των ζώων και την ειχνηλασιμότητα. Και στο συγκεκριμένο πλαίσιο είχαμε συνομιλήσει και κάποιους ε, ευρωβουλευτές για να προβλέψουμε απόκληση για τα νεαρά πρόβατα και ε, κατσίκες και η σχετική τροπολογία εξετάζεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχετε ενώπιό σας λοιπόν ένα πακέτο τεσσάρων πράξεων που καλείστε να ελέγξετε. Η πρώτη φορά την επιτήρηση, εξάλληψη και εξαφάνιση της νόσου Ε, θα πρέπει να δούμε πότε μια φάρμα ή μια περιοχή είναι απαλλαγμένη από την νόσο, χωρίς νόσο. Δεύτερη κατεξοδότηση πράξη αφορά τα μέτρα ελέγχου των νόσων και σχετίζονται με το τρίτο τμήμα της σχετικής νομοθεσία. Σας έδειξα προηγουμένως τις διαφάνειες τα οχτώ διαφορετικά κεφάλαια. Η δεύτερη κατεξοδότηση πράξη αφορά το δεύτερο κεφάλαιο, ε, το τρίτο συγγνώμη κεφάλαιο, τα μέτρα ελέγχου και τα δύο τελευταία, οι δύο τελευταίες εκτελεστικές πράξεις κατεξοδότηση πράξη αφορούν τις κινήσεις των χερσαίων ζώων και την χρησιμότητα και, και τις κινήσεις των αναπαραγωγικών προϊόντων. Αυτές οι τέσσερις κατεξοδότηση πράξεις είναι αλληλένδετες. Και υπάρχουν και πολλές παραπομπές από τη μια στην άλλη. Το πακέτο αυτών των τεσσάρων κατεξοδότηση πράξεων θεωρείται και από εμά και από τα κράτη-μέλη ως ενιαίο πακέτο που καλύπτει τα πάντα. Και είναι και ογκώδες, 500 περίπου σελίδες αυτό το πακέτο των κατεξοδότηση πράξεων. Περνάμε τώρα στην πρώτη πράξη που αφορά την επιτήρηση των νόσων, τα προγράμματα εξάλληψης και το καθεστώς χωρίς νόσο. Όπως είπα προηγουμένως, έχουμε τους ε, υφιστάμενους κανόνες που αναφέρονται εδώ. Είχαμε κανόνες δηλαδή από την Οδηγία 64-432 που έχει επανειλημμένως τροποποιηθεί μέχρι πρόσφατα. Υπήρχαν στην οδηγία τότε οι υπάρχοντες κανόνες. Υπήρχαμε την, είχαμε την οδηγία για τα μικρά μυρικαστικά, την οδηγία για μια αρρώστια των Blue Tank, την τρομόδη νόσο των προβάτων. Επίσης, είχαμε διάφορες νομοθετικές πράξεις και στα παραρτήματά τους που κατέληξαν στη νέα κατεξοδότηση πράξη που έχετε ενώπιόν σας και που αποτελούν την νέα νομοθετική πράξη. Έχουμε αποκτήσει μεγάλη πείρα σε όλα αυτά τα χρόνια που ασχοληθήκαμε με την υγεία των ζώων και γι' αυτό θέλουμε να τροποποιήσουμε τους κανόνες και γι' αυτό ζητήσαμε και τη γνώμη το, του Οργανισμού Ασφάλειας Τροφίμων, εμπειρογνώμονες και φυσικά τα πρότυπα του Διεθνούς Γραφείου Επιζωτιών, του OIE, που είναι η παγκόσμια οργάνωση που θεσπίζει τις κατευθυντήριες γραμμές που ισχύουν για το εμπόριο σε παγκόσμιο επίπεδο. Όλα αυτά αποτέλεσαν τη βάση για μας για να εκπονήσουμε αυτές τις καταξιοδότησες πράξεις και στόχος είναι να υπάρχει μια σαφήνεια για τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς, ε, μεγαλύτερη ευελιξία για τις αρμόδιες αρχές και να έχουμε μια προσέγγιση που θα στηρίζεται στον κίνδυνο προσέγγιση βάση κινδύνου, ώστε οι πόροι που αφιερώνονται για τη χρήση ε, για τη διατήρηση αυτού του καθεστώτος χωρίς νόσο να χρησιμοποιούνται από τα κράτη-μέλη. Όπως είπα και προηγουμένως, το περιεχόμενο αυτής της ε, κατεξιδότηση πράξης ε, είναι συμπληρωματικό του τμήματος 2 ε, που αφορά του, σχετικού νόμου που αφορά την επιτήρηση, την εξάλληψη των προγραμμάτων και το καθεστώς χωρίς νόσο, απαλλαγμένο από την νόσο. Οπότε έχουμε το κατάλογο των ε, νόσων και κριτήρια για τα προγράμματα επιτήρησης. Έχουμε ζώνες ή χώρες που έχουν αναγνωριστεί ως ε, ελεύθερες από την νόσο, χωρίς νόσο. Βρίσκουν και τα κριτήρια για να διατηρήσουν αυτό το καθεστώς. Επίσης, έχουμε και τα προγράμματα εξάλληψης. Για κάποιες ζωνώσεις θα πρέπει να υποβάλλονται από τα κράτη-μέλη, βρουκέλωση, λύσα, MTBC, είναι οι πιο συνηθισμένες κατηγορίες Β. Και έχουμε και άλλες νόσους, για τις οποίες τα κράτη-μέλη δίνανται, προαιρετικά δηλαδή, εθελοντικά να προβούν σε εξάλληψη, από τη στιγμή που φτάσει η ζωνόσος σε κάποιο επίπεδο οι εμπορικέ ευκαιρίε είναι μεγαλύτερε και οι περιορισμοί στο εμπόριο πολύ μικρότεροι. Οπότε έχουμε και τους κανόνες για το πώς θα χορηγηθεί το καθεστώς ε, χωρίς νόσο για χώρες, ζώνες ή περιοχές και επίσης, επίσης λέμε πώς θα διατηρηθεί αυτό το καθεστώς ε, χωρίς νόσο σε όλε τι ζωνώσεις. Δεν περιορίζεται δηλαδή στι ζωνώσεις που ανέφερα, αλλά μπορεί να, ισχύσει, να ισχύσουν οι κανόνε αυτοί και για μία σειρά άλλων νόσων. Η δεύτερη κατεξοδότηση πράξη αφορά την πρόληψη και τον έλεγχο των καταχωρημένων ζωνώσεων. Έχουμε εδώ την Αφρικανική Πανόλη των Χείρων ή τον ε, αυτόδη Πυρετό Επίσης, πήραμε κάποιους κανόνες από τις ε, υφιστάμενες οδηγίες. Λάβαμε υπόψη την εμπειρία που συγκεντρώσαμε όλα αυτά τα χρόνια και δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε και πολύ κακή πείρα με πολλές ζωονόσους όλα αυτά τα χρόνια. Mm-hmm. Όλα αυτά τροφοδότησαν το νέο νομικό πλαίσιο και φυσικά και τα πρότυπα του Διεθνούς Γραφείου Επιζωτιών ελήφθησαν υπόψη. για τις ε, κατηγορίες ε, της ε, πρώτης για τις ανανώσεις πρώτης κατηγορίας Αφρικανική Επανόλη των Χείρων γρήπη πουλερικών έχουμε άμεση επέμβαση από τις αρμόδιες αρχές και θανάτωση των ζώων για τις ζωνώσεις κατηγορίας Α. Πάντως, αντί να έχουμε ένα κατακαιρματισμένο νομοθετικό τοπίο, τα έχουμε συγκεντρώσει όλα σε μία εξοδότηση πράξη. Και βλέπετε στα δεξιά τις ε, σαφέστατες υποχρεώσεις των παρόχων και την ε, δέουσα ευελιξία για τις αρμόδιες αρχές. Επίσης έχουμε κάποιους ε, κανόνες για την επαγρύπνηση, την ετοιμότητα και τον έλεγχο των νόσων. συμπληρώνει το τμήμα 3 της νομοθεσίας για, τις, για την υγεία των ζώων. Έχουμε νέες διατάξεις για την δειγματοληψία και κάποια μέτρα που λαμβάνονται σε περίπτωση που υπάρχει υπόνοια νόσου. Προβλέπονται υποχρεώσεις του παρόχου, του επιχειρηματία, ή υποχρεώσεις για τις αρμόδιες αρχές, το εύρος της ζώνης, πώς θα εκενωθεί η εγκατάσταση, πώς θα επανέλθουν τα ζώα στην, στην εγκατάσταση και τι μέτρα θα ληφθούν σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί ε, η νόσος αυτή και σε άγρια ζώα. Για να, για να σας φέρω ένα παράδειγμα, η παθογονική, η υψηλής παθογένειας μάλλον ε, γρήπη των πουλερικών όταν εμφανίζεται σε μία φάρμα τότε ισχύουν άλλοι κανόνες που προβλέπονται και καταγράφονται σε αυτή την κατεξοδότηση πράξη. Περνάμε τώρα στην τρίτη κατεξοδότηση πράξη που αφορά τις μετακινήσεις και τις απαιτήσεις υγείας των ζώων για τις μετακινήσεις ε, χερσαίων ζώων και αυγών επόασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. ίσχυε από το 1964 μέχρι την ε, ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς η σχετική οδηγία και προβλέπουμε τις μετακινήσεις βοηδών, χείρων, ε, εγωπροβάτων και ύπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα όλες αυτές τις διατάξεις που είχαμε στο παρελθόν τις έχουμε συμπεριλάβει στην νομοθεσία για την υγεία των ζώων και η συγκεκριμένη κατεξουδότηση πράξη συμπληρώνει αυτό που υπάρχει ήδη στην νομοθεσία για την υγεία των ζώων. Σας είπα ποιοι κανόνες θα πρέπει να ισχύουν σε περίπτωση που, μετα που μετακινούνται πρόβατα από την Ιρλανδία στην Ελλάδα, τι κανόνες θα πρέπει να ισχύουν όταν μετακινούνται βοηδοί από τη Βόρεια Γαλλία στο Λουξεμβούργο, ποιοι κανόνες θα πρέπει να ισχύουν όταν, μετα, όταν μεταφέρεται γάλα, γιαούρτι, τυρί, όλοι οι κανόνες καλύπτονται από τη συγκεκριμένη κατεξοδότηση πράξη που αφορά τις μετακινήσεις, μετατοπής. Επίσης, συμπεριλαμβάνουμε και τα πρότυπα του Διεθνούς Γραφείου Επιζωτιών με σαφείς υποχρεώσεις για τους ε, επιχειρηματίες και περισσότερη ελαστικότητα για τις αρμόδιες αρχές. Επίσης, η σχετική πράξη καλύπτει και τα αυγά επόασης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι παγκόσμια ολική παραγωγός αυγών προς επόαση. Επίσης, ε, προβλέπει τα κριτήρια για τα μέσα μεταφοράς, που είναι σημαντικό στοιχείο της ασφάλειας, και προβλέπει και κάποιες απαιτήσει υγείας για τις ε, μετακινήσεις σε περίπτωση που μετακινούνται ζώα από τη μία πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε άλλη, περνούν από κάποια κέντρα στα οποία χρειάζονται κάποιοι κανόνες βιοασφάλειας που θα εφαρμόζονται για να αποφευθεί πρόβλημα. Για παράδειγμα, να μην εξαπλωθεί η λίμωξη σε περίπτωση που κάποιο ζώο είναι φορέας. Επίσης, προβλέπονται ειδικοί κανόνες για περιορισμένες, για περιορισμένες εγκαταστάσεις, για εγκαταστάσεις δηλαδή που αφορούν ειδικά ζώα, που επίπτωση ειδικό καθεστώς, προβλέπονται ειδικοί κανόνες και εξαιρέσεις για τις μετακινήσεις ζώων που δεν είναι τόσο γνωστά όσο είναι η χείρη και τα βοηδή. Και επίσης προβλέπονται πιστοποιητικά υγείας για ύπους ε, που συμμετέχουν σε αθλητικές οργανώσεις, υποδρομίες κτλ. Και η τελευταία κατεξοδότηση πράξη αφορά τις απαιτήσει υγείας για αναπαραγωγικά προϊόντα. Ε, υπάρχουν πολλά προϊόντα ε, σπέρματος βοηδών και εμβρίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν τέσσερις ε, σχετικές νομοθεσίες Βέβαια είχαμε και την αγνομοδότηση του ΕΦΣΑ και τις επιστημονικές ε, εξέλιξεις και τα πορίσματα, γιατί μπορούν ε, κάποιες ε, νόσεις, ζωνώσεις, να μεταδοθούν μέσω του σπέρματος. Οπότε θα πρέπει να επικαιροποιήσουμε τους κανόνες μας για να αποφύγουμε τη μετάδοση νόσων μέσω σπέρματος αναπαραγωγής, από κέντρα αναπαραγωγής. Επίσης έχουμε διεύρυνση του πεδίου εφαρμογή ώστε να καλύπτονται και άλλες νόσοι που δεν είναι τόσο γνωστές Και αυτό είναι το περιεχόμενο της τέταρτης κατεξοδότησης πράξης. Επίσης προβλέπεται η καταγραφή και η έγκριση των κέντρων αναπαραγωγής ε, από τις αρμόδιες αρχές. Και λέμε τι αρχή θα πρέπει να κρατά ο επιχειρηματίας σε περίπτωση προβλήματος ώστε να εξασφαλιστεί η χνηλασιμότητα της προέλευσης του σπέρματος ή του εμβρίου σε αυτά τα κέντρα γονιμοποίησης. Ε, καλύπτονται και άλλα προϊόντα σπέρματος ε, για γάτες, σκύλους, ε, για ένα παραγωγικό υλικό που βρίσκεται σε τράπεζες και επίσης προβλέπεται και κοινοποίηση του εμπορίου τέτοιων προϊόντων μέσω του ολοκληρωμένου συστήματός μας που επιτρέπει την εχνηλασιμότητα των ζώων των ζώων, των ζωντανών ζώων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει απόλυτη διαφάνεια, όλα αυτά που σας είπα υπάρχουν και στην ιστοσελίδα μας. Και εδώ ολοκληρώνεται η παρουσίαση του πακέτου των τεσσάρων κατεξοδότηση πράξεων. Πολύ ωραία. Μόνο τρεις ε, συνάδελφοι έχουν ερωτήσεις. Ε, προφανώς ήσασταν ιδιαίτερα κατατοπιστικός. Η κυρία Μαγκίνες, α, ε, μισό λεπτό, και άλλοι υποβάλλουν ερωτήσεις. Η κυρία Μαγκίνες είναι η πρώτη που θα κάνει την ερώτηση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και την Επιτροπή για την παρουσίαση και το συνάδελφο που ζήτησε να γίνει αυτή η παρουσίαση. Μια γενική παρατήρηση. Είναι πολύ δύσκολο για την Επιτροπή στο τέλος της διαδικασίας να κατανοήσει τις πράξεις που έγιναν μέσα σε μια κατεξοδότηση πράξη. Και ε, πρέπει να τη δούμε λιγάκι τη διαδικασία, να δούμε αν μπορούμε να τη βελτιώσουμε, γιατί τελικά τι γίνεται. Παίρνουμε την πληροφορία όταν πια έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Τέλο πάντων, θα τα δούμε αυτά κάποια άλλη μέρα. Εμένα ε, θα με ενδιέφερε ε, η επικαιροποίηση των πληροφοριών για τα πρόβατα και τις έγιες που αναφέρατε. Εγώ έρχομαι από την Ιρλανδία. Θα γνωρίζετε ότι υπάρχουν πολλές ανησυχίες ε, σχετικά με ένα συγκεκριμένο θέμα που αφορά στο νόμο για την υγεία των ζώων που προβλέπει ε, τεστ 30 ημών εκτός εάν το ζώο είχε μία δοκιμή για TB ε, Υπάρχει λοιπόν μια γενικότερη ανησυχία ότι αυτό είναι μια πολύ γενικευμένη, ε, μη στοχευμένη προσέγγιση. Καλύτερα θα ήταν να, έχουμε, να στοχεύουμε σε εκείνες τις αγέλες ε, που έχουν πραγματικό πρόβλημα. Γιατί το 97% δεν έχουν εφηματίωση, αλλά υπάρχει και πρόβλημα εφηματίωση που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Κάτι πρέπει να γίνει. Το δικό μου το ερώτημα είναι δεν, θα ήταν, δεν είναι καλύτερα να έχουμε έτσι μια στοχευμένη προσέγγιση από μια γενικότερη, γενικευμένη Κατά την άποψή μου, εδώ έχουμε δύο επιλογές. Ε, είχαμε μια συζήτηση στους ε, συντονιστές, ίσως να αναβληθεί το θέμα. Για μένα όμως είναι σημαντικότερο το να διορθώσουμε τα κακό κείμενα. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει στοχευμένη προσέγγιση ή να δούμε κατά πόσον οι έξι μήνες μπορούν να επεκταθούν και στους 12 μήνες. Γιατί υπάρχουν θέματα τα οποία επηρεάζουν πάρα πολύ την εκμετάλλευση, γραφειοκρατικά, κόστος. Ε, να το κάνουμε όπως κάνουμε και με τα ζώντα ζώα. Ε, υπάρχουν πολλά θέματα, όλα είναι σημαντικά, σημαντικό να ενημερωθούμε και επίσης ε, να εμπλέκεται και ο άμεσα ενδιαφερόμενος. Ε, πρέπει αυτό να το κατανοήσετε. Αν υπάρχει αντίδραση δεν θα πετύχουμε τίποτα. Ε, πρέπει όλοι οι γεωργοί κτηνοτροφοί να συμμετέχουν και αυτή τη στιγμή πρέπει να σας πω δεν το κάνουν. Αυτά τα αντιμετωπίζουν ως μια ανεπιθύμητη επιβολή ε, όρων στη δουλειά τους. Εγώ λοιπόν ρωτώ σχετικά με τη θυματίωση τι ακριβώς πιστεύετε ότι πρέπει να κάνουμε. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Δεν είμαι μέλος της Επιτροπής, αλλά με ενδιαφέρει το θέμα. Κάποια σημεία να θίξω. Θέλω περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ. Καταρχάς, στη διαδικασία διαβούλευσης για την υγεία όσον αφορά τους εμπλεκομένους φορείς. Εκφράστηκαν ανησυχίες για αυτή την πρόταση, σημαντικές θα επιβάλλει βάρος στις μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις, στις εκμεταλλεύσεις στην Ιρλανδία. ε, είναι πρόβλημα η φυματίωση, πρέπει να κρυζωθεί. Αλλά εδώ τα μέτρα έπρεπε να στοχεύουν τα κοπάδια που αντιπροσωπεύουν μεγάλο κίνδυνο. Οι μικρές εκμεταλλεύσεις είναι μικρού κινδύνου. Επιβαρύνονται οι οικογενειακές, οι μικρέ επιχειρήσει. Πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι από δοκιμές ετήσιες πάμε σε εξαμηνίες δοκιμές στα κοπάδια. Στην Ιρλανδία ένα ζώο μπορεί να μετακινηθεί τέσσερις-πέντε φορές στη διάρκεια της ζωής του πριν σφαγιαστεί. Άρα θα έχουμε πολλαπλές μετακινήσεις. Και αυτό θα επηρέαζε πολύ αρνητικά τις μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις που αντιδρούν στις συνθήκες αγοράς. Θέλουν να πουλήσουν το ζώο τους γρήγορα σε σύγκριση με το προσχεδιασμένο αυτό προγραμματισμό για πώληση. Γιατί από ετήσια πάτε σε εξαμηνία ε, δοκιμή στα ζώα με δοκιμές 30 ε, ημέρες πριν τη μετακίνηση και 30 μέρες μετά υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία να το στηρίζουν. Όπως είπε και η κυρία Μαγκίνες, οι γεωργοί στην Ιρλανδία θέλουν να εκριζωθεί η φυματίωση των βοηδών. 32 εκατομμύρια κάθε χρόνο πληρώνουν σαν εισφορά για φόρους για τις ζωασθένειες, για τις νονόσους και για τα κοπάδια τους. Θέλουν να εκριζωθεί η ασθένεια. Αυτό θα έχει πολύ όμως μεγάλο αντίκτυπο αυτό το μέτρο ε, στις οικογενειακές επιχειρήσεις και στη βιωσιμότητά τους. Χρειάζεται περισσότερη εξέταση, συζήτηση με τους ενδιαφερομένους και ανάλυση εκ νέου, πιστεύω. Ευχαριστώ, συνάδελφε Ζάντο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ που διοργανώσατε αυτή τη συζήτηση. Θέλω να επιμείνω επί της ανάγκης να θεθεί κάποια ευελιξία, να μην είμαστε πολύ άκαμπτοι για να είμαστε αποτελεσματικοί. Να δώσω ένα παράδειγμα. Η κατηγοριοποίηση ασθενειών σε θελοντικά προγράμματα εκρίζωσης ε, του, ε, της ασθένειας της καταρροής των, προβάτων προβλέπει ένα πρόγραμμα, πρέπει να καταπολεμηθεί όλη όλα τα μικρόβια που προξενούν αυτή την ασθένεια. Η καταπολέμηση ασθένειας περνά μέσω και εμβολιασμού. Δεν υπάρχει διαθέσιμο όμως εμβόλιο στην Ευρώπη για την καταρροή αυτή νόσο των προβάτων και αυτού του είδους τα μικρόβια. Ποιος είναι ο κίνδυνος πολλαπλασιασμός των απαιτήσεων όσον αφορά τις μετακινήσεις των ζώων, ανάλογα με τις καταστάσεις, όχι μόνο την παρουσία των διαφόρων ιών ή δυνατότητα να καταπολεμηθεί η ασθένεια. Πώς μπορούμε να επιτρέψουμε μια διαχείριση πιο ευέλικτη. Κατά σειρότυπο και πώς μπορεί να γίνει αυτός εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο επίπεδο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Λοιπόν, για να είμαστε αποτελεσματικοί θα πρέπει να προσαρμοστεί η μέθοδος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλύει την κατάσταση. Μήπως μπορεί βάση, τα μέτρα να λαμβάνονται βάσει αποτελεσμάτων, όχι βάσει των μέσων. Στην νομοθεσία λοιπόν να αναγνωρίζετε, τα, να αναγνωρίζετε τα προγράμματα τα οποία έχουν ισοδύναμα αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Συνάδελφε Μέτς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα μιλήσω τώρα αγγλικά ε, για να αποφευθεί ο μαζικός σφασμός ο μαζικός φαγισμός ε, των ε, ε, ζώων όταν μετακινούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση νομίζω ότι χρειάζονται περισσότερα προληπτικά μέτρα. Παραδείγματο χάρη να περιστεί η βιομηχανική κτηνοτροφία, να υπάρχει υπευθυνότητα απέναντι στο περιβάλλον και στην μη επέκταση των ασθενειών. Γι' αυτό λοιπόν ερωτώ, τα κοπάδια και η ε, ευζοία των ζώων πώς μπορούν να ενταχθούν μέσα στην έννοια της ευβιωσιμότητας και της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Και έχω και κάποιες άλλες ερωτήσεις. Μιλήσατε για τις μετακινήσεις των ζώων. Για να μπορεί κανείς να εγγυηθεί την ζωή ε, των ζώων σε γενικές γραμμές, πιστεύετε ότι οι έλεγχοι που γίνονται στα κράτη-μέλη είναι επαρκείς. Συνάδελφος Μπούντα, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε, ε, μιλήσατε και για την Αφρικανική Πανόλη των Χείρων ε, και θα ήθελα να γνωρίζω ποια είναι τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και να επισημάνω το εξής. Υπάρχουν προβλήματα που βασίζονται στην παραδοχή ότι αυτή η ασθένεια θα μπορούσε να λάβει τη μορφή επιδημίας. Ε, στην περίπτωση αυτή ερωτώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τις απαραίτητες εγκαταστάσεις ε, για, το κάψιμο, για την κάψη των ζώων, γιατί δεν υπάρχουν αρκετές εγκαταστάσεις ε, για την περίπτωση που πρέπει να καταπολεμηθεί αποτελεσματικά ο ιός. Πώ είναι δυνατόν, παραδείγματο χάρη, να έχουμε εδώ και αρκετό καιρό την ασθένεια των πτηνών στην Πολωνία ε, και έχουμε πολύ συχνά μολυσμένο κρέας στη Ρουμανία. Γιατί δεν υπήρξε άμεση παρέμβαση στα σφαγεία όπου εμφανίστηκε αυτός ο ιός. Και γιατί έπρεπε να ε, περιμένουμε μέχρι να εμφανιστούν ε, ε, τα προϊόντα μεταποίηση σε άλλες χώρες. Νομίζω ότι θα ήταν καλό να εμφαρμόζεται τα μέτρα στην πράξη και όχι απλά να τα παρουσιάζετε σε διαφάνειες και ομιλίες. Σάλφος Ρούσεν. Ευχαριστώ. Στην πατρίδα μου, τις κάτω χώρες, ο κλάδος, οι κτηνοτρόφοι έχουν παραπονεθεί ότι η κατεξιδότηση πράξη θα αποτελέσουν φραγμό στο εμπόριο γιατί είναι πολύπλοκες, περίπλοκες και δύσκολες εφαρμογής. Υπάρχουν πολλά προβλήματα κυρίως για τα βοηδή, γιατί για τα μοσχάρια, για παράδειγμα, έχουμε ε, καραντίνα 40 ημερών. Αυτή η καραντίνα όμως δεν χρειάζεται για τις περιπτώσεις της νόσου IBR που ελέγχεται πολύ καλύτερα. Γιατί την ρινοτραχεΐτιδα, την λιμόδι ρινοτραχεΐτιδα των βοηδών Οπότε ίσως ε, την καραντίνα των 40 ημερών θα μπορούσαμε να την ε, περιορίσουμε σε 30 μέρες για νόσου που είναι εύκολες. Ε, εύκολο ελέγχο όπω η IBR, η ρευδραχύτητα των βοηδών. Πολύ ωραία. Αν δεν έχετε άλλε ερωτήσει, θα δώσω το λόγο στον εισηγητή μα για να απαντήσει σε αυτά που ελέγχθησαν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να απαντήσω στους συναδέλφους από την Ιρλανδία Τι θέλουμε. Τι θέλουμε όλοι. Εκρίζωση της ε, φυματιώσεως από την Ιρλανδία Σε δύο κράτη-μέλη η κατάσταση δεν είναι καλή. Από τον επόμενο μήνα θα είναι μια χώρα. Θέλουμε να βοηθήσουμε την Ιρλανδία. Και γι' αυτό δίνουμε πολλά χρήματα στην Ιρλανδία για την εκρίζωση της φυματιώσεως. Και ένας από τους λόγους που αναφέρατε κι εσείς για αυτό το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν πολλές μετακινήσεις κοπαδιών. Α, είχατε πρόβλημα με τα γερμανικά. Με τη διερμηνία δεν περνάει, τεχνικό πρόβλημα. Εντάξει, διορθώθηκε το τεχνικό πρόβλημα. Έλεγα λοιπόν, ότι ένας από τους λόγους που αναφέρθηκε και τονίστηκε από τους εκπροσώπους της Ιρλανδίας είναι ότι υπάρχουν πολλές μετακινήσεις κοπαδιών μεταξύ εκμεταλλεύσεων στην Ιρλανδία. Και σίγουρα ένας από τους λόγους, ίσως όχι μοναδικός, αλλά ένας από τους λόγους για τους οποίους είναι πολύ δύσκολο να εκριζωθεί η φυματίωση στην Ιρλανδία Δώσαμε πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο τα τελευταία χρόνια για να βοηθήσουμε την Ιρλανδία να εξαλείψει τη φυματίωση και θα εξακολουθήσουμε την προσπάθεια. Τι κάναμε. Βασιστήκαμε στις κατευθείαν γραμμές του Οργανισμού Υγείας και την εμπειρία του Διεθνές Γραφείου Επιζωτιών και τα διάφορα προγράμματα που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση επί σειρά ετών και στην Ιρλανδία όλες οι παρεκκλήσεις χρησιμοποιήθηκαν από την προηγούμενη νομοθεσία για να καθυστερήσουμε τις δοκιμές. Στη νέα κατοξιδότηση πράξη που δεν θα ισχύσει τώρα, αλλά τον Απρίλιο του χρόνου, εκεί λοιπόν σε αυτή την πράξη λέμε ότι όταν τα κοπάδια δοκιμάστηκαν, ελέγχθηκαν τους τελευταίους έξι μήνες δεν απαιτείται μετά ξεχωριστή ανάγκη για έλεγχο αν μετακινηθεί ένα ζώο, αν είσαι σε μια συγκεκριμένη περιοχή, αν είσαι σε περιοχή περισσότερο μολυσμένη από άλλες, αν είσαι σε άλλη περιοχή, μπορείς να παρεκκλίνεις μέχρι ένα χρόνο. Λεπτομερέστατοι οι κανόνε. Δεν χρειάζεται να αναφέρω όλε τι λεπτομέρειε τώρα. Με τα χαράς να σας συναντήσω και τους γεωργούς να τα εξηγήσουμε. Να δούμε αν μπορούμε να βρούμε μέσω του προγράμματος να βρούμε λύση. Θα εξακολουθούμε να χρηματοδοτούμε, βλέπετε, το πρόγραμμα εκρίζωσης Ιρλανδίας και το 2020 να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε καλύτερα τους Ιρλανδούς γεωργούς που πραγματικά, τους, τους κοινοτρόφους που θέλουν να ε, εκριζώσουν την ε, φυματίωση. Αυτό θέλουν όλοι και την ιατρική υπηρεσία της Ιρλανδίας και εμείς. Όλοι αυτό το στόχο έχουμε. Σχετικά με την εκρίζωση άλλης ασθενείας του καταρροϊκού πυρετού των προβάτων πράγματι έχουμε 24 οροτύπους που υπάρχουν και κάποιοι ορότυποι επηρεάζουν τα ζώα, όχι σε κάποιες χώρες. Η Γαλλία έχει ένα-δύο διαφορετικούς ορότυπους και πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι μέσω εμβολιασμών εκτινοτρόφοι δεν θα υποφέρουν από την ασθένεια αυτή, τον καταδικό πυρετό των προβάτων. Κατά το παρελθόν είχαμε τεράστια επιδημία στη Γαλλία, πέρασε μετά Ολλανδία, Βέλγιο και λόγω εμβολιασμών, χάρη στους εμβολιασμούς, σώσαμε τους κτηνοτρόφους από σοβαρές απώλειες και θα συνεχίσουμε να παρέχουμε την αναγκαία και απαραίτητη υποστήριξη στους κτηνοτρόφους για να αποφύγουν την καταστροφική συνέπεια αυτής της ασθένειας στην Ευρώπη και με την αλλαγή του κλίματος και τις συνέπειες αυτής της αλλαγής όλο και περισσότερο θα πληγούν οι βόρειες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Για τη βιομηχανική κτηνοτροφία εξαιρετισμό μεταξύ ευημερίας των ζώων και υγείας των ζώων υπάρχει σχέση. Στην Πράσινη Συμφωνία θα το αναλύσουμε αυτό σε σχετική στρατηγική που θα παρουσιαστεί ε, προς το τέλος της Άνοιξης. Υπάρχει συσχετισμός πράγματι, αλλά όπως ανέφερα αυτή η σχέση δεν εντάσσεται αυτόν τον κανονισμό, δεν συμπεριλαμβάνεται. Νομίζω ότι στην πρώτη διαφάνεια το είπα ξεκάθαρα ότι αυτός ο κανονισμός δεν καλύπτει την ευμερία των ζώων. Το θέμα αυτό της καλής κατάστασης των ζώων θα αντιμετωπιστεί από, στην στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το χωράφι στο πιάτο. Τώρα, όσον αφορά την πανόλη των χείρων είναι μεγάλο πρόβλημα. Η αφρικανική πανόλη των χείρων. Θα απαντήσω στην ερώτηση μετά, διότι θα παρουσιάσω την κατάσταση του αυθόδη πυρετού των χείρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επίσης ε, τη γρήπη των πτηνών, οπότε σίγουρα θα έχετε μία απάντηση από την παρουσίαση που θα κάνω. Δεν ξέρω τις λεπτομέρειες για την καραντίνα των 30 ε, ημερών για τα μοσχαράκια ε, στην ε, Ολλανδία. Θα το συζητήσουμε αυτό μετά τη συνεδρίαση. Σκοπός του κανόνα είναι η διευκόλυνση της καταστάσεως, η απλούστευση, ταυτόχρονα διατηρώντας υψηλό επίπεδο της υγείας των ζώων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνδυάζουμε διάφορα νομοθετήματα σε μερικές πράξεις, λίγες πράξεις. Το κάναμε αυτό σε τέλεια εναρμόνιση συντονισμού με τα κράτη-μέλη. Θέλουμε να συνεχίσουμε να είμαστε αρρωγοί, θέλουμε να διατηρήσουμε τα υψηλά επίπεδα υγεία των ζώων και να υποστηρίζουμε τα κράτη-μέλη που αντιμετωπίζουν δυσκολίες για την επίτευξη αυτού του επίπεδου, όπως η Ιρλανδία για τη φυματίωση και πολλά άλλα κράτη-μέλη για άλλες ασθένειες. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς ε, για ε, όλα αυτά που μας είπατε. Συνάδελφος Μαγκίνες ε, θέλει και πάλι το λόγο. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας ευχαριστώ θερμά για τις διεξοδικές απαντήσεις σας. Ε, να κάνω μια ερώτηση και μια διευκρίνηση. πολύ ωραία αυτά που είπατε ότι θα μιλήσετε με τους εκπροσώπους των κτηνοτροφικών μονάδων για να δείτε αν μπορεί να εξευρεθεί κάποια λύση. Θα πω κάτι για τη χρηματοδότηση, γιατί βεβαίως η εξάλληψη των ασθενειών προέρχεται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, για το Ιρλανδικό πρόγραμμα δόθησαν 27 εκατομμύρια ευρώ και για το 20 προβλέπονται 5,4 εκατομμύρια. Ε, γι' αυτό ρωτώ μήπως υπάρχει αύξηση των ασθενειών επειδή αυξάνονται και τα κονδύλια. Ξέρω βέβαια ότι υπάρχουν υπάρχει πίεση στον προπολογισμό ε, και κάπως πρέπει να είσαστε πιο στοχευμένοι. Ε, σας παίρνω κατά λέξη, το, ε, θεωρώ ότι δεσμεύεστε αυτό που είπατε, ότι πραγματικά θα λάβετε μέτρα για να δείτε πώς μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση. Τόντι μπορείτε να θεωρήσετε ότι είναι λόγος τιμής. Παρακαλώ. Πάρα πολύ σύντομα. Χαιρετίζω αυτά που μας είπατε, τις εξηγήσεις, αλλά ε, το θέμα είναι ότι ε, η θέση στην οποία θα βρεθούν ε, οι Γεωργοί, αυτό είναι το σημαντικό. Δεν είναι απλά ανησυχία. Αυτοί που συμμετέχουν στην παραγωγή, στην εκτροφή στην Ιρλανδία ανησυχούν πάρα πολύ. Και σωστά είπε κύριε Μακίνης, αν πρόκειται να κάνουμε περισσότερα τεστ, ε, και αυξηθούν τα ποσοστά ε, ασθενειών, θα πρέπει να αυξηθούν οι δαπάνες και από τα Εθνικά Υπουργεία αλλά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί αν κάνουμε αυτά που λέτε, υποτίθεται θα εντοπίζουμε περισσότερες ασθένειες, αλλά με βάση αυτά που βλέπουμε είναι ότι εντοπίζονται λιγότερες ασθένειες. Μας ανησυχούν πάρα πολύ αυτές οι προτάσεις, ε, γιατί αλλιώς οι κτηνοτρόφοι είναι εκείνοι οι οποίοι θα κληθούν να χρηματοδοτήσουν εξ ολοκλήρου το πρόγραμμα κάτι το οποίο είναι άδικο θα έλεγα. Κοιτάξτε, ε, αν θέλετε να σας δείξω τα στοιχεία. Για μένα λοιπόν στην ε, Ολλανδία ε, τα φαινόμενα θα αυξηθούν περισσότερο αντί να μειωθούν. Ε, το θέμα είναι, ο στόχος είναι να εξαλείψουμε την ε, φυματίωση στην Ιρλανδία. Ήδη έχουμε κάνει πάρα πολλά για να βοηθήσουμε τις αρμόδιες αρχές να σχεδιάσουν ένα πρόγραμμα το οποίο θα ταιριάζει στη συγκεκριμένη περίπτωση στην Ιρλανδία. Αυτό δηλαδή που είπατε, ότι τα ζώα μετακινούνται μέχρι και έξι φορές ε, κατά τη διάρκεια της ζωής τους από το ένα κοπάδι στο άλλο πριν ε, φτάσουν στο σφαγείο. Πολύ ωραία λέει ο πρόεδρος. Ε, Άλφα Φλάνιγκαν, αν την καλοσύνη όμως να είστε πολύ σύντομος. Θα είμαι σύντομος. Χαίρομαι που ε, υπάρχει τέτοια υποστήριξη για την πρόταση που υπέβαλε η Γκουε. Νομίζω ότι είναι πολλά τα ωφέλη από την πρόταση αυτή. Πρόεδρος, να σας ενημερώσω ότι οι συντονιστές ε, σήμερα ε, παρέτειναν ε, κατά δύο μήνες τη δυνατότητα κατάθεσης ενστάσεων, άρα δηλαδή θα έχουμε ακόμα δυνατότητα για να συζητήσουμε για το θέμα αυτό. Πάμε τώρα στο σημείο υπερθμών 11, ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την Αφρικανική Πανόλη των Χείρων. Γνωρίζετε όλοι σας ότι σε διάφορα κράτη-μέλη ήδη έχουν εμφανιστεί τέτοια κρούσματα, κυρίως τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Λιθουανία αλλά και την Πολωνία. Εχθές, σε παραδείγματος χάρη, μου ανέφεραν ότι και στην Πολωνία 12 ε, χιλιόμετρα μακριά από τη δική μου τη γενέτειρα που είναι στη Γερμανία έχουμε κρούσματα. Ε, κάθε μέρα λοιπόν ε, έχουμε ειδήσει όπου βλέπουμε ότι εξαπλώνεται όλο και περισσότερο αυτή η ασθένεια. Πρόκειται ως εκ τούτου για ένα ιδιαίτερα επίκαιρο θέμα που μπορεί να έχει πολύ δυσάρεστες προεκτάσεις. Ε, και γι' αυτό λοιπόν σας δίνω και πάλι το λόγο για να μας παρουσιάσετε την κατάσταση στην Ευρώπη αλλά και στα μέτρα ε, τα οποία λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλώς. Θα σας εξηγήσω το εξή. Τι, τι είναι αυτός ο ιός, πώς έχει παγκόσμια κατάσταση, πώς έχει κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τι επιτυχίες έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα, ποιες, ε, ποια είναι αυτά τα παθογόνα μεγάλων αποστάσεων τα περίφημα, επιρροή στην υγεία και πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εδώ και πάρα πολλά χρόνια για την αντιμετώπιση της ζώνος αυτής. Ποιος είναι ο ιός λοιπόν. Δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειες. Πρέπει να ξέρουμε όμως ότι έχουμε σίγουρο θάνατο από τη στιγμή που μολύνεται το ζώο. Είναι πολύ αποτελεσματικός ο ιός που σχεδόν ε, σκοτώνει το 100% των ζώων που μολύνει και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ε, και κυρίως ε, από τους αγριόχειρους περνάει. Ο ιός αυτός είναι πολύ πιο αποτελεσματικός στους αγριόχειρους. Θα πρέπει από τη στιγμή που εμφανιστεί κρούσμα να τον περιορίσουμε τους αγριόχειρους στην περιοχή, γιατί ούτε θεραπεία υπάρχει ούτε εμβόλιο και χτυπάει μόνο τους χείρους. Αγριόχειρους και χείρους. Κανένα άλλο ζωικό είδος δεν προσβάλλεται από τον ιό αυτό. Πώς έφτασε στην Ευρώπη η Αφρικανική Πανόλη των Χείρων, γιατί είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στην Αφρική. Στην Αφρική υπάρχει παντού. Είναι γενικευμένη. Είναι τόσο παντού που δεν τη βλέπουν καν και περνά μέσω από την ε, ε, ε, το χυλό που τρώνε τα, τα ηχείρη, κάτι που έχουμε ε, καταργήσει εδώ και 30 χρόνια. Είναι η υπόλοιπα τροφών, υπόλοιπα φαγητού που εδώ και 40 χρόνια καταστρέφουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά στην Αφρική τα χρησιμοποιούν για τροφή. Το ίδιο και στην Γεωργία. Χρησιμοποιούνται ακόμη αυτά τα υπόλοιπα τη κουζίνα. Χρησιμοποιούνται αυτά τα υπόλοιπα των τροφίμων για, να, για χειροτροφή. Έτσι εξαπλώθηκε η νόσος στην Ευρώπη. Ξεκίνησε από τη Γεωργία που εξακολουθούν να χρησιμοποιούν για χειροτροφή τα υπόλοιπα των τροφίμων και μέσω του πληθυσμού αγριοχείρων και της μετακίνησης ε, μολυσμένο κρέατος εξαπλώθηκε και στην Ευρώπη η νόσος αυτή. Θα σας δείξω ένα βίντεο από τον Ιανουάριο του 2014 όταν εντοπίστηκε το πρώτο κρούσμα στα σύνορα Λιθουανίας-Πολωνίας και βλέπετε την επέλαση της νόσου μήνα με το μήνα. Και βλέπουμε και τις περιοχές που έχουν μολυνθεί μπλε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πορτοκαλί είναι το χρώμα των περιοχών που έχουν μολυνθεί στην Ασία. Και μέχρι τα τέλη του 2018, μέχρι πρόσφατα δηλαδή, ε, ξεκίνησε και από την Κίνα και από εκεί μεταδόθηκε σε όλη την Νοτιοανατολική Ασία. Μέχρι στιγμής δηλαδή όλο το νοτιοανατολικό τμήμα της Ασίας έχει μολυνθεί από τον ιό της Αφρικανικής Πανόλης των Χείρων. Πώς έχει κατάσταση φέτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εν έτη 2020. Βλέπετε τις πράσινες κουκίδες που είναι οι μολυσμένοι αγριόχειροι που έχουν εντοπιστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κίτρινες κουκίδες είναι οι φάρμες που έχουν κρούσματα αφρικανικής πανόλης χείρων. Στην Εστονία, στην Λετονία έχουμε πολλά κρούσματα. Ε, ήδη εδώ και πολλά χρόνια. Και επειδή έχουν αποδεκατιστεί αγριόχειροι, έχουν ελάχιστους ε, ζωντανούς πια αγριόχειρους στις περιοχές αυτές, οπότε ε, το φορτίο του ιού στο περιβάλλον στην Εστονία και Λετωνία είναι πολύ χαμηλό. Γιατί, επαναλαμβάνω, οι αγριόχειροι που είναι οι πιο επιρρεπείς έχουν εξολοθρευθεί από την όσο. Πριν το 2014, στην Εστονία, είχαμε πάνω από 1.300 φάρμες. Τώρα έχουν απομείνει 130 περίπου φάρμες στην Εστονία χειροτροφία με υψηλή ζώνη ασφάλειας γύρω από τις φάρμες και με απαγόρευση οποιασδήποτε επαφής μεταξύ άγριων και οικόσιτων ζώων. Ρουμανία και Βουλγαρία. Ε, έχουμε ακόμη πολλά κρούσματα, κυρίως από τα οικόσιτα ζώα. Τα οικόσιτα ζώα είναι μεγάλη πρόκληση για την Αφρικανική Πανόλη των Χείρων, γιατί ελάχιστα μέτρα βιοασφάλειας χρησιμοποιούνται από τους μικρούς κτηνοτρόφους για να αποφευθεί η επαφή άγριων ζώων με τα οικόσιτα γουρούνια. Γι' αυτό έχουμε μεγάλη μόλυνση στη Βουλγαρία και Ρουμανία. Επίσης έχουμε μια περιοχή γύρω από την Ουγγαρία, τη Σλοβακία και την Ουκρανία, εκείνη η γωνία που βλέπετε. Και στην περιοχή αυτή είχαμε πολλά μολυσμένους αγριόχειρους στα δάση. Και βλέπετε τις μικρές κουκίδες ε, στο νότιο Βέλγιο όπου είχαμε σε ένα δάσος κάποια κρούσματα ε, λόγω του ανθρώπινου παράγοντα και οι βελγικές και οι γαλλικές αρχές τότε ανέλαβαν ε, πολλές δράσεις και μέτρα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πια ιός στο Βέλγιο. Το ίδιο συνέβη και στη Τσεχία πέρυσι. Και έχουμε και μια κουκίδα σαν την Τσεχία και το Βέλγιο έχουμε παρόμοια κουκίδα στη Δυτική Πολωνία, πολύ κοντά με τα γερμανικά σύνορα. Και εκεί είχαμε μόλις κρούσμα σε ένα δάσος. Τώρα, πώς τα γνωρίζουμε αυτά και γιατί υπάρχουν σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και όχι αλλού τέτοια κρούσματα. Καταρχήν, η Τσεχία έχει κηρυχθεί ε, χωρίς ιό από τις ε, αρχές του περασμένου έτους. Και αυτή τη διαδικασία εφαρμόζουν τώρα και στο Βέλγιο για να κηρυχθούν ως ελεύθερη από νόσο περιοχή και χώρα. Βλέπετε πάρα πολλά κρούσματα σε 20 ζώα. Έχουμε την μπλε στήλη στη Ρουμανία που είχαμε ε, λόγω των 20 των ζώων πολλά κρούσματα. Ξεκίνησαν αυτά στο Δέλτα του Δούναβη στο βόρειο τμήμα δηλαδή της Ρουμανίας, στα σύνορα με την Ουκρανία και από εκεί η νόσος εξαπλώθηκε σε όλη τη Ρουμανία. Τώρα, Τσεχία. Στη Τσεχία έχουμε κρούσμα όπως και στο Βέλγιο και στην Πολωνία. Ανακαλύφθηκε ε, η νόσος λόγω του ανθρώπινου παράγοντα, δηλαδή κάποιος κάπου με κάποιο τρόπο κατάφερε να μολύνει έναν αγριόχειρο στο δάσος, δίνοντάς του να φάει σαλάμι, κάποια τροφή που περίχε μολυσμένο κρέας. Το έπιασαν όμως στην αρχή το πρόβλημα, στη Τσεχία, Βέλγιο και Πολωνία και απαγόρεψαν το κυνήγι στην περιοχή, έλαβαν έκτακτα μέτρα και περίμεναν μέχρι να οριοθετηθεί η κατάσταση της μόλυνσης, γιατί οι αγριόχειροι κινούνται λίγο, αλλά πολύ περιορισμένα. Και από τη στιγμή που χαρτογραφήθηκε με την υποστήριξη των εμπειρογνωμόνων η ακριβής περιοχή της μόλυνσης ε, στην Τσεχία, την ε, περιέφραξαν και άφησαν τους αγριόχειρους να κυκλοφορούν εκεί είτε θα τους νικούσε η αρρώστια είτε θα νικούσε την αρρώστια αλλά τελικά δεν κράτησε πολύ ο ιός εκεί και η Τσεχία απαλλάχθηκε από τον ιό. Βέβαια, σε νεκρό ζώο μέχρι 6 μήνες επιβιώνει ο ιός. Και σημαντικό έργο των αρμοδίων αρχών είναι να συγκεντρώσουν τα νεκρά σφάγια στο δάσος, τα νεκρά σφάγια των αγριοχείρων στο δάσος, για να αποφευθεί η μόλυνση του ιού σε άλλα ζωντανά ζώα. Το ίδιο και στο Βέλγιο. Έγινε περίφραξη που χρειάστηκε να επεκταθεί από την αρχική ζώνη, γιατί η νόσος επεκτάθηκε και πέραν των φραχτών, οπότε χρειάστηκε διαδοχικά να επεκτείνουν τους φράχτες. Τελικά κατάφεραν και την περιόρισαν την νόσο και κατασκευάστηκαν φράχτες και νοτιοδυτικά του Βελγίου για να προστατευτεί κυρίως η Γαλλία και να αποφευχθεί μετάδοση της Αφρικανικής Πανόλης των Χείρων και στη Γαλλία. Και οι Γάλλοι από τη δική τους πλευρά επίσης κατασκεύασαν φράχτες για να οριοθετηθεί η μόλυνση στα σύνορα με το Βέλιο και να μην περάσει στη Γαλλία. Βέβαια, η αρρώστια, όπως είπα, αποδεκατίζει τα μολυσμένα ζώα, αλλά αποδεκατίζει και το εμπόριο. Είναι ολέθρια τα αποτελέσματα της νόσου και για το εμπόριο. Τώρα, τι έγινε στη Δυτική Πολωνία. Το πρώτο κρούσμα επιβεβαιώθηκε στα μέσα Νοεμβρίου και αμέσως στείλαμε την έκτακτη ομάδα ακτινιάτρων μας. Πρόκειται για ομάδα εμπειρογνωμόνων κτηνιάτρων από τα κράτη-μέλη. Είναι κτηνίατροι που εργάζονται είτε σε ερευνητικά κέντρα είτε σε Ινστιτούτα και είναι απόλυτα εξοικειωμένοι με τη συμπεριφορά των άγριων ζώων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μπορούν να δώσουν τεκμηριωμένες συμβουλές στα κράτη-μέλη ε, για να αποφύγουν την εξάπλωση της νόσου. Και είναι γνωστή σε όλο τον κόσμο για παροχή συμβουλών στις αρμόδιες αρχές σε περίπτωση εμφάνισης ζώων νόσου. Οπότε εδώ προβαίνουμε σε μια αποκέντρωση, μια περιφερειοποίηση, ώστε να περιορίσουμε την αρρώστια και να μην εξαπλωθεί περαιτέρω. Δεν ε, εντοπίστηκαν άλλα κρούσματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, από το εμπόριο. Όλα τα κρούσματα που καταγράφησαν προέρχονταν από παράνομες δραστηριότητες. Από νόμιμο εμπόριο κανένα κρούσμα δεν προέκυψε. Και στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, όλες οι αρμόδιες αρχές τουλάχιστον δύο φορές το μήνα επικοινωνούν μαζί μας και με μερικές αρμόδιες αρχές έχουμε και καθημερινή επικοινωνία. Ποιος είναι ο αντίκτυπος τώρα. Όπως βλέπετε, ο αντίκτυπος είναι απειλή όχι μόνο στα κοπάδια, στην κτηνοτροφία, αλλά και στην άγρια πανίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και του κόσμου. Επηρεάζει αρνητικά και τις, τους περιορισμούς και το εμπορικό εμπάργκο που έχει επιβληθεί σε πολλές χώρες. Υπάρχει μεγάλη επαγρύπνηση, ιδιαίτερα στην Βόρεια και Νότια Αμερική. Η Αμερική, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία είναι τα μόνα μέρη του κόσμου που δεν έχει εμφανιστεί καθόλου η νόσος αυτή. Και γι' αυτό έχουν εκστρατείες επαγρύπνησης, ενημέρωσης και πολλές δραστηριότητες για να αποφύγουν οπωσδήποτε την είσοδο της νόσου στις υπήρους αυτές. Λοιπόν, βλέποντας τι αντίκτυπο έχει όλο αυτό στο εμπόριο, για να πάρετε μια ιδέα για παραγωγή κρέατος περίπου 260 κομμάτια ε, χείρι σφαγιάστηκαν, εκατομμύρια χείρι σφαγιάστηκαν στην Ευρώπη ε, λιγότερο από ένα εκατομμύριο την ημέρα και σε μια διάσκεψη την περασμένη εβδομάδα στο Βερολίνο το συζητήσαμε αυτό θα αναφερθώ εκτενέστερα αργότερα. Σας δίνω μια γενική εικόνα τώρα. Έλλειψη κρέατος στην Κίνα. Οι Κινέζοι έλεγαν ότι 27 εκατομμύρια τόνοι, εκατομμύρια τόνοι χειρίου κρέατος έλειπαν από την Κίνα για φέτος. 27 εκατομμύρια τόνοι, εκατομμύρια, δεν είναι 27 εκατομμύρια τόνοι λέω, χειρίου κρέατος θα λείψει από τους Κινέζους αυτή η ποσότητα φέτος. Αν όλες οι εισαγωγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης πηγαίνουν στην Κίνα και πάλι θα τους έλειπε χοιρινό στην Κίνα. Και για πρώτη φορά τον Αύγουστο του 2018 ανακοινώθηκε επίσημα αυτή η ασθένεια και είδατε πώς μεταδόθηκε στην Ασιατική Ήπειρο. Μεσοπρόθεσμα χρειάζονται διαστατικές αλλαγές όσον αφορά την κτηνοτροφία των χείρων σε όλο τον κόσμο. Για τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας έχω ξαναμιλήσει επανειλημμένα για αυτές. Εμείς ήμασταν έτοιμοι. Όταν είδαμε ότι οι πανόλοι των χείρων έφτασε, πλησίαζε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αναλάβουμε πρωτοβουλίες ετοιμότητας. Ξεκινήσαμε ελέγχου στα σύνορα και επίσης ελέγχαμε και τα αγριογούρουνα. Επικαιροποίησαμε την νομοθεσία μας, λάβαμε υπόψη επιστημονικές συμβουλές, λάβαμε περιφερειακά μέτρα. Αυξήσαμε τους ελέγχους στα σύνορα, εφαρμόσαμε συνδυασμένες πρωτοβουλίες για ευαισθητοποίηση στα σύνορα, στις περιοχές της μεθοριακές. Αυξήσαμε την ε, παρέμβαση ταχείας δράσης, το EUVETS, και επικαιροποιήσαμε επίσης και τις κατάλληλες βάσεις δεδομένων και της οργάνωσης για τα τρόφιμα και τη γεωργία. Θέλαμε γενική ευαισθητοποίηση, όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε όλη την Ήπειρο. Όσον αφορά την Αφρικανική Πανόλη των Χείρων. Βλέπετε στο χάρτη θα δείτε αργότερα, ότι υπάρχει μια μαύρη τρύπα, η Λευκορωσία στην Ευρώπη, που δεν δηλώνουν και δεν επιβεβαιώνουν κανένα τέτοιο, τέτοια κρούσματα. Παρόλο που βρίσκουμε πολλά μολυσμένα ζώα στην Πολωνία, στη Λιθουανία και στη Λετωνία, κοντά στα σύνορα με τη Λευκορωσία. Πρέπει να αντιμετωπιστεί το θέμα και ο Επίτροπος συνάντησε τον Υπουργό Γεωργίας της Λευκορωσίας την περασμένη εβδομάδα στα περιθώρια συνάντηση στο Βερολίνο για να του επιστήσει την προσοχή στο ζήτημα της διαφάνειας ότι χρειάζεται διαφάνεια για να αντιμετωπιστεί καλύτερα η εξάλληψη ε, των προβλημάτων αυτών. Πρόληψη εντοπισμός, έλεγχος, διαφάνεια. Στην ιστοσελίδα μπορείτε να βρείτε την παρουσίαση αυτή. Μπορεί να διανεμηθούν επίσης τα έντυπα αν χρειαστεί στα μέλη. Έχουμε την ΕΦΣΑ που έπαιξε και αυτή κρίσιμο ρόλο. Πρόσφατα δημοσιεύθηκαν κατάλληλα έγγραφα με συμβουλές για να βοηθήσουν εμά και τις αρμόδιες αρχές να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Περιφερειοποιούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κράτη-μέλη που έχουν πληγεί γνωρίζουν το χάρτη, τα χρώματα. Κόκκινο είναι οι περιοχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου έχουμε κρούσματα σε εκμεταλλεύσεις και στους αγριόχειρους. Περιοχές που έχουν πολλά κρούσματα και κυκλοφορεί ο ιός. Ροζ περιοχές. Εκεί έχουμε μόνο κρούσματα σε αγριόχειρους. Οι εκμεταλλεύσεις εκεί βελτίωσαν την ασφάλειά τους κατά των ασθενειών και δεν έχουμε κρούσματα στις εκμεταλλεύσεις και έχουμε γαλάζιες περιοχές που είναι και αυτές μολυσμένες αλλά είναι ζώνη απομόνωσης αν θέλετε. Γιατί έχουμε αυτές τις ζώνες απομόνωσης. Όταν εντοπίσουμε αγριόχειρο μολυσμένο Α, ξέχασα, στη γαλάζια περιοχή κάθε νεκρός αγριόχειρος που βρίσκεται αγριόχειρος αποστέλλεται σε εργαστήριο για εξετάσεις. Βλέπουμε τη διάδοση της ασθένειας λόγω των μετακινήσεων των αγριοχείρων. Και εάν δεν υπάρχει παρενόχληση στο περιβάλλον, θα διαδίδεται ε, η νόσος κατά ένα με δύο χιλιόμετρα το μήνα λόγω της μετακίνησης των αγριοχείρων. Σημαντική ε, η γαλάζια περιοχή για τους ε, εμπορευόμενους εταίρους μας, διότι η υπόλοιπη η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ελεύθερη από την ασθένεια. Λόγω των γαλάζιων τμήματων που είναι ζώνες απομόνωσης, καραντίνας, δίνουμε την εγγύηση. Δηλαδή, οι υπόλοιπε περιοχέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουν την ασθένεια και μπορούν να εμπορεύονται ελεύθερα όσον αφορά το χοιρινό και να εξάγουν το χοιρινό και σε άλλες χώρες που αναγνωρίζουν αυτή την περιφερειοποίηση. Καναδά, ΣΥΠΑ, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Τρινιδάδ, υπάρχουν πολλές χώρες που αναγνωρίζουν αυτή την αντιμετώπιση. Δυστυχώς όχι όλοι οι εμπορικοί εταιροί αναγνωρίζουν αυτή, αυτό το σύστημα που απομονώνουμε τι μολυσμένε περιοχέ και αυτοί οι εμπορικοί εταίροι που αναγνωρίζουν την περιφερειοποίηση απαγορεύουν την εισαγωγή, θα απαγορεύσουν την εισαγωγή κρέατος από τη Γερμανία, αν βρεθεί έστω και ένας μολυσμένος αγριόχειρος στη Γερμανία. Προσπαθούμε μέσω χωρικής απομόνωσης, που επικαιροποιείται εβδομαδία ή δύο φορές το μήνα, να παρακολουθούμε τα κρούσματα και προστατεύουμε με τις απομονώσεις τις υπόλοιπες περιοχές που είναι υγιείς και έτσι και τις εξαγωγές σε τρίτες χώρες. Βλέπετε λοιπόν Βλέπετε ένα μικρό κομμάτι του Βελγίου που είναι γαλάζιο και ροζ και μια περιοχή στην Πολωνία που και αυτή είναι μολυσμένη. Όλοι αυτοί οι χάρτες είναι στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής. Μιλούσα για την ομάδα εμπειρογνωμόνων. Τους ξέρουν πολύ καλά σε όλο τον κόσμο. Πήγαν στις χώρες εκείνες που βλέπετε για να βοηθήσουν να προετοιμαστούν. Δεν πάνε μόνο σε κράτη-μέλη, πάνε και σε τρίτες χώρες τους το ζητούν να πάνε, πήγαν στη Σερβία, Φερρυπίν, τέλος του έτους, πέρσι, διότι είχε μολυνθεί η Σερβία. Έχουμε και τους ελέγχους, ε, κάνουμε ελέγχους στην Ιρλανδία, οι αρμόδιοι, η ομάδα μας, για να τονοήσουν την κατάσταση και να κάνουν και ελέγχους να δουν κατά πόσο εφαρμόζουν τη στρατηγική και τις κατευθυντήριες γραμμές σε διάφορες χώρες. Μιλούσα για το το G7 δεν αφορά μόνο την Ευρωπαϊκή Ένωση, όλη την Ήπειρο της Ευρώπης. Από το 2014 μέχρι τώρα συναντηθήκαμε με όλους τους επικεφαλείς κτηνιατρικών υπηρεσιών όλων των χωρών της Ευρώπης που είχαν πληγεί από την ε, πανόλη των χείρων. Συζητήσαμε όλα τα σχετικά θέματα. Βέβαια, το πιο σημαντικό, τη διαχείριση των αγριοχείρων Πολύ χρήσιμες συναντήσεις και έτσι ανταλλάσσονται οι εμπειρίες που είχαμε γενικά. Έχουμε δύο φορές το χρόνο συνάντηση σε διπουργικό επίπεδο με τα κράτη-μέλη που έχουν πληγεί. Το 2015 ξεκινήσαμε και βλέπετε τη φωτογραφία και με του υπουργού Γεωργίας και τους Υπουργούς Περιβάλλοντος των κρατών μελών συναντηθήκαμε διότι η πανίδα είναι πολύ σημαντική στη διάδοση των όσων. Η τελευταία συνάντηση έγινε στη Σόφια. Σεπτέμβριο πέρσι. Και μία συνάντηση που θα αναφέρω τώρα. Οργανώσαμε στα περιθώρια της βόχια της Πράσινης Εβδομάδας την περασμένη εβδομάδα την Παρασκευή στο Βερολίνο μια διάσκεψη που ήταν πιο παγκόσμιο χαρακτήρα από ό,τι Ευρώπη. Είχαμε Κορέα, Ιαπωνία, είχαμε κι άλλους. Πάνω από 25 υπουργούς είχαμε εκεί, Υπουργοί Γεωργίας και ο Επίτροπός μου βεβαίως ήταν παρόν. Πολύ ψηλό επίπεδο διάσκεψη αυτή. Στόχος η ευαισθητοποίηση στα ύψιστα πολιτικά επίπεδα σχετικά με το κίνδυνο της αυθόδους ε, του, της πανόλης των χείρων. Είδατε ότι είχαμε πολύ υψηλό επίπεδο εκπροσώπηση, παγκόσμιοι φορείς επίσης ήταν παρόντες, διάφοροι οργανισμοί. Δυστυχώς ήταν πολύ μικρή αίθουσα. Έπρεπε να αρνηθούμε την είσοδο σε κάποιους που επιθυμούσαν να παραστούν. Είναι ύψιστη προτεραιότητα σε παγκόσμιο επίπεδο αυτή η ασθένεια. Είναι ένα πρόβλημα ασφαλείας τροφίμων. Επίτηδες το λέω, μιλάω για ασφάλεια τροφίμων. Ήταν και είναι και φέτος θέμα ασφαλείας τροφίμων στην Ασία 500 εκατομμύρια χείρους έχει η Κίνα μόνη της. Η μισή από αυτούς ε, πέθαναν λόγω της ασθένειας. Λίγα προσβληθέντα ζώα απομένουν ζωντανά. Τα γουρούνια που τρέχουνε, τρέχανε στα χωριά στην Κίνα δεν υπάρχουν πλέον. Πάμε σε μια αλλαγή παγκόσμιας εμβελίας όσον αφορά την κτηνοτροφία σε όλο τον κόσμο. Άρα, χρειάζεται σε παγκόσμιο επίπεδο δράση. Εκτός, εάν δεν υπάρξει εμβόλιο, θα είναι πολύ δύσκολο να εξαλειφθεί η ασθένεια σε παγκόσμιο επίπεδο. Η εξάλληψη είναι εφικτή σε μικρή έκταση. Το είδαμε αυτό στην Τσεχία και σύντομα και στο Βέλγιο θα το δούμε αυτό. όπου δεν υπάρχουν αγριόχειροι γίνεται να εξαλειφθεί. Όταν έχουμε τεράστιες εκτάσεις και δάση, δεν μπορείς να εξαλείψεις 100% την ασθένεια και τους αγριόχειρους. Θα παραμείνει ο ιός στις περιοχές αυτές. Ξοδέψαμε πολλούς πόρους ήδη να βοηθήσουμε τη διεξαγωγή έρευνας και να υπάρχει ανταλλαγή εμπειριών όχι μόνο ενδευρωπαϊκή, αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο, επανειλημμένα. Αναφερόμαστε ως ε, επικεφαλής ότι ηγούμεθα όσον αφορά την αντιμετώπιση της ασθένειας. Η ετοιμότητα είναι κάτι πολύ σημαντικό. Ανέφερα την Αμερικανική Ήπειρο. Ήταν παρόντες και εκπρόσωποι από τη Βόρεια και Νότια Αμερική. Το πιο σημαντικό είναι η αναγνώριση της περιφερειοποίησης. Να επιτρέπεται η συνέχιση του εμπορίου, εμπορίου με περιοχές που είναι ελεύθερες από την ασθένεια. Χρειάζεται επίσης διαφάνεια, εμπιστοσύνη, ανταλλαγή πληροφοριών. Είναι πολύ σημαντικά στοιχεία για αντιμετώπιση της πρόκλησης. Τα βλέπετε όλα αυτά στην ιστοσελίδα μας. Ακροθυγός, να σας δείξω μια διαφάνεια που χρησιμοποίησε ένας ομιλητής στη διάσκεψη την περασμένη εβδομάδα ποια θα είναι η μορφή της γεωργίας πολύ σύντομα στην Κίνα. Τεράστιες εκμεταλλεύσεις, εντελώς απομονωμένη κάθε εκμετάλλευση, δεν θα υπάρχουν άγρια ζώα γύρω. Ε, οι εργαζόμενοι που θα εισέρχονται θα απολυμένονται και θα μένουν εκεί μήνες όσο εργάζονται πριν να μπορέσουν να φύγουν. Και αυτό θα είναι ο μόνος τρόπος πιθανότατα να μπορεί να συνεχίσει η Κίνα να παράγει χείριο κρέας σε περιοχές όπου υπάρχουν ακόμα αυλ... αυλές μικροχώροι με προβλήματα όπου υπάρχουν τα ζώα και τι θα κάνουμε θα προσπαθήσουμε να εξακολουθήσουμε να υποστηρίζουμε τα κράτη-μέλη. Υπάρχουν πολλοί συνεργάτες μου που βοηθούν τα κράτη-μέλη να αντιμετωπίσουν την ασθένεια. Μοναδικός στόχος είναι να προσπαθήσουμε να ελέγξουμε την ασθένεια στο βαθμό του δυνατού, να είναι όσο πιο μακριά γίνεται από εκμεταλλεύσεις και να μην διαδοθεί, να μην μεταδοθεί πολύ γρήγορα. Και γι' αυτό πρέπει να πω ότι η συνεργασία πάει καλά. Αυτά λοιπόν για την Αφρικανική Πανόλη των Χείρων. Να θέλω και να παρουσιάσω και για την ε, γρήπη των πτηνών ε, κάποιες διαφάνειες, διότι η γρήπη των πτηνών ξανά ξεκινάει. Το ανέφερε κάποιος ευρωβουλευτής πριν από αυτό. Τώρα είμαστε στο H, στο H5N8. Από την 31η Δεκεμβρίου έχουν ε, μολυνθεί αρκετέ πόρε Πολωνία, Σλοβακία, Ουγγαρία, Τσεχία. Ε, η ασθένεια αυτή έχει πλήξει και την Τουρκία, τα μικρά οικόστα ζώα. Ε, δεν έχει πληγεί κάποια μεγάλη φάρμα, αλλά το h 58 H598 με ε, προέρχεται και πάλι από την Βόρεια Ασία σε συνδυασμό με διάφορους άλλους ε, ιούς που βρίσκονται στην Αρκτική. Αυτά όλα έλαβαν χώρα την προηγούμενη χρονιά ε, με επιρροή από κοπάδια από τη Ρωσία και από την Αφρική. Ε, κάποια ζώα τα μετέφεραν όλα αυτά προς νότο. Ίσως εδώ η διαφάνεια μην είναι και πολύ σαφής, αλλά βλέπετε τις ε, κίτρινες ε, κουκίδες, ε, Πολωνία, Τσεχία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Σλοβακία, όπου δυστυχώς ο, εντοπίστηκε αυτός ο ιός ε, και οδήγησε στη διαδικασία που αναφέραμε και προηγουμένως, δηλαδή ε, στην ε, θανάτωση των μολυσμένων ζώων, ε, στο να μπορεί με τον τρόπο αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει ελεύθερες εμπορικές ανταλλαγές. Όλα αυτά λοιπόν, όλα αυτά τα στοιχεία είναι στη διάθεση των βουλευτών και μπορείτε να δείτε μόνοι σας ε, τα μέτρα που λαμβάνουμε, ε, κάνουμε για την ε, νόσο των πτηνών, ό,τι κάναμε και κατά παρελθόν. Αλλά να πούμε και για άλλη μια φορά ότι αυτή δεν επηρεάζει την υγεία των ανθρώπων. Ζητώ συγγνώμη που μακρηγόρησα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την ε, ε, εντελεχέστατη παρουσίαση της Αφρικανικής Πανόλης των Χείρων. Ε, και τώρα θα τεθούν οι ερωτήσεις. Έχουμε ερωτήσεις που θέλουν να... Συναντέρφους που θέλουν να υποβάλουν ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλους... Η κυρία Σαντέρ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την εξονυχιστική αυτή παρουσίαση. Πληρέστατη ήδη απαντήσατε σε κάποιες απορίες μας. Εγώ θα ήθελα να καταθέσω μια μαρτυρία εδώ και να σας εκφράσω τη μεγάλη ανησυχία του αγροτικού κόσμου, κυρίως στη δική μου πατρίδα, στην Ανατολική Γαλλία, πολύ κοντά στα σύνορα δηλαδή με το Βέλγιο. ένα από τα βασικά ζητήματα που μας προβληματίζει, ένα από τα βασικά ερωτήματα είναι αν ε, ο φράχτης που κατασκευάστηκε και τα όρια που θέσαμε μεταξύ Βελγίου και Γαλλίας είναι αποτελεσματικά. Αν θα μπορέσουμε να αναχαιτήσουμε το πέρασμα της νόσου από το Βέλγιο στη Γαλλία. Γιατί υπάρχει ανησυχία των κτηνοτρόφων, των χειροτρόφων. Ήδη είχαν ένα σωρό στο κεφάλι τους. Έχουν μία ακόμη κρίση που πραγματικά ε, δεν τη χρειάζονταν. Γιατί αντιμετωπίζουν ήδη δυσκολίες και αυτό ήταν το κερασάκι στην τούρτα. Και ειδικά στη δική μου περιοχή, αλλά αυτό που λέω εγώ για την Ανατολική Γαλλία σίγουρα ισχύει και για τις άλλες περιοχές και περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουμε υπερπληθυσμό αγριοχείρων σε πολλές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ίσως α, αυτός ο συνοστισμός, αυτός ο υπερπληθυσμός των αγριοχείρων α, δημιουργεί πρόσφορα έδαφος για τη μετάδοση της νόσου. Δεν ξέρω αν μπορεί σε αυτό να επέμβει η Ευρωπαϊκή Ένωση και με ποιο τρόπο για να μειώσει τον πληθυσμό των αγριοχείρων. Ευχαριστούμε πολύ. Ο συνάδελφος κύριος ε, Μπούσμαν έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμο εκπρόσωπε της Επιτροπής. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά που μας είπατε σήμερα. Από το 2007 ε, έχει εξαπλωθεί η πανόλη των χείρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ιός ε, είναι ιδιαίτερα ανθεκτικός, επιβιώνει ακόμα και σε κατεψυγμένο κρέας και σε μεταποιημένα προϊόντα όπως είναι τα λουκάνικα. Ε, και αρκεί τα ζώα να ακουμπήσει το ένα το άλλο για να μεταδεθεί ο ιός. Δυστυχώς μέχρι τώρα δεν υπάρχει εμβόλιο. Ο λόγος για αυτή την ε, ε, ταχύτατη εξάπλωση της ασθένειας ε, στην Αφρική είναι ελψιγίνης και μεταφέρονται και τα ζώα σε μεγάλες αποστάσεις. Όλα αυτά υπάρχουν όμως και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό σας ερωτώ τι είδου μέτρα προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να περιορίσει την εξάπλωση του ιού, να θεραπεύσει τα ζώα, αλλά επουδενή όμως δεν πρέπει να ξεχνάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την προστασία των ζώων και το ίδιο προφανώς ισχύει και για την ε, γρήπη των πτηνών. Σάλφος Αντέμο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η Βουλγαρία είναι μία από τις χώρες εκείνες που επλήγει ιδιαίτερα από την Αφρικανική Πανόλη. Μέχρι σήμερα έχουμε θανατώσει 230.000 ζώα, που είναι το 15% του ζωικού κεφαλαίου στη Βουλγαρία. Τώρα, ε, συμπέρασμα. Χρειαζόμαστε κοινέ δράσεις ε, στην Ευρώπη. Ε, χρειαζόμαστε επίσης πανευρωπαϊκά μέτρα για να εμποδίσουμε την εξάπλωση αλλά και για πρόληψη. Και γι' αυτό ερωτώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Προσπαθείτε να βρείτε ενδεχομένω ε, κοινά μέτρα έτσι ώστε να υπάρχουν αυστηρότερες προδιαγραφές ε, ε, σχετικά με την ασφάλεια στις κτηνοτροφικές μονάδες και πιστεύετε ή προγραμματίζετε να υπάρχουν κάποια μέτρα για την επαναφορά του ζωικού κεφαλαίου στις πληγήσεις περιοχές. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε αξιότιμε κύριε εκπρόσωπε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Νομίζω ότι το θέμα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δυστυχώς είμαστε αναγκασμένοι να διαπιστώσουμε ότι το θέμα αυτό γίνεται όλο και πιο σημαντικό ανεξάρτητα από τις προϋποθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών μελών. Διαπιστώνουμε ότι το πρόβλημα αυτό έχει ήδη εμφανιστεί σε ε, τέσσερα κρατημέλη και εξαπλώνεται σιγά σιγά η χώρα μου, η Λιθουανία και οι γειτονικέ χώρες όπως η Λετωνία και η Εστονία. Ε, σχεδόν το σύνολο της επικράτειας αυτών των κρατών έχει πληγεί από αυτή την ασθένεια. Μιλάμε κυρίως για μικρές ε, μονάδες που έχουν μέχρι και 100 ε, χείρους ε, που αυτές οι εκμεταλλεύσεις, οι μονάδες ε, αναγκάζονται να κλείσουν, δεν μπορούν να επιβιώσουν. Άρα απομένουν μόνο οι μεγάλες εκτενοτροφικές μονάδες που είναι πάρα πολύ κακό. Εξαφανίζονται πολλές μικρές μονάδες και δεν υπάρχουν πολλές εναλλακτικέ λύσεις. Πριν από έξι χρόνια, 20.000 γουρουνάκια ε, αναγκάστηκαν, εξωθήθηκαν σε ενταφιασμό, τάφηκαν στο χώμα και τα μέτρα που ελήφθησαν δεν ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικά. Δυστυχώς ε, η επιδημία ε, εξαπλώθηκε εξαπλώθηκε περαιτέρω. Στη δική μου την περιοχή δεν κατέστη δυνατόν να εντοπιστούν τα αίτια της εξάπλωσης. Εξετάστηκαν ε, πάρα πολλές παραδοχές, αλλά δεν μπορέσαμε να καταλήξουμε κάπου. τώρα βέβαια σκεφτήκαμε να χρησιμοποιήσουμε και τους ε, ε, κυνηγού, αλλά οι κυνηγοί αρνούνται να σκοτώσουν ε, γουρουνάκια θηλυκά. Αν λοιπόν θέλουμε να λύσουμε το πρόβλημα, πρέπει να έχουμε πρότυπα που να ισχύουν παντού. Κοιτάξτε, δεν το βρίσκω σωστό να αγνοείτε τον πρόεδρο. Τέλο πάντων, μπα περιπτώσει. Κύριε Μάκεντάιρα. Κύριε Πρόεδρε, είναι η τελευταία φορά που μιλάω στην Επιτροπή και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για την υποστήριξή τους. Ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να λάβω το λόγο. Όσον αφορά την Αφρικανική Πανόλη των Χείρων, ανισχύει πάρα πολύ το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά ιδιαίτερα την περιοχή μου. Πρέπει να κατανοήσετε ότι από το πρίσμα του Ηνωμένου Βασιλείου εμείς πληγήκαμε ιδιαίτερα το 2001 από την ασθένεια του αυτόδους πυρετού που οδήγησε στη θανάτωση περίπου 6 εκατομμυρίων αγελάδων και προβάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ε, ξέρουμε πολύ καλά το τι μπορεί να μας συμβεί. Ε, έτσι λοιπόν μπορώ να σας μιλήσω για έναν Γεωργό ο οποίος ε, εκτρέφει ε, χείρους μιας ειδικής κατηγορίας ε, που είναι ακόμα πιο σπάνια από τα πάντα. Και αυτό το κάνει ε, στα, ε, έξω από το Forest of Dean, που εκεί αυτή η δασόδης περιοχή έχει άγρια ζώα που δεν ελέγχονται εύκολα. Αντί λοιπόν να τα συγκρατούν στην περιοχή εκεί τα άγρια ζώα, αυτά μπαίνουν στη μονάδα του παρότι έχει λάβει πολλά μέτρα ασφάλειας. Δεν ξέρω αν εσείς έχετε προσπαθήσει να κρατήσετε ε, μακριά από τα σπίτια σας, από τους ε, κήπους σας, ε, τους αγριόχειρους, γιατί αυτοί έρχονται, πηδάνε πάνω από φράχτες, τα κάνουν όλα ενωκάτω και φεύγουν. Και γι' αυτό αν τι ε, μολυστούν θα εξαφανίσουν όλα τα άλλα κοπάδια. Θέλω λοιπόν να σας υπογραμμίσω πόσο σημαντικό είναι αυτό το θέμα και να ερωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι σκοπεύει να κάνει για να περιορίσει τους αγριόχειρους. Ich glaube, ich kann für alle sprechen. Wir bedauern alle miteinander, dass das Ihr letzter Redebeitrag hier äh, in diesem Ausschuss äh, war und dass leider Ihr. Ε, πρόεδρος, ε, ήταν βέβαια μία από τις τελευταίες ε, παρεμβάσεις σας και λυπούμεθα πάρα πολύ που η χώρα σας θα μας αφήσει στις 31 Ιανουαρίου. Συνάδελφος Γιούργελ. Ευχαριστώ. Δύο θέματα. Το 2017 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύτηκε να βοηθήσει την Ουκρανία και τη Λευκορωσία να καταπολεμήσουν την Αφρικανική Πανόλη των Χείρων. Για τη Λευκορωσία μας μίλησε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Με την Ουκρανία τι γίνεται, υπάρχει συνεργασία με την Ουκρανία. Ε, μα, σε ενημερώνει για την κατάσταση απειλής που υφίσταται λόγω πιθανών κρουσμάτων. Ε, η Πολωνία έχει σύνορα με την ε, Λευκορωσία και την ε, Ουκρανία και είδαμε τις κουκίδες στην Πολωνία λόγω των επικίνδυνων καταστάσεων στα σύνορα. Τι γίνεται επίσης με τον εμβολιασμό. Υπάρχει διαθέσιμο εμβόλιο. Σε ό,τι αφορά τη γρήπη των πουλερικών, εμείς εξάγουμε ε, κάποιος είπε ότι εξήχθη πολωνικό μολυσμένο κρέας στην Ρουμανία. Σας διαβεβαιώ ότι στην Πολωνία έχουμε πολύ αυστηρούς ελέγχους για να περιορίσουμε την εξάπλωση ε, νόσων. Δεν μπορεί να έχει εξαχθεί μολυσμένο πολωνικό κρέας από την γρήπη των πουλερικών. Όπου βρέθηκαν μολυσμένα κρέατα έχουν καταστραφεί και έχουμε ε, θεσπίσει και ζώνες ασφαλείας γύρω από τις φάρμες που έχουν εντοπιστεί ε, τέτοιο μολυσμένο κρέα. Θα ήθελα λοιπόν ο συνάδελφο που δήλωσε ότι εισήχθη στη χώρα του μολυσμένο κρέα από την Πολωνία να ανακαλέσει γιατί αποκλείεται να έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, έχει κάποιο σύστημα για να καταπολεμήσει τον ιό H5N8 της γρήπης των πουλερικών. Τώρα, και τι χρηματοδότηση επίση θα προβλέψει για την καταπολέμηση τη γρήψης των πολεμικών. Σε ό,τι αφορά του αγριόχειρου, όντω η μεγαλύτερη απειλή για την Αφρικανική Πανόλη προέρχεται από αυτά τα ζώα. Ο κύριο Μπούντα, παρακαλώ, για να απαντήσει μάλλον σε μια ίσω προσωπική μόρφη. Ευχαριστώ. Έκανα μία παρατήρηση προηγουμένως ότι στην Ρουμανία υπάρχει μολυσμένο από την Πολωνία κρέας με τη γρήπη των πουλερικών, από τον ιό της γρήπης των πουλερικών. Είναι γεγονός, είναι σημαντικό να έχουμε υπόψη τι συμβαίνει στη χώρα μας ο καθένας. Ήδη από το 2015 λέγαμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κατασκευάσουν χάρτες, ε, φράχτες συγγνώμη, στα σύνορα με την Ουκρανία. Ε, τότε βέβαια δεν υπήρχε μεγάλο πρόβλημα και μας είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν χρειαζόμαστε φράχτες. Κι όμως σήμερα έχουν λάβει τέτοια έκταση τα φαινόμενα αυτά και τόσε πολλέ αιστείε παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση που αναγκαστήκαμε τελικά να κατασκευάσουμε και φράκτε για να περιορίσουμε την εξάπλωση τη ε, νόσου. Έχουμε υψηλά πρότυπα και προδιαγραφέ βιοασφάλεια για την κτηνοτροφία. Παρ' όλα αυτά όμω δεν μπορούμε να αναχαιτήσουμε την επέλαση του ιού. Θα πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε πολύ σοβαρά τα βήματα που θα πρέπει να γίνουν μετά τον εντοπισμό του ιού. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναπτύξει ικανότητες για να μπορούμε να αποτεφρώνουμε τα μολυσμένα σφάγια. Να μην τα ενταφιάζουμε, γιατί με τον ενταφιασμό δεν εξασφαλίζεται η εξόντωση του ιού και υπάρχει κίνδυνος ε, ε, να επανακάμψει η ασθένεια. Ο κύριος Χόισλινγκ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να μην σας αγνοήσω κύριε Πρόεδρε όταν μου επισημαίνετε ότι ε, πλησιάζω στο να εξαντλήσω το χρόνο μου. Ε, παρακολουθούμε την όσο αυτή περίπου μια δεκαετία και όσο περνάει ο χρόνος τόσο πιο κοντά στη Δύση έρχεται. Υπάρχουν κάποιες περιοχές στην Ευρώπη, όπως η Σαρδινία, όπου τέτοια πανόλη χείρων έχουμε εδώ και δεκαετίες. Θα πρέπει να ετοιμαστούμε για να συνδυώνουμε με αυτή την νόσο. Δεν μπορούμε να φτιάχνουμε φράχτες, να κατασκευάζουμε φράχτες παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλωστε η μόλυνση δεν γίνεται μόνο από αγριόχειρους, αλλά και από μολυσμένα τρόφιμα. Οπότε εκεί θα μας χρησιμεύσουν τίποτα οι φράχτες. Θα ήθελα να σας ρωτήσω για τα εμβόλια. Επενδύει καθόλου η Ευρωπαϊκή Ένωση σε εμβόλια για την Αφρικανική παρόλη των Χείρων. Νομίζω θα χρειαστεί αυτό στο μέλλον. Στην ε, Κίνα υπάρχουν ε, κάποιες μονάδες ε, που είναι σαν ένα πυρηνικά καταφύγια. Μα δεν μπορεί αυτό να είναι η λύση. Και γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει μακροπρόθεσμα να βρούμε κάποια λύση. Έχουμε δύο υπήρους που δεν έχουν μολυνθεί, αυτό είναι αλήθεια, αλλά και εμείς κάποια λύση πρέπει να βρούμε δεν νομίζω ότι είμαστε καλά εξοπλισμένοι για το μέλλον. Το μόνο που κάνουμε είναι να προσπαθούμε να γύρουμε φράχτες και αυτό δεν μπορεί να είναι η λύση. Ευχαριστούμε που ε, τηρήσατε το χρόνο σας. Ε, παρακαλώ, ε, Κισάνθος Κούτσμουκ. Σας ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την διεξοδικότατη παρουσίαση για την Αφρικανική Πανόλη των Χείρων και τη γρήπη των πουλερικών. Δυστυχώς στην Πολωνία έχουμε και τα δύο προβλήματα και γι' αυτό θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε δύο θέματα. Σε ό,τι αφορά την Αφρικανική Επανόλη των Χείρων, από το 2014 ασχολούμαστε με το θέμα και μέσα σε έξι χρόνια καταφέραμε να καταλήξουμε σε κάποια μέτρα που είναι απαραίτητα και τα οποία εφαρμόζουμε πάρα αυτά. Έχουμε διδαχθεί λοιπόν από το πάθημά μας. Σε ό,τι αφορά τώρα την οριοθέτηση των περιοχών που απειλούνται από την εξάπλωση και την προειδοποίηση, κοινοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη χαρακτήρι, το χαρακτηρισμό μιας περιοχής χωρίς αρρώστια, αυτό είναι πιο περίπλοκο θέμα. Πάντως, με τις πληροφορίες που έχετε από την Πολωνία, πώς γίνεται η υιοθέτηση των απειλωμένων περιοχών, γιατί νομίζω ότι υπάρχει μια μεγάλη βραδιπορία στην ε, διαδικασία αυτή. Και οι κτηνοτρόφοι ενδιαφέρονται το συντομότερο δυνατό να γίνει η οριοθέτηση για να ξέρουν ποιε περιοχέ είναι ασφαλεί. Αυτό για την Αφρική παρόλο το χείρο. Θα ενδιαφερθεί το ίδιο με του κτηνοτρόφου ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη γρήπη των πουλερικών. Είχαμε πέρυσι κάποια κρούσματα της γρήπης των πουλερικών στην Πολωνία, αλλά αφορούσε κυρίως μεγάλες κτηνοτροφικές μονάδες και εκεί ε, 175.000 ε, σμήνοι ε, πουλερικών θανατώθηκαν. Ερωτώ λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αποζημιώσει τους κτηνοτρόφους που υφίστανται τεράστιες ε, ζημίες λόγω της ανάγκης θανάτωσης σμηνών πουλερικών από την... που έχουν μολυνθεί από την κρήτη των πουλερικών. Η κυρία Μαγκίνες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την παρουσίαση και ευχαριστώ για το βαθμό λεπτομέρειας που περιέχει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλό θα ήταν να δραστηριοποιηθεί όχι μόνο εντό Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και παγκοσμίω. Αν δεν υπήρχε αυτή η κατάσταση επικοινωνίας, αν δεν υπήρχε αυτή η προσπάθεια οριοθέτηση και περιορισμού, φανταστείτε σε τι κατάσταση θα βρισκόμαστε σήμερα, γιατί φαίνεται υποτιμούμε την κατάσταση. Υπάρχει το θέμα της βιοσφάλειας που είναι απαραίτητο. Ο κύριος Χόισλινγκ είπε ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να μάθουμε να συνεπάρχουμε με τη νόσο αυτή. Επί, το θέμα είναι όταν η άγρια πανίδα βρίσκεται κοντά στα τα ζώα είναι εύκολη η μετάδοση τέτοιων νόσων. Επίσης, άλλο πρόβλημα για τη δημόσια υγεία είναι ο, κοροναϊός που εμφανίστηκε στην Κίνα. Ε, μπορεί να προέλθει από ε, τρόφιμα, από μολυσμένα τρόφιμα και σε τι πορεία βρίσκεται ανωδική ή καθοδική, πώς έχει η κατάσταση. κατασταση Ντονάτο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Έχω ερώτηση. Δύο ερωτήσεις για τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η πρώτη, για να έχουμε εξάλληψη του ιού, πρέπει να έχουμε μηδέν κρούσματα ανάμεσα στους χείρους, η θετικότητα, ή μηδέν κρούσματα στους αγριόχειρους. Το ρωτάω, διότι αντιπροσωπεύω, εκπροσωπεύω τη Σικελία και τη Σαρδινία και παρακολουθώ το πώς διαδίδεται η ασθένεια στη Σαρδινία. Δεύτερη ερώτηση. Ο μεγάλος αριθμός των αγριοχείρων προφανώς είναι ένα πρόβλημα, ένας κίνδυνος. Διότι αυξάνει το κίνδυνο διάδοσης της ασθένειας και είναι επιβλαβής για το περιβάλλον. Πρέπει να μειωθεί συνεπώς ο αριθμός των αγριοχείρων. Νομίζω ότι πρέπει να εξετάσει αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λαμβάνοντας δε υπόψη ότι υπάρχουν οι πράσινοι που θεωρούν το κυνήγι σαν επίθεση κατά του περιβάλλοντος. Νομίζω όμως ότι πρέπει να αλλάξει αυτή η προσέγγιση διότι η προστασία του περιβάλλοντος σημαίνει και προστασία άλλων ζώων και άλλων ειδών. Να προστατευτεί η βιοπικιλότητα από αυτού του είδους τον κίνδυνο. Ευχαριστώ. Η κυρία Καβαγιές έχει το λόγο. Thank you very much. Um, uh, Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας. Έχω μια ερώτηση από περιέργεια ορμόμενη την υποβάλλω. Ίσως να είναι εκτός θέματος. Είδα σε μία διαφάνεια την παρουσίασή σας τον τρομέα των ζωοτροφών. Διερωτώ με. Υπάρχει κάποιος αντίκτυπος για, τις, ε, για τη διατροφή για τα τρόφιμα μάλλον. Ξέρω ότι υπήρχε μεγάλο τρομερό, τρομερή επίδραση στα τρόφιμα στην Κίνα. Επειδή έγινε αυτή η μηνύα, παρουσιάστηκε αυτό στην παρουσίαση. Ευχαριστώ. Σμιτ Μπάου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά που είπατε. Μας ενισχύσαν πάρα πολύ. Ξέρετε, εμείς ε, στην Αυστρία ευτυχώς ακόμα δεν έχουμε πληγή από αυτή την ασθένεια. Όσον αφορά τη διαχείριση του κυνηγιού αγριόχειρου, πρέπει να το λύσουμε πανευρωπαϊκά, γιατί αυτό το κυνήγι είναι επικίνδυνο και δεν σταματάει σε κάποια εθνικά σύνορα. Κατά τα άλλα, επειδή αυτή η έκτακτη κατάσταση απαιτεί και έκτακτα μέτρα, εγώ θεωρώ ότι όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να δεσμευτούν και κατά την διαχρονική στιγμή να ξεκινήσουν ενημερωτικές εκστρατείες. Αυτά μπορούν να γίνουν, ε, δηλαδή ευαισθητοποίηση μέσα από εργαστήρια στη Ρουμανία, στη Γερμανία. Αυτό λειτουργήσε πάρα πολύ καλά και επίση και αυστηρότερη έλεγχη στα σύνορα και αυτό είναι απαραίτητο. Για να γίνει όμω κάτι τέτοιο πρέπει όλα τα κράτη να συμφωνήσουν ω εκ τούτου οι ταξιδιώτες, οι τουρίστες αλλά και οι κυνηγοί θα πρέπει ε, να είναι καλύτερα ενημερωμένοι έτσι ώστε να μπορούμε ε, να αποφεύγουμε καταστάσεις σαν αυτές που μας παρουσιάσετε στις ε, διαφάνειες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ο Πρόεδρος. Ολοκληρώθηκαν οι ερωτήσεις. Ε, και θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο και πάλι ε, στο συναδελφό μας ε, για να απαντήσει σε ερωτήσεις αυτές. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πολλές ερωτήσεις. Να ξεκινήσω από την τελευταία. Εκστρατεία ευαισθητοποίησης για τους ε, ταξιδιώτες και όλους που ασχολούνται με τον τομέα. Τα προγράμματα εξάλληψης που μπορούν να υποβληθούν από τα κράτη-μέλη, ακόμα και αν δεν έχουν τη ζωνόσο. Καλέσαμε και υποστηρίξαμε τα κράτη-μέλη, ούτως ώστε να παρουσιάσουν εκστρατείες ευαισθητοποίησης, τις οποίες θα χρηματοδοτήσουμε. Αν κάποιοι από εσά πάτε στη Γερμανία, θα δείτε στον αυτοκινητόδρομο στη Γερμανία, στους χώρους στάθμευσης, μεγάλε ανακοινώσει που λένε μην πετάτε το σάντουιτ σα, όχι μόνο γερμανιστή αλλά και σε άλλε γλώσσε. πολωνικά, ρωσικά, ουκρανικά όλα αυτά χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται αυτό σε πολλά κράτη-μέλη έχουν επενδυθεί χρήματα τα έχουν επενδύσει τα κράτη-μέλη και τους αποζημιώνουμε γι' αυτό, του τα επιστρέφουμε για να ευαισθητοποιήσουν τον κόσμο σε όλη την Ευρώπη το κάναμε Μιλήσαμε για την πρωτοβουλία GFTAD που την υποστηρίζουν οι αρμόδιοι φορείς και παραδείγματα στο, της ευαισθητοποίησης των εξτατιών ε, ευαισθητοποίησης βλέπετε στην ιστοσελίδα GFTAD ε, σε όλη την Ευρώπη, όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα δείτε τέτοια παραδείγματα. Μπορούν τα κράτη-μέλη να πάρουν παραδείγματα πώς γίνονται αλλού εκστρατείες ευαισθητοποίησης. Και επιμένω και σας το λέω ότι εμείς χρηματοδοτούμε μέχρι 100% αυτές τις εκστρατείες ευαισθητοποίησης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ξέρω ότι υποτίθεται όλοι γνωρίζουν τον νόμο, αλλά για το συγκεκριμένο ζήτημα όπου ο καθής μπορεί να μεταδώσει την ασθένεια μέσω σάντουιτς από μολυσμένο ζώο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αυτό που συνέβη στην Πολωνία, στα δυτικά της χώρας, στην τσεχική δημοκρατία, στο Βέλγιο, θα μπορούσε να συμβεί σε οποιαδήποτε άλλο μέρος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου μολυσμένο κρέας, ίσως παράνομα, αγοραστεί από ταξιδιώτες, οδηγούς φορτηγών, από οποιονδήποτε. και μπορεί να πετάξουν το σάντουιτς και να προσελκύσει κάποιο αγριόχειρο. Χρειάζεται ευαισθητοποίηση. Το ίδιο προσπάθειες γίνονται και σε αεροδρόμια ευαισθητοποίησης μετά την ε, ε, επιδημία την, του αυθόδου πυρετού που ανέφερε η συνάδελφος από την Ηνωμένο Βασίλειο. Όταν ε, υποτίθεται ότι όταν μπαίνει στην, στην Ευρωπαϊκή Ένωση βλέπεις μεγάλες οθόνες, αφήσει που καλούν τους ταξιδιώτες να μην φέρνουν γάλα, κρέας ε, ή ζαμπών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με τον νέο κανονισμό για επισήμους ελέγχους που, θα, που ετέθη σε ισχύ τον περασμένο χρόνο, τέλος του χρόνου, κάνουμε το ίδιο και για τα φυτά, για να προστατεύσουμε την υγεία των φυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρω ότι δεν εφάρμοσαν τα μέτρα ακόμα όλα τα κράτη-μέλη. Από 14 Δεκεμβρίου θα έπρεπε όμως να έχουν αυτές τις αφήσει και να κάνουν εκστρατείες ευαισθητοποίησης ε, να προστατευτούν από την ξυλέλα και άλλες ε, ασθένειες στα φυτά. Τι μπορώ να πω για τους φράκτες. Αυτή είναι μια πρώτη αντίδραση μιας χώρας. Ας υψώσουμε φράκτες γύρω μας για να προστατευτούμε. Η ΕΦΣΑ υπήρξε σαφέστατη. Οι φράκτες δεν βοηθούν. Οι φράκτες που έχουν μεγάλη, μεγάλο μήκος δεν θα εμποδίσουν τα αγριαζώνα να μετακινηθούν από τη μία άκρη του φράκτη στην άλλη. Γι' αυτό ποτέ δεν υποστηρίξαμε φράκτες μεγάλων αποστάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την προστασία της πανίδας ε, του ενός κάτω μέλους από άλλο κάτω μέλος. Για μικρές αποστάσεις οι φράκτες λειτουργούν. Το είδαμε στη Τσεχική Δημοκρατία. Τους δώσαμε αυτή τη συμβουλή. Το έκανα στο Βέλγιο. Θα θυμόσαστε ένα μικρό κομμάτι στο Νότιο Βέλγιο, Γαλλία, σε συγκεκριμένη περιοχή ύψος εφράκτες έχει αποτελέσματα σε μικρή κλιμάκα το μέτρο αυτό. Οι φράκτες που κατασκευάζονται, κατασκευάστηκαν από τη Γαλλία σε πλήρη συντονισμό με τις βελγικές αρχές ε, στηρίχθηκαν και από τους εμπειρογνώμονές μας που ήταν επιτόπου. Θέλαμε να μειώσουμε τον πληθυσμό των αγρίων ε, χείρων από μικρή περιφέρεια. Για μια ασθένεια χρειάζεσαι τον φορέα και τον ιό. Αν δεν έχεις το φορέα δεν έχεις την ασθένεια. Δεν έχεις την ασθένεια... Αν δεν έχεις φορέα δεν έχεις την ασθένεια. Εάν μειώσει τον πληθυσμό, εξαλείψει τον πληθυσμό σε μικρή κλίμακα, σε μικρή περιοχή, αυτό είναι κάτι που δίνει αποτελέσματα και αυτό συνέστησαν στην Πολωνία και στη Γερμανία οι εμπειρογνώμονες μας και υπάρχουν επαφές μεταξύ Πολωνίας και Γερμανίας σε πολύ ψηλό πολιτικό επίπεδο για να εξασφαλιστεί ότι τα πάντα θα γίνουν ούτω ώστε να αποφευθεί μετάδοση τη ασθένεια. Σε μεγάλη κλίμακα όμω στην πράξη δεν δίνει αποτελέσματα ο φράκτης και το ίδιο μας είπε Οι κυνηγοί παίζουν μεγάλο ρόλο κάνουν τα πάντα για να αποφύγουν τη διάδοση των ασθενείων, ένα Σαββατοκύριακο μπορεί αυτοί πάνε κοινοί για να καταστρέψουν έξι μήνε δραστηριοτήτων. να μην κάνουμε προσπάθειε για να απομονώσουμε τα ζώα. Είναι σαφέστατο αυτό. Επανειλημμένα αναφέρθηκε. Όταν εμφανιστεί σε ένα δάσο η ασθένεια. Στην Πολωνία, στο Βέλγιο, στη Τσεχική Δημοκρατία. Οι πρώτες οι ιδέες που λένε κάποιοι είναι πάμε να σκοτώσουμε τους αγριόχειρους εκεί, να σπυροβολήσουμε. Αυτό είναι το αντίθετο από αυτό που πρέπει να κάνεις. Ακριβώς το αντίθετο. Όταν βρεις ότι υπάρχει ασθένεια σε κάποιο δάσος, πρέπει να αφήσει τον πληθυσμό των αγριοχείρων. Μιλάει για του αγριοχείρου. Όταν λέω για πληθυσμό, δεν μιλάει για ανθρώπινο πληθυσμό, για του αγριόχειρου. Μιλάω για τον πληθυσμό των αγριόχειρων. Του αφήνει στην ησυχία του μέχρι να ξέρει σε ποιο βαθμό έχει μεταδοθεί ασθένεια. Και καμιά φορά είναι πολύ δύσκολο να το εξηγήσει κανείς αυτό. Και υπήρξαν κάποιοι υπουργοί πληγέντων κρατών μελών που εξέφρασαν τις απόψεις, αλλά είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί αυτό. Η κυνηγή, ο κυνηγός θέλει να μπει στο δάσος και να κυνηγήσει. Και το μόνο που κάνει ο κυνηγός κυνηγώντα είναι να μεταδίδει την ασθένεια πολύ μακριά το πρώτο που πρέπει να κάνεις είναι να αφήσει το δάσος στην ησυχία του, χωρίς παρέμβαση. Μέχρι να ξέρεις ακριβώς πού έχει πάει ο ιός και μετά υψώνεις φράκτες και μετά μειώνεις ε, τον πληθυσμό ή προσπαθείς να εξαλείψεις τον πληθυσμό. Όπως είπα και στην παρέμβασή μου, ο ιός είναι πολύ αποτελεσματικότερος από, από τους κυνηγούς. Εάν Βάζει φράχτη γύρω από την περιοχή, 100% του πληθυσμού θα πεθάνει μέσα. Και μετά τι κάνει, μαζεύει μετά τα νεκρά ζώα. Γιατί για έξι μήνε είναι δραστήριο ο ιός εντό του πτώματο. Εάν βρει ένα νεκρό ζώο που είναι τεσσάρων ή πέντε μηνών νεκρό, όπω έγινε και στο Βέλγιο την περασμένη εβδομάδα, ακόμα μπορεί να βρει στο νεκρό σώμα τον ιό. Δεν λέω ότι είναι δραστήριο, ενεργό, αλλά υπάρχει στο πτώμα. Βασικό θέμα λοιπόν, όταν βρεις έναν ιό στο δάσος, είναι να τον κρατήσεις, να μείνεις έξω, μην μπει μέσα. Προσπάθησε να δεις σε ποιο βαθμό έχει μεταδοθεί ασθένεια. Μετά υψώνεις φράκτες και κάνεις αυτό που κάνεις στη Τσεχία, επιτυχέστατα. Η πρώτη χώρα που κατάφερε να εκριζώσει, να εξαλείψει αυτό τον ιό στην Ήπειρο ήταν αυτή, όπως και το Βέλγιο ελπίζουμε. Θα μπορέσουμε σύντομα να ανακοινώσουμε ότι είναι ελεύθερο από την ασθένεια το Βέλγιο και ελπίζουμε ότι και οι Πολωνοί μαζί με τους Γερμανούς θα το πετύχουν και αυτοί. Τώρα για τους κυνηγούς. Κυνηγοί, κυνηγοί. Είναι το κλειδί. Έχουν, έχουμε επαφή με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Κυνηγών και το Διεθνή Σύλλογο, τη Διεθνή Οργάνωση Κυνηγών και οι δύο ήταν παρόντες στην Πράσινη Εβδομάδα του Βερολίνου. Επίσης συμμετείχαν στη διάσκεψη που οργανώσαμε στα τέλη του 2019 με Υπουργούς Γεωργίας και Περιβάλλοντος. Προσπαθήσαμε εκεί να εξηγήσουμε το ρόλο που παίζουν οι κυνηγοί στην προσπάθεια εξάλληψης ε, της νόσου. Ό,τι αφορά τον κοροναϊό, τον ανθρώπινο κοροναϊό που μεταδίδεται από την Κίνα, η Παγκόσμια Οργάνωση της Υγείας θα συνεδριάσει, η συνεδρία σήμερα το πρωί θα συνεδριάσει το απόγευμα και σήμερα το απόγευμα θα συνεδριάσει και η Επιτροπή Ασφάλειας της Υγείας των 28 χωρών μελών για να δούμε τι μέτρα θα προταθούν σε συνεργασία με τον ΩΣΑ για να αποφευθεί περαιτέρω εξάπλωση της γρίπης του κοροναϊού. Η Σαρδινία είναι ειδική περίπτωση. Δεν έχει σχέση με τις επιζώτιες που βλέπουμε στην υπόλοιπη Ευρώπη. Η Σαρδινία έχει ένα ιδιαίτερο τρόπο εξάπλωσης, οπότε δεν θα συνέκρινα την κατάσταση της Σαρδινίας με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντως είμαστε απόλυτα διαφανείς. Ό,τι κάνουμε είναι καθαρό και εξάστερο και μπορείτε να το βρείτε στη ιστοσελίδα μας ανα πάσα στιγμή. Σας ευχαριστούμε για την πληρέστατη και αρτιότητα παρουσίαση που μας κάνετε. Μία πολύ σύντομη ερώτηση του κυρίου Μπούντα. Έχω μία ερώτηση κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από του πολλού συναδέλφους γιατί το μολυσμένο κρέας στη Ρουμανία δεν προερχόταν από την Πολωνία αλλά από την Ουγγαρία. Ζητώ συγγνώμη λοιπόν, ανακαλώ. Μάλιστα, σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υπομονή του και τις πολύ αναλυτικές απαντήσεις που έδωσε. Φυσικά θα συνεχίσουμε να προβληματιζόμαστε γιατί το θέμα της Αφρικανικής πανόλε των Χείρων δεν πρόκειται να καταλήψει το φοβάμαι, το χάρτη της Ευρώπης. Τώρα, 28 με 30 Νοεμβρίου, επίσκεψη της ε, αντιπροσωπείας της Επιτροπής Άγκρη στη Γαλλία. Επικεφαλής της αντιπροσωπείας μας ήταν ο κύριος Ντόρφμαν και οργανωτές η κυρία Σαντέρ και ο κύριος Δεσδέ. Σας ευχαριστούμε θερμά για την διοργάνωση αυτής της αποστολής. Μιλήσαμε για πολλά θέματα. Γάλα, κρασί, ε, Βόιο κρέας, ε, πρόβιο κρέας, αλλά θα μας τα πει αυτά πιο αναλυτικά ο επικεφαλής αντιπροσωπείας, ο κύριος Ντόρφμαν. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τρεις ημέρες κράτησε η αποστολή της αντιπροσωπείας μας και ενημερωθήκαμε για διάφορους κλάδους της Ευρωπαϊκής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας. Ξεκινήσαμε την αποστολή στη Λιόν και την ολοκληρώσαμε στο Στρασβούργο. Καλύψαμε δηλαδή μία διόλου καταφρόνητη απόσταση. Η προεργασία και η προετοιμασία της, ακρο... της επίσκεψης αυτής ήταν εξαιρετική και ο κύριος Ρίντεγκερ και η ε, συνάδελφος Αν Σαντέρ έκαναν μια αρτιότατη προετοιμασία και γι' αυτό ήταν και πολύ επιτυχημένη η αποστολή μας. Επισκεφτήκαμε τα κέντρα αριστείας της ε, γαλλικής ε, γεωργίας και κτηνοτροφίας. Είδαμε πώς παράγεται το κρέας ρολέ, πήγαμε στην Βουργουνδία, ε, είδαμε την παραγωγή κρασιού, πήγαμε στο Κοντέ για το τύρι, στην Αλσατία. Περισσότεροι το γνωρίζουμε γιατί όλοι πηγαίνουμε στο Στρασβούργο. και είδαμε διάφορες μορφές οργάνωσης και των παραγωγών. Στην περιοχή Φρανς Κοντέ συναντήσαμε πραγματικά μία τέλεια οργάνωση της αλυσίδας παραγωγής. Χάρη σε αυτή την άρτια οργάνωση, η προστιθέμενη αξία των προϊόντων είναι πολύ μεγάλη. Συναντήσαμε εκπροσώπους οργανώσεων παραγωγών, αλλά και μεμονωμένους παραγωγούς. Συζητήσαμε με τους αμπελαργούς το θέμα της επιβολής δασμών ε, από τις Ηνωμένε Πολιτείες. Μιλήσαμε για το Βόλιο Κρέας και τη Συμφωνία Μερκοσούρ και πώς θα επηρεάσει το εμπόριο βοήου κρέατος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ούτω καθεξής. Τίποτα άλλο, απλώ ευχαριστήσω του συναδέλφου που συμμετείχαν και στην προετοιμασία που έγινε από τη Γραμματεία και του δύο οργανώτε. Νομίζω ότι είχαμε πολύ ενδιαφέρουσες ε, συζητήσεις ε, και νομίζω ότι όλα αυτά μπορούμε να τα εκμεταλλευτούμε στις εργασίες που θα διεξάγουμε εδώ στην Επιτροπή μας. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Ντόρφμαν για την έκθεση αυτή. Ευχαριστούμε πολύ όλου του ε, μετέχοντες. Ε, δεν ξέρω, επιθυμεί κανείς ε, να λάβει το λόγο, να πει κάτι, από ό,τι βλέπω όχι. Ως εκ τούτου το κλείνουμε αυτό το θέμα της ημερήσιας διάταξης και πάμε στο σημείο υπαρθμών 13, μεταβατικές διατάξεις για τη στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγύσεων. Όπως ξέρετε αυτή είναι η δεύτερη σημαντικότερη έκθεση όπου προσπαθούμε να πετύχουμε πρόοδο. Θα ήθελα λοιπόν να δώσω το λόγο στη συνάδελφό μας, ε, την κυρία Κατάινεν, για 8 λεπτά. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δίνετε να εργαστώ πάνω σε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο ε, θα είναι πραγματικότητα για τους Ευρωπαίους Γυργούς σε λιγότερο από 49 εβδομάδες. Εμείς ε, που είμαστε νομοθέτες είναι πολύ σημαντικό να προσφέρουμε ε, σταθερότητα στους γεωργούς και στο γεωργικό τομέα και να διασφαλίσουμε ένα σαφό σαφή δρόμο προς τη μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής. Η γεωργή ε, αυτούς αφορά ο κανονισμός, ε, σε αυτούς θα γίνουν αισθητέ οι προεκτάσεις. Ε, Αυτά τα βιώνουν ήδη και πριν εκπονηθεί, πριν θεσπιστεί ο κανονισμός. Εγώ που είμαι και η ίδια Γεωργός γνωρίζω πολύ καλά ε, περί τίνος ακριβώς ε, πρόκειται. Είναι σαφές ότι ε, θα πρέπει να συνεχίσουμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Όσον αφορά την Επιτροπή μας, εγώ θέλω να υπογραμμίσω ότι χρειαζόμαστε μία ταχεία διαδικασία λήψης αποφάσεων. Οι γεωργοί πρέπει να γνωρίζουν έγκαιρα το τι τελικά θα συμβεί. Και γι' αυτό το λόγο ο δικός μου στόχος είναι να ψηφιστεί μέχρι τα τέλη Απριλίου, να αρχίσει να δουλεύει αποτελεσματικά κατά τη διάρκεια της ε, Προεδρίας της Κροατίας, να υπάρξουν οι τριμερείς ε, διάλογοι, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι αυτό που χρειαζόμαστε κυρίως είναι να υπάρξει συμφωνία για το πολιετές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους και συζητητές για την συνεργασία που είχαμε σε αυτό το θέμα. Αγαπητοί συνάδελφοι, ο στόχος του σχεδίου έκθεσης του δικού μου είναι να συμπεριλάβω όσο δυνατόν ε, περισσότερες από τις ε, προτάσεις σας. Και γι' αυτό αυτή η ανταλλαγή απόψεων είναι πολύ σημαντική. Όσον αφορά το περιεχόμενο του σχεδίου της ε, έκθεσης και τις δικές μου απόψεις ως εισηγήτριας, πιστεύω ότι οι πρώτες κομισιόν να συνεχίσουμε με νέα χρήματα και με όλα τα εργαλεία, αυτό είναι πολύ καλό. Βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω οι πρώτες κομισιόν. Είναι εξάλλου σαφές ότι δεν μπορούν να ισχύουν οι παλιοί κανόνες με λιγότερα χρήματα εγώ πιστεύω ότι πρέπει την κοινή γεωργική πολιτική να την εξετάσουμε στο πρίσμα του ότι στηρίζουμε ε, τον τρέχοντα προεπλογισμό. Δεν μπορούμε να δεχτούμε μείωση των ε, κονδυλίων για την κοινή γεωργική πολιτική. Εγώ ως εισηγήτρια ε, θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει μία ε, μεταβατική εξέταση του θέματος, ξεχωριστά από την κοινή γεωρική πολιτική. Στην κοινή γεωρική πολιτική υπάρχει ένα παράθυρο ανοιχτό για μεγαλύτερες αλλαγές, ε, παραδείγματος χάρη ε, λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα που θα ληφθούν ε, στο πλαίσιο της ε, Πράσινης Συμφωνίας. Δεν μπορούμε να έχουμε δύο παράλληλες διαδικασίες μεταρρυθμίσεων. Το υπογραμμίζω αυτό. Αυτό είναι πάρα πολύ για τους γεωργούς. Και αυτό είναι και το βασικό μήνυμα που εξέπεμψαν σχεδόν όλοι οι άμεσα εμπλεκόμενοι του τομέα με τους οποίους συναντηθήκαμε πριν από δύο εβδομάδες. Ένα από τα βασικά θέματα της ε, έκθεσης είναι η διάρκεια η Επιτροπή προτείνει ένα χρόνο και αυτό ε, δεν μοιάζει πολύ ρεαλιστικό. Κατά τη δική μου άποψη, ε, δεν μπορού... τον ένα χρόνο μεταβατική περίοδο μπορούμε να τον φτάσουμε μόνο κάτω από ορισμένε προποθέσει. Η συμφωνία για το Πουδουπού και οι προσωρινέ ε, συμφωνίε για την ε, μεταρρύθμιση της ΚΑΠ θα έχουν ολοκληρωθεί πριν από το τέλος Ιουνίου 2020. Ε, τα κράτη-μέλη χρειάζονται 12 μήνες για την στρατηγική προετοιμασία και η Κομισιόν χρειάζεται 6 μήνες για έγκριση. Πρέπει λοιπόν να στηρίξουμε, να δείξουμε εμπιστοσύνη στους διαπραγματευτές μας της ΚΑΠ να διασφαλίσουμε ότι η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ ε, θα γίνει αποτελεσματικά. Να εμπιστευτούμε επίσης και τους διαπραγματευτές για το που που όπου ε, η συμφωνία θα πρέπει να επιτευχθεί την άνοιξη. Είναι σημαντικό όχι μόνο για τη Γεωργία, αλλά για το, ε, γενικότερα για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχοντας αυτά κατά νου, είναι σαφές ότι θα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί στο να να επεκταθεί ενδεχομένως η μεταβατική περίοδος σε τέσσερα έτη. Και με ενδιαφέρει δική σας άποψη επί της διάρκειας. Με συγχωρείτε, η μεταβατική περίοδος να είναι δύο έτη και όχι τέσσερα. Ε, θα ήθελα επίσης να εξετάσουμε τα προγράμματα της γεωργικής ανάπτυξης κυρίως ε, το πώς εγκρίνονται τα αιτήματα των κρατών μελών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης, να εξετάσουμε λειτουργικά προγράμματα και για πόσο χρονικό διάστημα ε, μπορούν να τρέξουν αυτά. Θα ήθελα με χαρά να ακούσω τις απόψεις σας επ' αυτού. Είναι επίσης ε, σημαντικό στο δεύτερο πυλώνα τα κράτη-μέλη να έχουν τη δυνατότητα αυξημένου ποσοστό συγχρηματοδότησης με βάση το επίπεδο που υπάρχει αυτή τη στιγμή ε, στον Πουδουπού και επίσης ε, να μπορούν να λάβουν και νέα περιβαλλοντικά μέτρα στα προγράμματά τους γιατί είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη και νέες προκλήσεις. Κατά την άποψή μου θα πρέπει να ακολουθήσουμε αυτή τη λογική ε, του να συνεχιστούν όλα αυτά τα μέτρα, μεταβατική, μεταβατικές ε, ενισχύσεις. Σε γενικές γραμμές η σημαντικότερη αρχή είναι να διασφαλίσουμε την ε, ε, υποστήριξη προς τους γεωργούς χωρίς καμία διακοπή και προς άλλους βέβαια αποδέκτες κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περίοδου. Μπορούμε να προετοιμάσουμε το έδαφος και για την νέα κοινή γεωργική πολιτική, αυξάνοντας την τεχνική αρρωγή και βοηθώντας τα κράτη-μέλη να προετοιμάσουν προσεκτικά τα στρατηγικά προγράμματα. Με τον τρόπο αυτό θα φτιάξουμε μια γέφυρα ανάμεσα στην μετάβαση και την μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη συνάδελφο κυρία Κατάινεν και θα πρότεινα πρώτα να ακούσουμε τους σκιώδεις εισηγητές με την σειρά που ακολουθούμε πάντα. Συνάδελφος Αμάρο, θα έλεγα για 1,5 λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να τονίσω την ανάγκη συνεργασίας ε, με την εισηγήτρια την κυρία Κατάινεν. Ήδη είχαμε μια αρκετά παρατεταμένη συνεδρίαση με πολύ θετικό πνεύμα και θεωρώ ότι η κυρία Κατάινεν επικεντρώθηκε στα ουσιώδη. Και συμφωνώ με αυτό. Εγώ θα ήθελα να σταθώ την εξάρτηση που υπάρχει μεταξύ του ΠΔΠ και της ΚΑΠ. Φυσικά η μεταρρυθμίση της ΚΑΠ θα εξαρτηθεί από το ΠΔΠ, αλλά αυτό θα πρέπει να μας δίνει κίνητρο και ανάβσματα να επιταχύνουμε τις διαπραγματεύσεις για το πολίτες δημοσιονομικό πλαίσιο. Επουδενή όμως δεν θα πρέπει ε, αυτή η επίσπευση των διαπραγματεύσεων για το ΠΔΠ να βλάψει τους γεωργούς ή να οδηγήσει καθυστερήσεις στην καταβολή των άμεσων ενισχύσεων. Γιατί έχουμε ΚΑΠ που ισχύει. Μέχρι ότου αναθεωρηθεί η κοινή πολιτική θα πρέπει να εφαρμόσετε η τρέχουσα δεν θα πρέπει να έχω μια και καλυμμένη αναθεώρηση μέσω μιας χρηματοοικονομικής μεταρρύθμισης που τελικά θα βλάψει τους γεωργούς και κτηνοτρόφους. Σε ό,τι αφορά το χρονικό ορίζοντα, η πρόταση για το μεταβατικό κανονισμό θα έχει διάρκεια ένα έτος, αλλά θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για παράταση μέχρι δύο έτη. Ξεκινάμε με την αρχική διάρκεια του ενός έτους, αλλά θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για παράταση για δύο έτη, προκειμένου να εξασφαλιστεί απρόσκοπτη καταβολή των ενισχύσεων στους Γιώργους. Η κυρία Γιλέρα, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την κυρία Κατάινεν, γιατί είναι πολύ πρόθυμη και συνεργάσιμη και αυτό φάνηκε, γιατί από την πρώτη στιγμή ε, ανάμειξε και έναπλεξε και τους και οδησηγητές στην όλη διαδικασία και την ευχαριστούμε γι' αυτό. Είμαστε φυσικά όλοι θερμοί υπέρμαχοι της διαφύλαξης του κανονισμού της κοινή γεωργικής πολιτικής και φυσικά θέλουμε και μεταβατικό κανονισμό. Και η πρόταση περικοπής ε, των γεωργικών κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, θα μας βρει απέναντι. Εμείς θα υποστηρίξουμε την διασφάλιση του τρέχοντος προϋπολογισμού της ΚΑΠ. Επίσης θεωρώ ότι μεταβατική περίοδος ενός έτους δεν είναι ρεαλιστική. Αν ε, ολοκληρωθούν όλες ε, οι διαπραγματεύσεις, ε, μπορεί να μπει αμέσω σε ισχύ ο κανονισμός. Οπότε δεν έχει περισσότερη αξία το επιχείρημα του ενός έτους από τα δύο και διετή είναι η παράταση. Από τη στιγμή που θα είναι έτοιμος ο κανονισμός και θα ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις, αμέσως μπορούμε να περάσουμε στη νέα κατάσταση. Σε ό,τι αφορά τα απορροκυπευτικά τώρα, Ήδη από το Σεπτέμβριο του 2021 ζητούμε νέα πρόταση αναθεώρησης των λειτουργικών προγραμμάτων. Γιατί όμως, ε, ενώ για την μελισσοκομεία, για τα μπελονικά έχουμε διαφορετικές διατάξεις, για τα προκυπευτικά θέλετε ε, άμεση αναθεώρηση. Επίσης, έχουμε 118 ε, PDR και οι δικαιούχοι είναι πολλές περιφέρειες. Δεν θα τροποποιήσουμε τον στρατηγικό μας σχεδιασμό από την 1η Πρώτου του 2021. Το PDR θα πρέπει να το ολοκληρώσει ε, η περιφέρεια, ακόμη και στη συνέχεια το σύστημα αλλάξει. Ευχαριστώ κύριο Σροπέ. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να συμφωνήσω με τους ε, συναδέλφους. Ε, θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τη συνάδελφο κυρία Κατάινεν. Είναι λυπηρό το γεγονός ότι χρειαζόμαστε αυτό τον κανονισμό και εγώ πράγματι πιστεύω ότι το ένα έτος είναι πολύ λίγο. Επίσης, ε, πιστεύω ότι πρέπει να απορρίψουμε τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα δικά μας, τα στοιχεία δική μας οι αριθμοί είναι πολύ καλοί και επικυρώθηκαν και κατά την προηγούμενη θητεία. Κατά τα άλλα, έχω και επιφυλάξεις ε, ε, όσον αφορά σε κάποιες ε, τροπολογίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, παραδείγματο χάνει τη μετάβαση στην βιολογική γεωργία, αναφέρονται τα τρία έτη και αυτά περιορίστηκαν σε ένα έτος. Αυτό όμως δεν είναι ρεαλιστικό. Πέρα από αυτό έχουμε και προγράμματα για τα κρατη που σημαίνει όμως ότι ορισμένα προγράμματα δεν θα μπορούν να εφαρμοστούν ε, και τα κρατη θα κληθούν να επιστρέψουν χρήματα. Αυτό είναι μειονέκτημα, ε, πρέπει να το έχουμε κατά νου. Κατά τα άλλα, θα ήθελα να μιλήσω για την εξωτερική σύγκληση η οποία πρέπει να διασφαλιστεί, αλλά αυτό δεν το προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όμως πρέπει να το διεκδικήσουμε. Ε, διεκδικήσουμε επίσης ε, και τη βιωσιμότητα. Άκουσα πολύ προσεκτικά την κυρία Κατάινεν και η κυρία Κατάινεν είπε πραγματικά τα σημαντικότερα. Θα ήθελα να υπογραμμίσω κάτι το οποίο ελέγχθη καθαρά διαδικαστικά από πλευράς χρόνου δεν είναι ρεαλιστικό η μεταβατική περίοδος να είναι ενό έτου. Θα πρέπει ευθύ εξ αρχή να μιλήσουμε για δύο έτη. Ευχαριστούμε πολύ. Συνάλφος κυρία Αγγιλάρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την εισηγήτρια, την κυρία Κατάινερ. Σας διαβεβαιώ ότι ε, βρισκόμαστε σχεδόν απολύτως στην ίδια γραμμή πλεύσης. Ε, μικρές ε, δευτερεύουσε ε, τροπολογίε θα προτείνω, όπω για τα προκυπευτικά που σχολίασε ήδη η κυρία Αγγιλέρα. Πέραν τούτου, θεωρούμε ότι ο σεβασμό τη αρχή τη συνέχεια και αποφυγή μια μεταρρύθμιση τη μεταρρύθμιση είναι υπέρ και των γεωργών και των κρατών μελών που θα κληθούν να διαχειριστούν την κοινή γεωργική πολιτική. Και αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστέ, όπω ζήτησαν και οι προλαλήσαντε, ο μεταβατικό κανονισμό μα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον διετή ώστε να εξασφαλιστεί επιπλέον σταθερότητα για τους γεωργούς μας. Επίσης, ο μεταβατικός κανονισμός δεν μπορεί να περιλαμβάνει τις δημοσιονομικές ε, προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά θα πρέπει να περιλαμβάνει τις, γραμ... τις προτάσεις του τρέχοντος ΠΔΠ ή τις προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μακάρι να υιοθετηθεί το συντομότερο δυνατό ο κανονισμός, αλλά έχουμε απόλυτη εξάρτηση από την πιθανή συμφωνία για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Επαναλαμβάνω, ε, βρισκόμαστε σε απόλυτη σύμπνοια με την εισηγήτρια την κυρία Κατάινεν. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία, λέει ο πρόεδρο. Οι διερμηνεί και πάλι μα παρακαλούν να μιλάτε ή δυνατόν λίγο πιο αργά. Ο κύριο Κόκαλη, παρακαλώ. Να, ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου την κυρία Κατάινεν και το Στάφτη για την συνεργασία που είχαμε. Ε, Συμφωνούμε και εμείς ότι είναι δύσκολο σε ένα χρόνο να συμβούν όλα αυτά. Είναι όμως ε, χρήσιμος αυτός ο χρόνος δεδομένης της ε, πράσινης συμφωνίας που πρέπει να ε, εντάξουμε στην καινούργια ΚΑΠ και σε αυτόν και είναι καλό όπως στην Πράσινη Συμφωνία έχουμε ε, φιλοδοξίες, υψηλές φιλοδοξίες. Ας δοκιμάσουμε να το κάνουμε σε ένα χρόνο και αν το καταφέρουμε, εδώ είμαστε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία και συνεχίζουμε Ähm, και εμεί ε, σα ευχαριστούμε. Ε, έχουν ζητήσει και άλλοι το λόγο ε, προηγουμένως είχαν ζητήσει πάρα πολύ το λόγο, ίσως να ξέχασα κάποιον, να διαβάσει τον κατάλογο και να πούνε κάποιοι αν δεν ακούσουν το όνομά του. Αντριέ, κολέγη Κουτσμουκ, Χιτβεγγι, Τομάσικ, Alieva Veli, Ademov, Buda, De Castro, Jürgil und der Kollege Le Breton. Gibt es noch weitere Kollege äh, Lavacek? Ja. Lavacek. Gut, dann ähm, der, die Kollegin äh, Tolleré. Συνάδελφος Τολερέ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ την κυρία Κατάινεν και όλη την ομάδα της για την πολύ καλή συνεργασία. Ήταν χαρά μας και το βλέπουμε και σε αυτό που είπαν οι διάφοροι που έχουν ασχοληθεί με το θέμα αυτό και πήραν το λόγο. Υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες τεχνικής φύσης όσον αφορά την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κυρίως κάποια βεβαιότητα σχετικά με το πώς, ε, τελικά θα υπάρχει κάλυψη των προθεσμιών. Η πρόταση δεν επιτρέπει να παρατείνουμε μέχρι πέντε χρόνια το πρόγραμμα σύγκριση για τη βιολογική ε, γεωργία. Όμω αυτό το πρόγραμμα μετατροπή προ τη βιολογική καλλιέργεια, τα προγράμματα χρειάζονται μια προθεσμία πενταετία. Υπάρχουν και χώρε όπω είναι η Γαλλία που ήδη έχουν δεσμευτεί ε, να δώσουν οικονομική υποστήριξη για πέντε χρόνια για τέτοια προγράμματα που καλύπτουν τι δύο θητείε. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν και την επόμενη περίοδο πέρα από το 2021 πόρου για να εγγυηθούμε αυτές τις, να τηρηθούν αυτέ οι δεσμεύσει που ε, συνάδουν με την Πράσινη Συμφωνία για τις νέες δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν το 2021 μέγιστη διάρκεια των για τα πρημοδοτήσεις στην ανάπτυξη πέθρου είναι κάτι πολύ περιοριστικό όσον αφορά τα αγροπεριβαλλοντικά και τα βιολογικά προγράμματα και προβράζει διοικητικής για ένα κάτω μέλος να χειριστεί προγράμματα τριετή και πενταετή ταυτόχρονα είναι περίπλοκο Απόλυτα συμφωνώ με του συναδέλφου, δηλαδή ότι τα οπορικεπιστικά δεν υπάρχει πρόβλημα, να, δεν πρέπει να αντιμετωπιστούν διαφορετικά από όλου τομεί. Όσον αφορά τον Ίνο, θα πρέπει να συνεχιστούν τα μέτρα τα ατομιακά μέχρι την εκπνοή που προβλέπεται από την αρχή, από την αρχικά προβλεπόμενη περίοδο εκπνοής των μέτρων. Ευχαριστώ, καμπάγέ. Συνάδελφα Καμπαγέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θέλω πάνω απ' όλα να υπογραμμίσω ότι ο μεταβατικός κανονισμός είναι πολύ σημαντικός για να υπάρξει συνέχιση, συνέχεια για την υποστήριξη των γεωργών και να έχουμε προβλησιμότητα και ασφάλεια που είναι θεμελιώδη για την δραστηριότητά τους. Αλλά πιστεύω εξίσου ότι η οθέτηση μεταβατικής περίοδου δύο χρόνια πιο μεγάλη θα εγγυόταν καλύτερη σταθερότητα, σταθερότητα και συνέχεια. Το επαναλαμβάνω ότι αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλες τις πτυχές δυνατότητα να ολοκληρωθούν τα επιχειρησιακά προγράμματα για τα προκυπευτικά και δεν νομίζω ότι από αυτή την πρόταση έχουμε τέτοιο αποτέλεσμα. Δεύτερον, επανειλημμένα σε αυτή την Επιτροπή και σωστά αναφέρθηκε ότι εν γέννη στην ΚΑΠ υπάρχουν προτάσεις περικοπών μιλάω για το πρόγραμμα POSEIT για τις υπερπεριφερειακές περιοχές, τις απόμακρες περιοχές. Το Νοέμβριο το συζητήσαμε. Η περικοπή των οικονομικών πόρων για το πρόγραμμα POSEIT, αν και έχει σημαντική αξία για τους γενικούς λογαριασμούς, όμως θεωρούμε ότι είναι σημαντικό πρόγραμμα για μειονεκτούσες γεωγραφικέ περιοχέ και που έχουν δομικά προβλήματα και ιδιαιτερότητε που υπενθυμίζω ότι αναγνωρίζονται από τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ευχαριστώ, συνάδελφε Αντρία, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Εν συντομία, να επιμείνω, όπως έκαναν και διάφοροι συνάδελφοι, για τη διάρκεια της διετίας. Σήμερα χρειαζόμαστε μεγαλύτερη σαφήνη όσον αφορά το δημοσιονομικό πλαίσιο, το πολιτές. Θα πρέπει να, να, να διευκρινίσει τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπή ε, όσον αφορά την Πράσινη Συμφωνία, τι θα κάνουμε στο αγροτικό τομέα είναι σημαντικό να υπάρχει μεταβατική περίοδος, θα επέμενε επί δύο σημείων. Πρέπει να το υπενθυμίσουμε. Πρώτα απ' η παράταση των πολιτών μέτρων του δευτέρου πυλώνα. Πιστεύω ότι είναι απαραίτητο να τροποποιηθεί το ποσό υποστήριξη τη Ένωση για την περίοδο που παρατείνεται πέρα το 2020. Και δεύτερον, πιστεύω ότι είναι σημαντικό και το λέω σαν υποστηριχτή στο θέματο να υπάρχει ευθυγραμμισμό των τομιακών υποστηρίξεων σχετικών προγραμμάτων που θα πρέπει να ενταχθούν στα μελλοντικά στρατηγικά σχέδια. Είναι πτυχέ πρώτου-δεύτερου πυλώνα που είναι σημαντικά στοιχεία πρέπει να ληφθούν για την όλη ε, μετάβαση. Ευχαριστώ, συνάδελφε Κουτσμιούκ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ την κυρία Κατάινεν για την ε, παρουσίαση των μεταβατικών διατάξεων. Εγώ είμαι αναφαδόν υπέρ της διετούς διάρκειας του μεταβατικού κανονισμού. Νομίζω ότι θα πρέπει οι διατάξει αυτές να ισχύουν για μία διετία. Επίσης, απαραίτητη είναι και η διαφύλαξη της ευελιξίας. Η δυνατότητα δηλαδή μεταφοράς των κονδυλίων από τον πρώτο στο δεύτερο πυλώνα. Το ισχύον ποσοστό είναι 25%. Τουλάχιστον το ισχύον ποσοστό να διαφυλαχθεί. Επίσης, οι μεταβατικές διατάξεις θα πρέπει να προβλέπουν τη δυνατότητα ε, μεταβατικής ε, και κρατικής υποστήριξης με τις χείουσες διατάξεις ε, του άρθρου 37 του κανονισμού 1308. Σε ό,τι αφορά τη συνέχεια των ενισχύσεων, επίσης ε, για τη μεταβατική περίοδο θα πρέπει να ισχύσουν αυστηρότεροι κανόνες από τους ε, υφιστάμενους. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ντόρφμαν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συμφωνώ με αυτά που είπε η συγκητριά μας, η κυρία Κατάινεν. Ε, πράγματι πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε το ταμείο αυτό να μην παραμείνει διακοσμητικό ε, γιατί ε, αλλιώς ε, θα εμπλακούμε σε μια πολιτική συζήτηση που πρώτον θα διαρκέσει περισσότερο και δεύτερον θα επικαλύπτεται με την τρέχουσα συζήτηση που έχουμε για τις ε, τρεις εκθέσεις μας σχετικά με την κοινή πολιτική. Όσον αφορά το χρονικό διάστημα, γνωρίζω πολύ καλά ότι υφιστάμεθα όλο και περισσότερο χρονική πίεση, αλλά αν πούμε ευθύ εξ αρχής δύο χρόνια για τη μεταβατική περίοδο, τότε αυτό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 θα σημαίνει ότι τα κράτη-μέλη θα ολιγορήσουν, δεν θα κατασκευάσουν τα εθνικά στρατηγικά του προγράμματα, γιατί θα πιστεύουν ότι έχουν χρόνο. Όσον αφορά το μεταβατικό έτος, δεν είναι ένα κανονικό έτος. Δεν μπορούν να ξεκινήσουν πενταετή σε περίοδο, δεν μπορούν να ξεκινήσει το πρόγραμμα Leader. Αυτά ήταν και το 2014. Γι' αυτό λοιπόν, όσο πιο ε, σύντομοι είμαστε στο χρόνο, τόσο καλύτερα. Ένα χρόνο να πούμε, ε, το είπαν και κάποιοι άλλοι, και μετά από τον ένα χρόνο, αν δούμε ότι δεν φτάνει, κάνει, εντάξει, τότε μπορούμε να προσθέσουμε άλλο ένα χρόνο. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, ο μεταβατικός κανονισμός δεν σημαίνει παράταση των υφισταμένων κανόνων της ΚΑΠ. Ε, και σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ε, εισαγωγή νέων κανόνων. Οπότε ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλό θα ήταν να ακολουθήσει τη λογική του 2014, της προηγούμενης μεταρρύθμισης. Γιατί στην περίπτωση αυτή δεν ξεκινούμε από τις εθνικές ενισχύσεις όπως το παρελθόν. Αυτό δεν μας βρίσκει σύμφωνο. Δεν μπορούμε από τη μια στιγμή στην άλλη να διακόψουμε κάποιες μορφές ενισχύσεων. Αυτές οι κρατικές ενισχύσεις στηρίζουν ευαίσθητους τομείς. Αν τις καταργήσουμε, θα πλήξουμε πολύ σοβαρά τους Γιώργους. Οπότε, αν δεν συμπεριληφθεί η δυνατότητα κρατικών ενισχύσεων, δεν θα μπορέσουμε να υπερψηφίσουμε την πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ, κύριε Στομα... η κυρία Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Είναι πολύ σπουδαίο και περίπλοκο θέμα γιατί είναι θέμα που άπτεται πολλών διαφορετικών διατάξεων. Ε, δεν μπορούμε να δεχτούμε την πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπής για μονοετή παράταση. Μέσα σε ένα χρόνο δεν μπορούν τα κράτη-μέλη να ετοιμάσουν τα εθνικά στρατηγικά του σχέδια. Χρειάζεται παράταση της περίοδου και για τους φορείς πληρωμής για να προετοιμαστούν για την εφαρμογή των νέων νομοθετικών διατάξεων. Η μεταβατική λοιπόν διάρκεια θα πρέπει να είναι διετής, να καλύπτει και το 2021 και το 2022. Στο άρθρο 1 δεν σύμφωνα με την πρόταση ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να παρατείνουν την περίοδο, μόνο όμως όταν διαπιστώσουν ε, κίνδυνο ανεπάρκειας ε, χρηματοοικονομικών κονδυλίων και άρα μη τήρηση των υποχρεώσεων θα πρέπει να είναι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τα κράτη-μέλη, αλλά να μην ξεχνά και την επικορικότητα. Επίσης, το άρθρο 8, παράγραφος 6, το ποσό προτείνεται ουσιαστικά προεξοφλεί την έκβαση των διαπραγματεύσεων για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Εννοείται ότι θα καταθέσω τροπολογίες για το μεταβατικό κανονισμό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σόιντροβα.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 την εθνική υποστήριξη κατά τη μεταβατική περίοδο. Νομίζω ότι αυτό αναφέρθηκε από αρκετούς συγητές και αν ισχύει αυτό που είπε η συγητρία, ότι θα πρέπει να ισχύουν για τη μεταβατική περίοδο οι παλαιοί κανόνες, τότε αυτό σημαίνει ότι αυτά που ισχύουν τώρα θα πρέπει να ισχύουν και κατά το μέλλον. Αν αυξηθεί η μεταβατική περίοδος, τότε προτείνω να προβλεφθεί ε, μεγαλύτερη ευελιξία. Τώρα, όσον αφορά τη διάρκεια, νομίζω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τους γεωργούς που χρειάζονται τη σταθερότητα και οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν κατά πόσον αρκεί το ένα έτος. Αλλά αυτό το θέμα νομίζω ότι πρέπει να είναι πραγματικά προτεραιότητά μας. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, την κυρία Κατάινεν, ε, για την ε, πολύ καλή οργάνωση της εργασίας, πάρα πολύ καλή δουλειά. Και επίσης ε, να υπογραμμίσω ότι πρόκειται για μία συζήτηση που αφορά νομοθετικές προτάσεις. Ε, η συγκήτρια προσπάθησε να απευθυνθεί σε όλους τους άμεσα εμπλεκόμενους. Βεβαίως ε, και θέλει να προσφέρει σταθερότητα ε, το να έχουμε νέους κανόνες. Αυτό θα συμβάλλει στη σταθερότητα και εγώ συμφωνώ με όλους τους συναδέλφους οι οποίοι χρειάζονται εθνικές μεταβατικές διατάξεις για μας αυτές είναι πολύ σημαντικές, κυρίως για τους γεωργούς που θίγονται περισσότερο, κυρίως δηλαδή για τους μικρούς γεωργούς και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτές οι εθνικές ενισχύσεις ε, δεν πρέπει να έχουν καμία επιρροή στον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αναλύσεις έχουν ε, καταδείξει ότι αυτές οι ενισχύσεις δεν πρέπει να επηρεάζουν τα συμφέροντα άλλων γεωργών, να μην στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό αυτές οι μεταβατικές ενισχύσεις να συνεχίσουν να ε, χορηγούνται με τον ίδιο τρόπο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, την κυρία Κατάινεν. Ε, της ε, εύχομαι καλή επιτυχία στην έκθεσή της και να συμφωνήσω με τους συναδέλφους εκείνους που ανησυχούν για το ότι η μεταβατική περίοδος δεν εμπίπτει στις διατάξεις που υπάρχουν για μεταβατικές ε, περιόδους. Η μεταβατική περίοδος είναι πολύ σημαντική για χώρες όπως είναι η Βουλγαρία. Αυτή η μεταβατική περίοδος προβλέπει ενισχύσεις που θα ε, βοηθούσουν, θα βοηθήσουν και βοηθούν αυτούς που έχουν τη γη περισσότερο. Αν καταργηθούν θα έχουμε πτωχεύσεις, εγκατάλειψη της γεωργίας, ε, εγκατάλειψη της υπαίθρου, αναζήτηση άλλων μορφών μορφών απασχόλησης. Κύριε Πρόεδρε, ελπίζω να συμφωνήσετε με αυτά τα επιχειρήματά μου. Συνάδελφος Μπούντα, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ σύντομα, θέλω να αναφερθώ στη μεταβατική εθνική ενίσχυση. Είναι σημαντικό να παραμείνει μια δυνατότητα στα χέρια των κατών μελών. Φαίνεται ότι υπάρχει μια αντίφαση προ τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από τη μία πλευρά ζητά περισσότερα χρήματα από τα κάτι μέλη να μπουν για τη γεωργία στο κονδύλι της Ευρωπαϊκής, στον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω και από την άλλη μεριά περιορίζουμε τα κράτη-μέλη να δώσουν χρήματα στους ε, γεωργούς τους και να ικανοποιηθούν περισσότερο οι γεωργοί στον αγροτικό τομέα. Θα πρέπει να είναι σαφέστατο το μήνυμα. Δεν μιλάμε εδώ για ευρωπαϊκούς πόρους, μιλάμε για εθνικούς πόρους δεν εξαρτάται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρέμβει σχετικά με αυτά που γίνονται στο κράτο μέλο και τι κάνει το κράτο μέλο με τα λεφτά του. Δεν έχει σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξαρτάται από τι εθνικέ κυβερνήσει. Ευχαριστώ, συνάδελφε Ντίκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ γρήγορα. Συγχαρητήρια στην συνάδελφο Κατάινεν. Καταλαβαίνω απόλυτα αυτά που μα είπε στην παρέμβασή τη και χάρηκα που είδα ότι συνεργάστηκαν ισχυώδει άριστα σαν ομάδα. Λοιπόν, κοιτάξτε, το πρόβλημα δεν υπάρχει, συνάδελφοι. Αν καταφέραμε ποτέ να εγκρίνουμε τις τρεις νομοθετικές ε, πράξεις ε, πιο σύντομα, αυτομάτως θα τεθεί σε ισχύ. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνω γιατί έχουμε τέτοια ανησυχία και τέτοιο άγχος. Να βάλουμε ήσυχα τα δύο χρόνια από ό,τι κατάλαβα τα υποστηρίζουν περισσότερε ομάδε και θεωρούν την αναγκαία. Μετά από αυτό, αν είμαστε τόσο θαραλέοι και καλοί να εγκρίνουμε τι νομοθετικέ πράξει και να κάνουμε στιμερεί διαλόγου και να δώσουμε το χρόνο στα κράτη-μέλη για να γίνει αυτή η μετάβαση, ε, θα, θα μπουν σε ισχύ. Αυτό ήθελα να πω. Ευχαριστώ. Συνάδελφε. Κύριος Γιούργκελ. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, σίγουρα η νέα περίοδος προγραμματισμού είναι πολύ περίπλοκη γιατί θα έχουμε τα νέα στρατηγικά σχέδια και γι' αυτό θα συμφωνήσω με τους συναδέλφους που ζήτησαν μεταβατική περίοδο διετή και όχι μόνο ετή όπως προτείνει ο μεταβατικός κανονισμός. Επίσης, οι μεταβατικές διατάξεις θα πρέπει να προβλέπουν τη δυνατότητα ε, εφαρμογής ε, και των κρατικών ε, ενισχύσεων με βάση το άρθρο 37 του κανονισμού 1308 του 2013 ε, θα πρέπει να προβλέπεται και αυτή η δυνατότητα των κρατών μελών για τις κρατικές ενισχύσεις. Οι μεταβατικές διατάξεις ε, για το χαρακτηρισμό, την επιλεξιμότητα των ε, δαπανών με βάση άρθρο, το άρθρο 6 είναι πολύ περιοριστική. Η Πολωνία θεωρεί ότι οι μεταβατικές διατάξεις για την παρέμβαση στον τομέα των απορροκυπευτικών θα πρέπει να προβλέπει και τη δυνατότητα συνέχιση με βάση τους παλιούς κανόνες των λειτουργικών προγραμμάτων, και των οργανώσεων παραγωγών με βάση τον κανονισμό 1308 του 2013. Επίσης, ε, αυτό το είδαμε και στην προηγούμενη μεταρρύθμιση που όταν δεν συνοδεύεται με κατάλληλες μεταβατικές διατάξεις ε, ε, δημιουργεί προβλήματα στην συνέχιση των λειτουργικών προγραμμάτων και δημιουργεί αβεβαιότητα στις οργανώσεις παραγωγών για το ποιοι κανόνες θα πρέπει να ισχύσουν για τη συνέχιση των προγραμμάτων Του Ευχαριστώ. Ο κύριο Λεμπρετόν. Ευχαριστώ. Πάρα πολύ σημαντικό που ασχολούμαστε με αυτό το θέμα του μεταβατικού του κανονισμού. Είναι το πιο κατεπήγον πρόβλημα που θα πρέπει να διευθετηθεί προ όφελο των γεωργών μα. Δεν μπορώ παρά να επαναλάβω τα υποθέντα, διότι ευτυχώ υπάρχει κάποια συνένεση που διαμορφώνεται. Εγώ θα επέμενα επί τριών σημείων. Τρει αρχέ. Η πρώτη αρχή είναι η οικονομική σταθερότητα θα πρέπει να διατηρηθούν οι παρόντες κανόνες κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περίοδου. Δεύτερη αρχή, σημαντική ισοτιμίας. Τα απορροκεπευτικά θα πρέπει να αντιμετωπιστούν όπως τα άλλα προϊόντα. Και τρίτη αρχή, η αρχή λογική ευλόγου χρονικού διαστήματο. Ένα έτο δεν είναι κάτι ρεαλιστικό. Θα έπρεπε να προβλέπουμε από τώρα ένα χρόνο παραπάνω και να ανακοινώσουμε ε, να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους για να ξέρουν τι να περιμένουν ε, οι γεωργοί μας. Είναι ένα θέμα και ασφαλείας δικαίου. Να έχουν μια ασφάλεια, αν Ασφάλεια. Ευχαριστώ, συνάδελφε Λάβατσεκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον συνάδελφό μου Κατάινεν για τη δουλειά που έκανε με την ομάδα της. Η συζήτηση κατέδειξε σαφώς ότι λίγο πολύ έχουμε τέσσερις τομείς ε, προς διευκρίνηση. Ε, και νομίζω ότι αν το κάνουν αυτό θα διασκεδάσουν τι ανησυχίε μας και θα προχωρήσουμε αρκετά γρήγορα. Πρώτα απ' όλα, προβλεψιμότητα του προπολογισμού που σχετίζεται με το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Πρώτο, δεύτερο στοιχείο, συσχετίζεται με τη μεταβατική περίοδο και βλέπω μία τάση για πάνω από ένα χρόνο μεταβατική περίοδο, αλλά σημαντικότερο θα ήθελα να τονίσω ότι χρειαζόμαστε σαφήνεια για τη μετάβαση, όχι μόνο όσον αφορά τα μέτρα και του τομεί που καλύπτει, αλλά και τις δεσμεύσει στο δεύτερο πυλώνα και κυρίως το σημείο που ανεφέρθηκε επανειλημμένα σχετικά με την προβλεψιμότητα, με το καθεστώ το μεταβατικό των κρατικών ενισχύσεων. Και στην προηγούμενη μεταρρύθμιση τα είχαμε πάει καλά και θα έπρεπε να εμπνευστούμε από αυτό. Οι παρόντες κανόνες ε, για την κρατική ενίσχυση ε, εκπνέουν φέτος. Ευχαριστώ. Η κυρία Σάντορ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ την ομάδα της συγγήτριας και τους κοιόδης εισηγητές. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι το Κοινοβούλιο ήδη οθέτησε επανειλημμένα θέση όσον αφορά το δημοσιονομικό πλαίσιο και εντός αυτού ζητούμε τα απόθεμα για τις κρίσεις, για την έκτακτη ανάγκη να μεταρρυθμιστεί και ε, να ε, έχει ένα βασικό κεφάλαιο από την αρχή του προπολογισμού, 400 εκατομμύρια ευρώ, που θα προέρχεται από φρέσκα χρήματα που θα δίνονται επιπλέον του προπολογισμού της ΚΑΠ. Το προηγούμενο κοινοβούλιο φρόντισε να μεταφράσει αυτή τη θέση στον οριζόντιο κανονισμό, να συμπεριληφθεί. Αλλά ήθελα να ρωτήσω τη νομική υπηρεσία και τη γραμματεία αν μπορούν να διευκρινίσουν κατά πόσο για νομική και πολιτική συνοχή να συμπερι... αυτή τη θέση στον κανονισμό των μεταβατικό. Ε, σας ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Ε, ολοκληρώθηκαν λοιπόν οι ερωτήσεις. Ε, θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που σε τρία λεπτά παρακαλώ καλύτερα να τοποθετηθεί. Ευχαριστώ Πρόεδρε να ευχαριστήσω και την εισηγήτρια για την έκθεση που ετοίμασε πολύ γρήγορα. Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε επικοδομητικά αφού διαβάσουμε μεγάλο ενδιαφέρον την έκθεση και να επιλύσουμε τεχνικά προβλήματα που τη διαβάσουμε. Σε ένα τρίλεπτο θα περιοριστώ αναφερόμενος σε βασικά σημεία πολιτικής ε, σημασίας στο πολιτικο δημοσιονομικό πλαίσιο και τα χρήματα. Καταρχάς, όπως γνωρίζετε, όταν κάναμε την πρόταση, είχαμε μόνο ένα σημείο αναφορά για τα χρήματα, την πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Αυτό βλέπετε. Αλλά νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνετε ότι από τη στιγμή που θα έχουμε το νέο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο, θα έχει συμφωνηθεί ότι αυτή η πρόταση θα πρέπει να προσαρμοστεί δεόντω για να αντικαταστήσει τα στοιχεία που υπάρχουν τώρα στην πρόταση προ τα στοιχεία που θα συμπεριλαμβάνονται στο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Και τούτου λεχθέντο πρέπει να πούμε ότι βασιζόμεθα στο ενδεχόμενο ότι πράγματι το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο θα υφίσταται, θα συμφωνηθεί σε πολιτικό επίπεδο μέχρι ότου ο κανονισμό να εθετηθεί επίσημα. Είναι ένα εγχείρημα τεχνική φύσεω, αλλά θα πρέπει να είμαστε ε, συνεννοημένοι πάνω σε αυτό. Ε, δεύτερο σημείο, η περίοδο. Ε, σας καλώ ας ασχοληθούμε αυτό το θέμα στο τέλο τη διαδικασία, όταν θα έχουμε μεγαλύτερη σαφήνεια όσον αφορά την πιθανή διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα της μεγάλης μεταρρύθμισης της ΚΑΠ και μετά θα δούμε κατά πόσο είναι πραγματιστικό και εφικτό όπως προτείναμε εμείς σαν Κομισιό να παραμείνει ένα έτος υπάρχει μεγάλη ανάγκη χωρίς να, ε, ε, να επηρεάσουμε τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ να έχουμε μεγαλύτερη μεταβατική περίοδο τώρα για τις δεσμεύσεις για τα αγροτροφημικά και τα διάφορα μέσα στο δεύτερο πυλώνα, να σας υπενθυμίσω για μία ακόμη φορά το λόγο για τον οποίο κινηθήκαμε τούτο τρόπος. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να βάλουμε στο απόθεμα όσο περισσότερο, περισσότερα χρήματα από το νέο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο για τα νέα ε, προγράμματα της ΚΑΠ, γιατί εκεί θα πετύχουμε στόχους όσον αφορά το περιβάλλον και το κλίμα, να μην δεσμευτούν τόσα πολλά χρήματα με του παλιού κανόνε, να δεσμευτούν με, τα, με του καινούριου κανόνε. Γι' αυτό μειώσαμε την περίοδο, αλλά αυτό είναι μόνο για τις νέες αναλήψεις ε, υποχρεώσεων που θα αναλάβουν έναντι των δικαιούχων τα κράτη-μέλη το 2021 για τη μεταβατική κρατική ενίσχυση. Εκεί η θέση μας ήταν ότι δεν συμπεριελήφθη αυτό το θέμα, διότι το προτείναμε στα πλαίσια της μεταρρυθμίσεως. Αυτή η μεταβατική εθνική ενίσχυση θα έλεγε υποτίθεται το 2020 και γι' αυτό κάναμε στην πρότασή μας Πρέπει να καταλάβουμε βέβαια ότι υπάρχει και ένα θέμα συνέπεια ε, με του κανονισμού περιμεταρρύθμιση και αν το Κοινοβούλιο αποφασίσει τελικά να μην παρατείνει τη την εθνική μεταβατική ενίσχυση στα πλαίσια μεταρρύθμιση στο ΚΑΠ, θα ήταν λογικό να μην κάνουμε κάτι τέτοιο σε αυτή την πρόταση. Και αντιστρόφω βεβαίω ισχύει αυτό. Κάτι τελικό, τεχνική φύσεω, αλλά σημαντικότατο. Κάποιοι από εσά αναφερθήκατε στι κρατικέ ενισχύσει και ότι πράγματι υπάρχει ένα καθεστώ σχετικό για τι κρατικέ ενισχύσει. Ισχύει τώρα, υπήρχε μια ομαδική εξαίρεση στι κατευθυντήριε γραμμέ που καθόριζε από ποιου όρου τα κράτη-μέλη μπορούν να διαθέσουν εθνικού πόρου για του γεωργού και άλλου δικαιούχου και αυτό το πλαίσιο κρατική ενισχύσεω θα εκπνεύσει το 2020. Τελεία. 31 Δεκεμβρίου και ήδη προσπαθούμε να παραταθεί μέχρι το 2021 για να μπορέσουμε να συντονιστούμε και με την περίοδο που προβλέπεται για το μεταβατικό κανονισμό. Σταματάω εδώ και ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση θα λάβει το λόγο η συνάδελφος κυρία Κατάινεν που θα ήθελα να την παρακαλέσω να συνοψίσει σε 2-3 λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ όλους σας. Ήταν έξοχες οι προτάσεις σας. Αυτά που είπατε θα βοηθήσουν την ομάδα μας στο έργο της. Πράγματος χάρη τα θέματα των απορροκυπευτικών του Ίνου, το η Συμφωνία και τα προγράμματα που τρέχουν παράλληλα και διάφορα άλλα θέματα. Η χρονική πίεση είναι πολύ μεγάλη και είναι σαφές ότι χρειαζόμαστε συμπληρωματικό χρόνο προς τα χρόνο για τις εθνικές διοικήσεις και τους γεωργούς να προετοιμαστούν όλοι για τη μεταβατική περίοδο. Αυτό είναι ένας λόγος παραπάνω να προχωρήσουμε πιο γρήγορα στη λήψη αποφάσεων. Μην διστάξετε όμως να έρθετε σε επαφή μαζί μου ή με την ομάδα μου για οποιοδήποτε θέμα. Η παρουσίαση του σχεδίου εκθέσεως θα λάβει χώρα στις 17 ή 18 Φεβρουαρίου και η προθεσμία υποβολή τροπολογιών θα είναι 25 Φεβρουαρίου και όπως προανέφερα στόχος είναι να ψηφιστεί από την Επιτροπή Γεωργίας τέλος Απριλίου και να ξεκινήσουμε εργασίες το ταχύτερο δυνατόν με την Κροατική Προεδρία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τη συνάδελφο κυρία Κατάινεν και τους σκιώδης για την μέχρι τώρα δουλειά τους και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Περνάμε τώρα στο σημείο υπεριθμών 14 της ημερήσιας διάταξης. Είναι το τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξης για τη σημερινή ημέρα. Πρόκειται για την ε, Ευρωπαϊκή ε, Στρατηγική Δασοπονίας, Στρατηγική Δασών. Ε, αποφασίσαμε να καταρτήσουμε, να συντάξουμε μία έκθεση πρωτοβουλίας. Αυτό θα το κάνουμε από κοινού με την Επιτροπή Περιβάλλοντος στο πλαίσιο του κανόνα 57. Η συγητή είναι ο συνάδελφος Σάρβαμα και θα ήθελα να σε παρακαλέσω να μας κάνεις μια σύντομη παρουσίαση, το πολύ 15 λεπτά, 5 λεπτά ε, και την προηγούμενη εβδομάδα ε, στη διάσκεψη των Προέδρων Επιτροπών ε, κάνα μία ερώτηση προς τον κύριο Τίμερμαν και εκεί μας είπαν ότι το, φε... φθινόπωρο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να καταθέσει την άποψή της για την ε, στρατηγική δασών. Συνάδελφος Σάρβαμα. Αξιότιμοι συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Τα δάση, η δασοκομεία και όλος ο κλάδος των δασών διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην εξασφάλιση βιώσιμων λύσεων σε πολλές προκλήσεις των καιρών μας. Τα δάση και ε, άλλη ξυλώδης έκταση καλύπτουν τουλάχιστον το 43% της επιφάνειας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο δασικός κλάδος απασχολεί τουλάχιστον 500.000 Ευρωπαίους πολίτες άμεσα και 2,6 εκατομμύρια έμεσα. Επιπλέον, περίπου 60% των ευρωπαϊκών δασών ανήκουν σε ιδιώτες. Περίπου πριν από 30 χρόνια έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες μια προεκλογική εκστρατεία προεδρική με το σλόγγαν ε, «Είναι η οικονομία ηλίθια» ήταν το σλόγγαν του Μπιλ Κλίντον και πολύ επιτυχημένο. Φαίνεται τώρα ότι το κλίμα ε, είναι η λέξη κλειδί. Για να απαντήσουμε όμως ε, στο αν το κλίμα είναι χαζό ή αν η οικονομία είναι χαζή, θα πρέπει να βρούμε τη σωστή ισορροπία και στην ε, Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Διαχείριση των Δασών και θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι είναι διαφορετικά τα χαρακτηριστικά και διαφορετικές οι πραγματικότητες στα διάφορα μέρη της Ευρώπης. Υπάρχει μεγάλη πολυμορφία στη δομή, τη βιοπικιλότητα και διαχείριση των δασών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά τα θέματα λοιπόν θα ληφθούν υπόψη, όλε αυτέ οι διαφορέ και ιδιαιτερότητε, στην έκθεση πρωτοβουλία που θα συντάξουμε για την Ευρωπαϊκή Δασική Στρατηγική μετά το 2020. Καταρχήν, το παγκόσμιο περιβάλλον πολιτική έχει αλλάξει άρδιν από την τελευταία μα δασική στρατηγική του 2013 και αυτέ οι αλλαγέ επηρεάζουν ιδιαίτερω όλε τι πολιτικέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα δάση θα πρέπει να θεωρηθούν ως πρόβλημα της λύσης ε, και ταυτόχρονα την δέσμευσή μας για μια κοινωνία μηδενικών εκπομπών, την Νέα Πράσινη Συμφωνία, τους, κορός, τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, το πρωτόκολλο του Κιώτο και τη Συμφωνία των Παρισίων. Τα δάση είναι τμήμα της λύσης, δεν είναι πρόβλημα. Δεύτερον, ο αυξανόμενος αριθμός των ε, συναφών μεταδάσης πολιτικών δημιουργούν ένα περίπλοκο και κατακαιρματισμένο περιβάλλον πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, ας μην ξεχνούμε ότι η πολιτική για τα δάση αποτελεί εθνική αρμοδιότητα. Ως εκ τούτου, χρειαζόμαστε μία στεναρή, ολιστική και ανεξάρτητη στρατηγική για τα δάση μετά το 2020 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε μια σφαιρική άποψη για μια βιώσιμη αηφόρο δασική διαχείριση που θα λαμβάνει υπόψη τον πολυλειτουργικό ρόλο των δασών και τις, τους οικονομικούς, και περιβαλλοντικού πυλώνε με ισορροπημένο τρόπο. Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική Δράση θα πρέπει να είναι αναπόσπαστο τμήμα τη ε, μελλοντική ε, ευρωπαϊκή πράσινη συμφωνία. Και επίση θα ήθελα να πω ξεκάθαρα ότι η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα Δάση δεν θα πρέπει να υποταχθεί σε καμία άλλη στρατηγική. Δεν θα πρέπει να είναι υποδέστερη σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη στρατηγική θα είναι πολύ σημαντικό συντονιστικό μηχανισμό για τι πολιτικέ που αφορούν τα δάση και θα πρέπει να δημιουργήσει συνέργειε και συνοχή με άλλου τομεί που επηρεάζουν τη διαχείριση των δασών. Η στρατηγική για τα δάση επίση θα πρέπει να γίνει γέφυρα μεταξύ των εθνικών πολιτικών και τη Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει η εμπειρογνωσία για τα δάση να περιλαμβάνεται στα πρώιμα στάδια της διαμόρφωσης πολιτικής, ώστε να έχουμε συνεπείς ε, και συγκροτημένες ε, συναφείς δάση πολιτικές. Έτσι θα επηρεάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση το γενικό περιβάλλον πολιτικής. Η έκθεση πρωτοβουλίας μας θα επισημάνει τα εξή. Η σημασία της κοινή γεωρικής πολιτικής, η χρηματοδότηση των μέτρων για τα δάση και τα προγράμματα πλαίσιο για την έρευνα θα έχουν θεμελιώδη ρόλο. Η βιοπικιλότητα ε, και οι πτυχές της που ε, Συνάδων με το δάσο θα πρέπει να συμπεριληφθούν στη στρατηγική και να συναποφασιστούν με, με το δασικό κλάδο. Μία, διαχείριση, μία βιώσιμη διαχείριση και αποτελεσματική των δασών θα μας επιτρέψει να, να υλοποιήσουμε τους ενεργειακούς, περιβαλλοντικούς και κλιματικούς μας ρόλους. Ο μετριασμός των κλιματικών αλλαγών θα είναι μία από τις σημαντικές υπηρεσίες που θα μας προσφέρουν τα δάση. Επίσης, η προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές είναι πολύ σημαντικό για τα δασικά συστήματα και κάποιες επιδημίες με παράσιτα, ξηρασία ή δασοπερκαγιές θα πρέπει να προληφθούν ή να αποτραπούν. Άλλωστε έχουμε μια ολόκληρη αλυσίδα αξία ε, των δασών που είναι άρρηκτα δεμένη με τη βιοοικονομία που προσφέρει ευημερία και θέσεις απασχόλησης. Η επικαιροποίηση λοιπόν της ε, κυκλικής οικονομίας θα πρέπει να προωθηθεί με ισχυρές πολιτικές ε, έρευνας και καινοτομίας. Θα πρέπει επίσης να μειώσουμε την εξάρτησή μας από ορυκτά υλικά. Και θα πρέπει να αυξήσουμε τις ευκαιρίες, ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές. Ο δασικός κλάδος ε, με ψηφιακές λύσεις και βιώσιμες τεχνολογίες έχει δυναμικό να συμβάλλει όλο και περισσότερο στη διαφύλαξη της φύσης, να εξυπηρετήσει τους ανθρώπους και να προάγει μια κυκλική οικονομία με βάση τα βιοκαύσιμα. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δάση οπωσδήποτε. Και θα ήθελα να ολοκληρώσω με κάτι που είπα και στην αρχή. Πριν από 30 περίπου χρόνια στην προεκλογική εκστρατεία για τι προεδρικέ εκλογέ ε, τέθηκε το ερώτημα: Είναι χαζή η οικονομία, είναι ηλίθια η οικονομία. Νομίζω ότι ακόμη αυτό ισχύει. Γιατί αν ε, ισχυριστώ ότι η οικονομία είναι ηλίθια, δεν εννοώ ότι αυτοί που μιλούν για τον οικολογικό πυλώνα, ότι αυτοί που μιλούν για τον κοινωνικό πυλώνα κάνουν λάθο. Απλώ νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να αντιληφθούμε ότι και οι τρεις πυλώνες, όλες οι τρεις γωνιές του τριγώνου θα πρέπει να είναι σε σωστή ισορροπία. Χωρίς το οικονομικό πυλώνα θα υποφέρουμε και στον κοινωνικό αλλά και στον οικολογικό πυλώνα και δεν θα καταφέρουμε να νικήσουμε στην κλιματική μας μάχη. Και γι' αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να λάβουμε υπόψη και το θέμα της οικονομίας. Μόνο χάρη στην οικονομία θα έχουμε υγιή και ανθεκτικά δάση. Γιατί τα δάση δεν φυτρώνουν από μόνα τους. Ευχαριστώ. Vielen herzlichen Dank. Dann ähm, beginnen wir mit den äh, Schattenberichterstattern äh, jeweils eine ε, Ξεκινάμε με τους ε, σκέοντες ηγητές από 1,5 λεπτό έκαστος. Εγώ Χαιρετίζω αυτή την πρωτοβουλία για να υπάρχει μια νέα στρατηγική. Λοιπόν, είναι ένα θέμα το οποίο με ενδιέφερε επί πάρα πολλά χρόνια. Όπως ο κ. Σαβαρμάμος μας είπε, τα δάση θα είναι πολύ σημαντικός παράγον στην πολιτική του κλίματος και πρέπει γρήγορα και προσεκτικά να το εξετάσουμε το θέμα. Όμως, τουλάχιστον στα πλαίσια της Πράσινης Συμφωνίας, και λαμβάνοντας υπόψη την παρούσα κατάσταση, βλέπουμε ότι χρειάζεται κάποια κοινή προσέγγιση, κοινά μέτρα να εφαρμοστούν. Διότι, όπως είπε ο εισηγητή, είμαστε διαφορετικοί, αλλά θα πρέπει να δώσουμε τη μάχη κατά της αλλαγή του κλίματος μαζί. Πρέπει να κινηθούμε, θα πρέπει να πλησιάσουμε οι μεν δε, πιο κοντά από ό,τι μέχρι τώρα. Θέλω να αναφερθώ στη Ρουμανία, παρόλο που δεν είναι η μόνη περίπτωση που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ρουμανία πριν είχε τα περισσότερα παρθένα ε, δάση στην Ευρώπη, εκτός Σκανδιναβία. Σήμερα όμως η Ρουμανία είναι δραματικό παράδειγμα κακής διαχείρισης. Αυτή τη στιγμή από κάθε δύο δέντρα που κόβονται, το ένα από αυτά κόβεται παράνομα. 20 εκατομμύρια κυβικά μέτρα ξυλίας ε, το έτος εξαφανίζονται από τη Ρουμανία καταλήγουν, καταλήγουν σε κάποια κρεβατοκάμαρα ή σαλόνι της ε, Ευρώπης. Αυτό είναι, κοστίζει ένα δισεκατομμύριο ευρώ το χρόνο στην πατρίδα μου. Και απεριμόνονται τα βουνά, αποδασώνονται, ε, δημιουργούνται προβλήματα στις κοινότητες υπαίθρου, βλάπτεται η βιοπικιλότητα κλπ. Τελειώνω τώρα, τελειώνω. Νομίζω ότι θα πρέπει μέσω της νέας για τα δάση, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, να στείλουμε ισχυρό μήνυμα που δεν υποστηρίζουν τα σχέδια για τη βιώσιμη υλοτομία, να εφαρμόσουμε καλύτερα τα διαχειριστικά σχέδια, να ανανεωθούν ε, τα μητρώα, τα στοιχεία για τα δάση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θα πρέπει να έχουμε κανόνες για προστασία που θα είναι καλύτεροι για όλα τα δάση στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Συνάδελφε Φέντελ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Συγχαρητήρια για τον Πέτερ, ήταν πολύ καλή ομιλία. Κάλυψε όλα τα σημεία που ήθελα να θίξω. Προσβλέπω στην εξέταση του θέματος, είναι σημαντικότατο. Θέλουμε ισορροπία μεταξύ κοινοτικού δικαίου και τι αποτελεί αρμοδιότητα κράτους μέλους. Και η συνάδελφος από το Συριστικό Κόμμα έθεσε το πρόβλημα της Ρουμανίας. Μας προβληματίζει αυτό πολύ και μας. Χρειάζεται ισορροπία μεταξύ παράνομης υλοτομίας σε ένα κάτω μέλος που πρέπει να αντιμετωπιστεί σε, ένα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να μην δημιουργήσουμε προβλήματα για την λειτουργούσα βιοοικονομία. Να βρούμε ε, άλλα χημικά καινούρια με βάση βιολογικά προϊόντα που αντικαταστήσουν τα χημικά ε, να έχουμε κτίρια που θα είναι πιο δέτερα για το κλίμα στο μέλλον. Όλα αυτά θα δημιουργήσουν θέσει απασχόληση, αλλά τα μέτρα πρέπει να εφαρμοστούν με ένα βιώσιμο τρόπο, έχοντα υπόψη το μέλλον. Στι επικείμενε συζητήσει που θα εξαχθούν, θα αναφερθώ και στη ζωή που έχει ένα δέντρο. Εδώ, όταν μιλάμε για πολιτική για το κλίμα, όλοι ε, θεωρούν ότι μπορεί να μα σώσουν τα δάση από την αλλαγή του κλίματο. Όταν είναι πλήρω ανεπτυγμένο ένα δάσο όμω, σταματάει να εισπνέει διοξείδιο του άνθρακο και να απορροφά. Πρέπει να προστατεύσουμε κάποια τμήματα για λόγου βιοπικιλότητα, αλλά πρέπει να έχουμε και υπεύθυνη διαχείριση άλλων τμήματων του δάσου. Διαφορετικά, μετά από το 2050-2060 δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε τα δάση ε, σαν ε, χώρου που αποθηκεύεται το διοξείδιο του άνθρακο. Ευχαριστώ πολύ και προσβλέπω στην μελλοντική συνεργασία. Ευχαριστώ. Έχετε το λόγο εσείς, κύριε συνάδελφε. Ευχαριστώ πολύ. Είναι προφανές ε, ότι εμείς ε, είμαστε υπέρ του να υπάρχει μια νέα στρατηγική για τα δάση ως πράσινη. Στη συζήτηση αυτή βλέπουμε κάποια θέματα τα οποία ε, δυστυχώς ανακατεύονται ως κύβη που είναι άτακτα ερημένη. Ε, αυτό που έχει σημασία είναι να προστατεύσουμε την βιοπικιλότητα. Κατά νου μου έρχονται βέβαια τα Καρπάθια, αλλά ε, μην ξεχνάμε ότι και στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να γίνεται σεβαστή ε, το ενωσιακό δίκαιο. Αυτή τη στιγμή μόνο περίπου το 15% της προστασίας επιτυγχάνεται από αυτή που θα έπρεπε να επιτευχθεί. Από την άλλη υπάρχει εξή συζήτηση. Ε, ποια μορφή της δασοπονίας έχει σήμερα για την Ευρώπη. Και πρέπει να πω ούτε ε, τα δάση που είναι κακώς διαχειριζόμενα είναι καλή λύση, ούτε και το άλλο άκρο. Κατά την άποψή μου, στην Ευρώπη έχουμε πολύ διαφορετικά δάση, δάση που μερικές φορές έχουν χρησιμοποιηθεί πολύ, άλλα πάλι που είναι πολύ αραιά, ε, που ίσως θα ήταν καλύτερα να τα αφήσουμε στην ησυχία τους για κάποιο χρονικό διάστημα. Άρα δηλαδή θα πρέπει να διαφοροποιηθούμε λιγάκι στη συζήτηση που κάνουμε. Ε, το νέο τη νέα πράσινη συμφωνία θα πρέπει να την συσχετίσουμε με τη δασοπονία και για μας αυτό που έχει σημασία είναι να κάνουμε διορθώσεις στη βιοενέργεια και στη βιομάζα. Γιατί κάναμε κάποιους λάθος υπολογισμούς σήμερα και με περισσότερα ξύλα ε, και λέμε ότι αυτά είναι ανανεώσιμα. Ε, πρέπει όμως να αφήσουμε τα δάση να μεγαλώσουν για να ανθίστανται καλύτερα στο κλίμα και προφανώς ε, θα πρέπει να ασχοληθούμε με μια πολυλειτουργική δασοπονία αλλά πρέπει να ορίσουμε ποια λειτουργία για μας είναι σημαντικότερη. Και τέλος, αυτό που έχει σημασία είναι πώς μπορούμε να καλύψουμε τις ε, τις βιολογικές ελλείψεις. Ε, μιλήσατε με μια υπερβολική ταχύτητα, λέει ο πρόεδρος. Ε, προφανώς σας παρακάλεσαν διερμηνείς να μιλάτε Η δυνατόν λίγο πιο αργά. κυρία Γκυλάρ, ευχαριστώ. Είναι πολύ τη μόδα να μιλούμε για τάση και εντό και εκτό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πάντω είναι θετικό που όλο και περισσότεροι άνθρωποι συνειδητοποιούν το ρόλο των δασών στη ζωή και την οικονομία και τη συμβολή των δασών στη Νέα Πράσινη Συμφωνία. Ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όμως θα πρέπει να έχουμε συγκροτημένη στρατηγική. Έχουμε ε, τώρα σε τρεις διαφορετικές επιτροπές ε, τρεις εκθέσεις πρωτοβουλίας για τα δάση. Φοβάμαι ότι η εύλογη συζήτηση για την αποψήλωση των δασών σε τρίτες χώρες ίσως δημιουργήσουν μια υπεραπλουστευμένη εντύπωση απομακρυσμένοι από την πραγματικότητα του δασικού κλάδου και των προκλήσεων. Θα πρέπει να αλλάξουμε το status quo του δασικού τομέα. Θα πρέπει ε, να γίνουν αλλαγές, αλλά λαμβάνοντας υπόψη την, την πολυμορφία του δασικού τομέα και την αποκλειστική εθνική αρμοδιότητα για τη διαχείριση των δασών. Η ανταγωνιστικότητα των δασών προϋποθέτει ένα κατάλληλο νομικό πλαίσιο που θα αναδεικνύει την πολυλειτουργική διάσταση των δασών. Και μια δασική στρατηγική μετά το 2020 θα πρέπει να αποτελέσει το βασικό άξονα της νέας πολιτικής για τα δάση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ähm, Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο συνάδελφο Μπομπά δεν είναι παρόν. ω εκ τούτου περνάμε στου υπόλοιπου ε, ομιλητέ, ε, Έκαστος ε, εξ αυτών, παρακαλώ για ένα λεπτό, ο συνάδελφο Καβαγιέ. Ευχαριστώ. Τα δάση διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην διάρθρωση των κοινοτήτων. Είναι πυλώνας της αγροτικής οικονομίας και της παραμονής του πληθυσμού στις πιο απομακρυσμένες περιοχές που είναι εκτεθειμένες στην αποερήμωση. Και μάλιστα ε, τα δάση στην Πορτογαλία είναι πάνω από το 50% της ε, επιφάνειας της επικράτειάς μας και αυτό είναι πολύ σημαντικό στους ρόλου τους. Έχουν διάφορες υπηρεσίες οικοσυστημάτων τα δάση και πολύ λειτουργική διάσταση. Αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στη νέα στρατηγική για τα δάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, είναι σημαντικά τα, συστήματα, τα άγρο δασικά συστήματα. Θα συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και στο μετριασμό των κλιματικών αλλαγών. Αυτά τα συστήματα συνδυάζουν ε, την ε, αγροτική δραστηριότητα με την ε, δασοπονία και νομίζω ότι μπορούν να δεσμεύσουν και να αποθηκεύουν άνθρακα, να διασφαλίσουν την προστασία της πανίδας της φυσικής και έχουν και άλλα ωφέλη που δεν είναι μόνο περιβαλλοντικά αλλά και κοινωνικο-οικονομικά επιτρέπουν στους γεωργούς ε, να παράγουν προϊόντα με αυξημένη προστιθέμενη αξία, πιο ποικιλόμορφα και διαφοροποιώντας το γεωργικό του εισόδημα συνδυάζοντας τον, με τη δασοπονία. Όλα αυτά τα σημεία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στη χάραξη της νέας στρατηγικής για, τη, για τα δάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ. Και εμεί ευχαριστούμε. Συνάδελφος ε, Τολερέ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όσον αφορά τα δάση, Όλοι είδαμε να καίγεται η Αυστραλία. Και αν χρειάζεται να έχουμε μια στρατηγική ευρωπαϊκή όσον αφορά τα δάση, επίση χρειαζόμαστε να έχουμε μια στρατηγική παγκόσμια όσον αφορά την αναδάσωση. Όμως ε, γι' αυτό μία από τις προτάσεις που θα μπορούσε να γίνει είναι να έχουμε ένα σύστημα πιστοποίησης των ευρωπαϊκών δασών ούτω ώστε νομίμω να μπορούμε να ζητάμε εντό των διεθνών συνθήκων να γίνεται μνήμα του σεβασμού των ίδιων συνθήκων προστασίας των δασών, δηλαδή να απαγορεύονται προϊόντα που απορρέουν από την αποδάσωση, την αχαλήνωτη. Λυπάμαι διότι σε επίπεδο προπολογισμού λέμε ότι το δάσος είναι πάρα πολύ σημαντικό και πλευρά χρημάτων για την ώρα. Τα κονδύλια για τα δάση ουσιαστικά φεύγουν, βγαίνουν από την ΚΑΠ. αν είναι σημαντικά πρέπει να βρούμε από αλλού τα χρήματα για να μπορέσουμε να συμπληρώσουμε τις ανάγκες τις οικονομικές και όταν διαχειριζόμαστε τα δάση θα πρέπει να ε, αναπτυχθούμε τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ξυλία σε οικονομικό επίπεδο. Ευχαριστώ, συνάδελφε ε, Λαν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την πολύ καλή βάση που μας προσφέρει. Προβάλλει την πολυλειτουργικότητα των δασών. Αυτό που είναι γεγονός είναι ότι μέσα στην Ευρώπη Έχουμε δάση ε, τα οποία επεκτείνονται σε έκταση. Αυτό δεν το συνειδητοποιούν πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι όμως ένα σημαντικός παράγον τον οποίο πρέπει να προβάλλουμε εδώ στην Επιτροπή Γεωργίας. Με τα δάση μας και στη Γερμανία έχουμε δύο εκατομμύρια ιδιώτες ιδιοκτήτες δασών, οι οποίοι είναι πολύ υπεύθυνοι, πολύ υπεύθυνοι δασοπόνοι. Και σας το λέω ξεκάθαρα, δεν ξέρω αν το ξέρετε, σε ένα κυβικό μπετόν έχουμε 2,5 2,5 τόνοι ε, και καταβάλλονται πάρα πολλές μεγάλες ποσότητες οξυγόνου ε, για να κατασκευαστεί. 5 τόνοι είναι ένας, ε, ένα κεβικό ξύλου και δεσμεύει μεγάλες ποσότητες διοξίδι του άνθρακα. Αυτά ήταν έτσι κάποιες ε, πληροφορίες που είχα να σας δώσω. Τώρα δεν έχω λόγο να μιλήσω. Ό,τι άλλο έχω να πω θα το καταθέσω με τροπολογίες. Ευχαριστώ κύριε Σλεμπρετόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τα δάση είναι πολύ σημαντικό στοιχείο στην Ευρώπη αντιπροσωπεύουν το 43% της ευρωπαϊκής επικράτειας και αυξάνονται κατά 0,85% το χρόνο την τελευταία δεκαετία. Επίσης, ε, σημαντικό στοιχείο για την προστασία του περιβάλλοντος, μετριάζουν τις κλιματικές αλλαγές, αλλά σημαντικό στοιχείο και της οικονομίας συμβάλλουν στην αγροτική ανάπτυξη και δημιουργούν 3 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης. Είμαι υπέρ λοιπόν της ε, συνεργασίας για τα δάση, μια και η στρατηγική τη Ευρωπαϊκής Ένωση για τα δάση ε, ισχύει εδώ και 20 χρόνια θα πρέπει να προστατεύσουμε και να αξιοποιήσουμε καλύτερα αυτό το δασικό πλούτο. Αλλά θα πρέπει ταυτόχρονα να είμαστε συνετοί, γιατί τα δάση διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Αυτέ τι διαφορέ θα πρέπει να τι λάβουμε υπόψη και να προβλέψουμε αρκετή ευελιξία. Γιατί τα δάση είναι και θα πρέπει να παραμείνουν στην εθνική αρμοδιότητα και δεν θα πρέπει να θίξουμε αυτή την εθνική ε, αρμοδιότητα υπό το πρόσχημα της εφαρμογής της μελλοντικής ε, πράσινης συμφωνίας. Ευχαριστώ κύριο Σαντάμοφ. Горите в Европейския съюз са нашето Κύριε Πρόεδρε, τα δάση στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο πράσινος πλούτος μας και έχουν να διερματίσουν ένα πολύ σημαντικό ε, οικονομικό και κοινωνικό ρόλο. Τα δάση μας ε, βοηθούν να εξετερώσουμε τις ε, βλαβερές εκπομπές Βέβαια πρέπει να γνωρίζουμε ότι πάρα πολλά δάση στην Ευρώπη κινδυνεύουν Δυστυχώς υπάρχουν ακραία φαινόμενα που θέτουν σε κίνδυνο τα δάση, όπως οι δασοπυρκαγιές, η ξηρασία και παρεμφερή. Όλα αυτά βέβαια απαιτούν να υπάρχει μια βιώσιμη διαχείριση των δασών, όπως και στενή συνεργασία ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Γι' αυτό λοιπόν εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να είχαμε και να έχουμε περισσότερα δάση, να στηρίξουμε την αναδάσωση, γιατί χωρίς ε, δάση δεν μπορεί να υπάρξει και πράσινη συμφωνία. Εύχομαι καλή επιτυχία στον εισηγητή. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για την έκθεση που παρουσίασε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τη στρογγυλή τράπεζα που οργανώθηκε χτες και που είχαν προσκληθεί εμπειρογνώμονες από ολόκληρη την Ευρώπη. Είχαμε εκεί παρόντες εμπειρογνώμονες αλλά και ιδιοκτήτες δασών. Στην Σλοβενία επεκτάθηκαν τα τελευταία χρόνια τα δάση. Έχουμε βιώσιμη διαχείριση δασών και οι ιδιοκτήτες δασών ε, διερωτώνται τι θα γίνει ε, στο μέλλον. Ε, πολλοί ακούν ότι θα προστατεύονται πλήρως τα δάση. Νομίζω ότι πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες έτσι ώστε το δάσος να είναι ένα κομμάτι της λύσης. Χρειαζόμαστε λογική διαχείριση Ακούσαμε ε, το ρόλο που μπορεί να παίξουν τα δάση στο, στην περίπτωση του διοξιδίου του άνθρακα. Ε, τα δάση έχουν να διαδραματίσουν λειτουργικό ρόλο και τα δάση μπορεί κανείς και να τα χρησιμοποιήσει για την παραγωγή ενέργειας. Ε, τα δάση είναι τμήμα της λύσης και από αυτού συμφωνώ απόλυτα με τον εισηγητή. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Γιούργελ. κύριε Πρόεδρε. Μιλούμε για ένα τομέα που ανήκει στην εθνική αρμοδιότητα. Θα πρέπει να διαφυλάξουμε αυτή την εθνική αρμοδιότητα για τα δάση. Η νέα στρατηγική θα πρέπει να ενισχύσει την προηγούμενη στρατηγική και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε δάση και δασικό κλάδο που θα συμβάλλει στην υλοποίηση όλων των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης και θα πρέπει να εξασφαλίσει ποιοτική μετάβαση της δασικής ε, διαχείρισης, λαμβάνοντας υπόψη την πολυλειτουργικότητα των δασών. Επίσης θα πρέπει να καταλήξουμε σε μια ισορροπία μεταξύ της προστασίας του κλίματος, τους βιοποικιλότητες, αλλά και των κοινωνικο-οικονομικών στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα αυτά ε, περιλαμβάνονται και στις ε, άλλες στρατηγικές. Θα πρέπει να υπάρχει οριζόντια λήψη υπόψη των δασών. Και τέλος, ε, θα ήθελα να αναγνωρίσουμε την, την αρχή της επικορικότητας και την ε, αποκλειστική εθνική αρμοδιότητα για θέματα διαχείρισης των δασών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, συνάδελφε Κατάιν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Σαββάρμαν. Είναι πολύ σημαντική αυτή η έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας για τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Το ζητήσαμε στην προηγούμενη θητεία. Διάφορα τμήματα της Πράσινης Συμφωνίας θα επηρεάσουν άμεσα το δάσος, η νέα κυκλική οικονομία, η νέα νομοθεσία, το κλίμα και η στρατηγική για τη βιοπικιλότητα. Είναι παρόμοια αυτή η περίπτωση με τον κανονισμό για το Λούλουσεφ και την οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενεργείας που θα επανεξεταστεί. Η στρατηγική για τα δάση θα πρέπει να κατευθύνει την προετοιμασία της δημιουργίας αυτών των νόμων και της στρατηγικής. Ε, Μία βιώσιμη διαχείριση των δασών πρέπει να ενταχθεί στη στρατηγική με τις τρεις διαστάσεις που περιέγραψε άριστα ο κ. κοινωνική, ε, οικονομική και περιβαλλοντική πτυχή. Τέλος, να πω μόνο τα αναπτυσσόμενα δέντρα μπορούν να απορροφήσουν τον άνθρακα. Αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη. Ευχαριστώ, συνάδελφε Χόισλε. Ευχαριστώ. Αναφέρθηκε ότι η διαχείριση του δάσους θα βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα του κλίματος. Είδαμε όμως να γίνεται κακοδιαχείριση των δασών. Ε, τέσσερα δάση στην... Ε, μάλλον έχουν τα δάση με τα πέλατα, έχουν πάθει πολλές ζημιές στη Γερμανία, τα κονοφόρα έχουν υποφέρει και στη Γερμανία και στην Πορτογαλία και ήταν δάση που είχαν ενταχθεί σε ένα σύστημα διαχείρισης. Στη δική μου περιοχή έχουμε χάσει 30% των δασών μας ε, λόγω ξηρασίας και λόγω του θανάτου των κονοφόρων. Οπότε η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωση πρέπει να παίξει σημαντικό ρόλο εκεί. Δαχτυλοδειχτούμε τη Βραζιλία και τους λέμε προστατεύστε τα δάση σα. αλλά δείτε τι κάνουμε και εμεί στα δικά μας δάση και τι γίνεται. Θα πρέπει να ακολουθήσουμε νέε προσεγγίσεις για τη διαχείριση των δασών και θα πρέπει αυτά να συζητηθούν. Θα πρέπει να έχουμε περιφερειακή, αν θέλετε, περιφερειακούς κύκλους που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη αυτοί οι κύκλη, μια στρατηγική που μέχρι τώρα είχε αγνοηθεί. Ε, υπάρχουν επίσης ιδιοσυγκρασίες μεταξύ των διαφόρων περιοχών και ιδιαιτερότητες. κυρία Σνέμπολ, ευχαριστώ, συνάδελφε. Ε, συνάδελφε Πέτρη, ε, συγχαρητήρια για την εκπόνηση της έκθεσης πρωτοβουλίας. Για την πατρίδα σου, τη Φιλανδία, τα δάση είναι τόσο σημαντικά όσο και για μας τους Αυστριακούς. 48% της Αυστριακής επικράτειας καλύπτεται από δάση. Οπότε φαντάζεστε ότι είμαι και εγώ υπέρ μιας θετικής στρατηγικής. Η στρατηγική αυτή θα πρέπει να είναι και βιώσιμη, αλλά και να λαμβάνει υπόψη τις εθνικές ιδιαιτερότητες και διαφορές. Τα δάση δεν είναι και μουσείο διοξιδίου του άνθρακα. Δεν είναι το πάνθεον του διοξιδίου του άνθρακα θα πρέπει να δώσουμε έμφαση στην αναδάσωση και να προβούμε σε μία ενεργό διαχείριση των δασών. Αυτό είναι ένα δύσκολο έργο που συναρπάζει τους ε, ιδιοκτήτες των δασών. Και είναι σίγουρο ότι τα δάση δεσμεύουν διοξίδιο του άνθρακα, αλλά η δασοκομεία στην Ευρώπη δημιουργεί και 3 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης. Δημιουργεί θέσεις εργασίας στις αγροτικές περιοχές σχεδόν αποκλειστικά. Όταν μιλούμε ότι θέλουμε να κρατήσουμε τον αγροτικό πληθυσμό στην Ήπεθρο, είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη τη συμμετοχή των δασών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, στην Ουγγαρία δεν έχουμε μόνο στόχο τη διατήρηση των δασών, αλλά και την αύξησή τους, την επέκτασή τους. Η αύξηση της ιωρικής παραγωγής συνάδει και με την αύξηση της δασικής επιφάνειας. Δεν είναι αντιφατικοί αυτή η δύο στόχοι. Και σωστά λέμε ότι είναι σημαντικός ο ρόλος των δασών και για την οικονομία και για το περιβάλλον. Για να είναι επιτυχημένη η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα δάση, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε τη συνοχή μεταξύ της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Αυτό είναι μια καλή βάση για να αποτρέψουμε την αποψήλωση των δασών στον κόσμο. Και γι' αυτό θα πρέπει η στρατηγική μας για τα δάση μετά το 2020 να προτείνει αποτελεσματικές λύσεις για να ελοπίσουμε τους στόχους μας. Ευχαριστούμε πολύ. Συνάδελφος ε, Ντάβιτ, έχετε το λόγο. Ε, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εμείς ε, στην Τσεχία το 33% της έκτασής μας ε, είναι δάση. Από τον 19ο αιώνα τα δάση ήταν μονοκαλλιέργειες, ε, πευκοδάση είναι αυτά σε εμά, ναι. τα οποία υπέφεραν πάρα πολύ, ε, διότι τώρα έχουν πληγεί από την χρόνια ξηρασία. Αυτή τη στιγμή ε, τα δάση μας υποφέρουν Έχουμε πολλούς ε, φανατικούς ε, οι οποίοι δένονται μόνοι τους, προσδένονται πάνω στο δάση για να μην τα κόψουν οι ξυλοκόποι. Ε, εγώ θεωρώ ότι η δασοπονία είναι πάρα πολύ σημαντική για την κλιματική αλλαγή Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να ε, διατηρηθούν οπωσδήποτε τα δάση και εγώ ε, δεν θα δίσταζα να χορηγήσω ενισχύσεις. Αυτό θα ήταν πολύ καλύτερο από το να διοχετεύονται ενισχύσεις για την ηλεκτροκινητικότητα, για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το γεγονός είναι ότι στην Ευρώπη βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλά ε, μικρά δάση πρωταρχικά δάση, τα οποία δεν μπορεί κανείς ε, να τα δεκτείνει ε, ε, μόνο να τα προστατεύσει. Πιστεύω λοιπόν ότι μια καλή στρατηγική για τα δάση, μια τέτοια στρατηγική για τα πρωτογενή δάση θα πρέπει να προστατεύει αυτά, αλλιώς δεν είναι μια καλή στρατηγική. Συνάδελφος Σάντερ. Ευχαριστώ κύριε, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ όπως συνάδελφοι να επιμείνω στην ανάγκη ε, να έχουμε μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δάση. Μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δάση και να σκεφτούμε από κοινού πώς θα αναδείξουμε την αξία των δασών και την περιβαλλοντική που είναι αναφυσβήτητη γιατί τα δάση διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη δέσμευση του άνθρακα αλλά μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε και οικονομικά. Θα πρέπει να τα διαχειριστούμε λοιπόν κατάλληλα. Γιατί έχουμε πολλές θέσεις απασχόλησης που συνδέονται με το δασικό κλάδο. Είναι και θέμα χωροταξίας επίσης. Στη στρατηγική για τα δάση μετά το 2020 θα πρέπει από κοινού να προστατεύσουμε τα ευρωπαϊκά δάση, να τα προστατεύσουμε από τις δασοπυρκαγιές αλλά και από τα παράσιτα. Στην δική μας περιφέρεια έχουμε ένα παράσιτο που καταστρέφει τα δάση Σκολίτης και νομίζω ότι μόνο με ευρωπαϊκή λύση θα διορθώσουμε αυτό το πρόβλημα. Πρόεδρο, πολύ ωραία. Ε, εξαντλήθηκε λοιπόν ο κατάλογο των ερωτώντων και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, στον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή, κύριο Δημήτρου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα πρέπει να πω ότι καλωσορίζουμε αυτή την έκθεση. Νομίζω ότι η έκθεση είναι ένας πολύ καλός τρόπος ε, για να παρουσιάσουμε τα δάση γιατί εντοπίζονται όλες αυτές οι υπηρεσίες που προσφέρονται από τα δάση που είναι πολύ σημαντικά για την Ήπετρο, για την τοπική κοινωνία, για την οικονομία, ε, για τις ε, προκλήσεις που υπάρχουν. Εμείς είμαστε ευγνώμονες για το ρόλο που παίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτή την στρατηγική για τα δάση. Τώρα είμαστε στο τέλος της δεύτερης χρονιάς και έχουμε ακούσει την άποψη των θεσμών, των κρατών μελών, των άμεσα ενδιαφερόμενων, ανάγκη να υπάρξει μια νέα πολιτική. Όσον αφορά στο μέλλον, Πρόσφατα εγκρίθηκε μία ανακοίνωση για την Πράσινη Συμφωνία και έτσι η Κομισιόν δεσμεύεται να προετοιμάσει μία νέα χρονιά για τα δάση. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να προσφέρονται πολλές υπηρεσίες από τα δάση. Είναι λοιπόν μία δική μας στρατηγική που δεσμευόμεθα να προσφέρουμε. Αυτή η στρατηγική θα καθορίσει το πλαίσιο για τη δασοπονία για να είναι συμβατή αυτή η πολιτική με την Πράσινη Συμφωνία. Παράλληλα θα αντιμετωπίζονται και οι προκλήσεις. Και νομίζω όλοι αναγνωρίζετε ότι τα δάση μπορούν να προσφέρουν πολλές ευκαιρίες. Είναι μέρος της λύσης της Πράσινης Συμφωνίας. Συνεπάγονται πολλά πλεονεκτήματα. Βασική στόχη ε, στην Πράσινη Συμφωνία είναι η απορρόφηση του διοξιδίου του άνθρακα, ε, ο περιορισμός των δασοπυρκαγιών που ε, κατέστησαν καταστροφικές. Είδαμε τι εκτελήσεται στον κόσμο και προαγωγή της βιοοικονομίας. Επίσης, ε, πρέπει να συνεχίσουμε με τη νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βιοπικιλότητα που θα γίνει δεκτή τέλος του μήνα. Το θέμα της πολυλειτουργικότητας που συζητήθηκε εκτενώς εδώ και χτες και σε άλλες εκδηλώσεις αυτό είναι καθοριστική σημασία για να βρούμε τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στη δέσμευση διοξιδίου του άνθρακα, υλικό για τη βιοοικονομία, βιοπικιλότητα και παροχή άλλων υπηρεσιών ε, σε ένα κόσμο που έχουμε ε, κλιματική αλλαγή απαιτούνται πολλές καινοτομίε, γνώση, τεχνικές ικανότητες, τεχνογνωσία και ε, πρέπει να προσφέρουμε αυτή τη νέα στρατηγική. Η ε, Πράσινη Συμφωνία προβλέπει την διατήρηση των δασών, την αποκατάσταση, την αναδάσωση στην Ευρώπη. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε σωστή διαχείριση για να αποφύγουμε δαπανηρές επενδύσεις, να μπορούμε να ε, προσφέρουμε μια ισορροπία. Η βιώσιμη διαχείριση των υπαρχόντων δασών πρέπει να βοηθάει στην πρόληψη καταστροφών και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Υπάρχει κίνδυνος να χάσουμε και περισσότερα αξιόλογα δάση από τις ε, ασθένειες και από τις ε, δασοπυρκαγιές τα δάση θα εξακολουθούν να βρίσκονται στο κέντρο της νέας ΚΑΠ. Τα εργαλεία που έχουμε στα χέρια μας για τα δάση βρίσκονται στην ΚΑΠ. Πρέπει να συνεργαστούμε με τα κράτη-μέλη για να εντάξουν και τα δάση στα νέα τους εθνικά στρατηγικά σχέδια, να λάβουν και νέα μέτρα για τα δάση. Να έχουμε μια ολιστική προσέγγιση το 2020. Εμείς αυτό, ε, σε αυτό αποβλέπουμε και πολύ σύντομα θα σας το παρουσιάσουμε να το δείτε κι εσείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Επιτροπή και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον εισηγητή για να συνοψίσει τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ για τα θαυμάσια σχόλιά σας. Ε, πραγματικά πάρα πολύ ζωντανή και ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων. Πάρα πολύ σύντομα θα ήθελα να μου επιτρέψετε να αναφερθώ σε κάποιες παρεμβάσεις. Η κυρία Μούλνερ Κυρία Μίλνερ, ήταν πάρα πολύ καλό το γεγονός ότι υπογραμμίσατε την πολυλειτουργικότητα. Νομίζω όμως ότι αυτό που είπατε στο τέλος ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον, όπου διερωτηθήκατε, ε, ίσως ρητορικά να ήταν το ερώτημα, κατά πόσο γνωρίζουν όλοι οι υπόλοιποι επιστημονικά ε, το πόσες ποσότητες διοξείδου του άνθρακα εκλείονται όταν ε, καίγονται τα δάση και αντίθετα πόσε μεγάλε ποσότητε του άνθρακα δεσμεύονται όταν είναι ζωντανά τα δάση. Πρέπει να δούμε σε βάθο τα επιστημονικά γεγονότα. Και εδώ θέλω να πω και κάτι άλλο που είπε και ένα άλλο συνάδελφο. Κοιτάξτε, όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να προστατεύουμε τα δάση. Νομίζω όμω το κέριο ερώτημα είναι ε, πώς ακριβώς ε, κατανοούμε, τι ακριβώς εννοούμε όταν λέμε να προστατεύσουμε. Ίσως θα πρέπει σε αυτό να εμβαθύνουμε και να διερωτηθούμε ε, ποιες είναι οι δράσεις μας εκείνες που προστατεύουν τα δάση, τη βιοπικιλότητα και όλα τα συμπαρομαρτούντα. Και εκεί, σε αυτό το θέμα, επανέρχομαι στο συμπέρασμα ότι τελικά η βιώσιμη διαχείριση των δασών είναι Καταλητική σημασία Και πάω τώρα και σε αυτά που είπε ο κύριος Χόισλινγκ. Νομίζω έχετε ε, πράγματι δίκιο. Χρειαζόμαστε νέες ρηξικέλευτες μεθόδους στην Ευρώπη και υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν έχουν γίνει σε πολλά μέρη της Ευρώπης. Χρειαζόμαστε περισσότερα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, περισσότερες έρευνες ε, μέσα στα δάση, ε, να ε, υπάρχουν μηχανισμοί για να σβήνονται οι πυρκαγιές αν είναι δυνατόν. Και το πιο σημαντικό, χρειαζόμαστε ε, υγιή, επεκτηνόμενα δάση και μεγάλες εκτάσεις δασών, οι οποίες θα απορροφούν και θα αποθηκεύουν το διοξίδιο του άνθρακα. Και όταν θα έρχεται η στιγμή για υλοτομία, εκεί παίζει ρόλο κάτι άλλο πολύ σημαντικό που είναι η κυκλική οικονομία. Να κατασκευάζουμε προϊόντα τα οποία και αυτά πάλι με τη σειρά τους θα αποθηκεύουν διοξίδιο του άνθρακα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Υπάρχουν λοιπόν διάφορες φάσεις και η βιώσιμη διαχείριση δασών, όταν γίνεται σωστά, ενδελεχώς και σε βάθος, πραγματικά προσφέρει απάντηση σε όλες αυτές τις ε, ανησυχίες που εκφράστηκαν σήμερα για τα δάση μας. Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο. Ε, η έκθεση ίσως συζητηθεί στις 18-19 Μαρτίου. Ε, 25 Μαρτίου, καταληκτική ημερομηνία για κατάθεση τροπολογιών. Θα ψηφίσουμε τέλη Μαΐου, 25-26 Μαΐου και στην Ολομέλεια θα πάμε τον Ιούνιο. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σάβαμα. Επιτέλους φτάσαμε στο τέλος της σημερινής ε, ημέρας. Ευχαριστώ όλους όσοι Μείνατε εδώ μέχρι τέλους. Αύριο το πρωί θα τα πούμε στις 9 και θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με το νέο μας επίτροπο. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ τους, ε, τους και τις διερμηνείς ο Πρόεδρος.